Um, Συναδελφοί, καθίστε παρακαλώ. Έχουμε πολλούς ομιλητές και περιορισμένο χρόνο. Να αρχίσουμε στην ώρα μας λοιπόν. Πρώτα απ' όλα, σας παρακαλώ, μετακινηθείτε και ελάτε στα προστινά καθίσματα. Υπάρχει χώρος Ελάτε πιο μπροστά, παρακαλώ. Εντάξει, ξέρω, η αίθουσα είναι μεγάλη και όλοι αισθανόμαστε κάπως περίεργα εδώ, αλλά ελάτε πιο κοντά. Θα έρθουν κι άλλοι βέβαια κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Πάντως, ελάτε. Εκτός βέβαια από τις θέσεις που έχουν τα μπελίτσες που λένε ότι είναι για τους ευρωβουλευτές, έτσι. Αλλιώς στις υπόλοιπες θέσεις μπορείτε να καθίσετε. Ωραία. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, καλώς ήρθατε στην σημαντική αυτή ακρόαση για την κατάσταση και τα δικαιώματα των πολιτών τη Ευρωπαϊκή Ένωσης μετά τον Brexit και των Βρετανών που ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε πολλούς εμπειρογνώμονες, ε, ειδικού, εκπροσώπους των θεσμικών οργάνων και πέρυσι το Μάιο είχαμε οργανώσει κάτι για να συζητήσουμε το ίδιο αυτό θέμα. Τώρα συμμετέχουν εδώ και η Επιτροπή Απασχόλησης και η Επιτροπή Αναφορών. Η προηγούμενη ακρόαση... Α, και συνταγματικών υποθέσεων είναι εδώ. Και η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Λοιπόν, η ακρόαση εκείνη είχε θέσει διάφορα ζητήματα που σιγά σιγά βλέπουμε να εμφανίζονται μπροστά μας όσο περνάει ο καιρός και προχωρούν οι διαπραγματεύσεις. Τώρα έχουμε φτάσει στο τέλος αυτής της διαδικασίας. Αλλά όπως όλοι γνωρίζουν εδώ, τίποτα δεν έχει αποφασιστεί αν δεν έχουν αποφασιστεί όλα, αν δεν έχουν συμφωνηθεί δηλαδή όλα. Οπότε πρέπει να δούμε τι θα γίνει στη διάρκεια αυτού του διαζυγίου. Ο κύριος Γκαλτιέρη ήταν στην ε, διευθύνουσα ομάδα για το Brexit και είναι και πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων βέβαια. Μας έχει ενημερώσει και μας έχει εξηγήσει ότι πολλά μπορούν να γίνουν ακόμα μέχρι την ημερομηνία που έχει οριστεί για το Brexit και όπως έχουμε ακούσει σήμερα Είμαστε πραγματικά σε μια μεταβατική περίοδο. Λοιπόν, σε αυτή την ακρόαση θα ακούσουμε διάφορα και θα προσπαθήσουμε στο τέλος της να έχουμε κατανοήσει το εξής. Τι έχουμε πετύχει σε αυτό το στάδιο διαπραγματεύσεων για το διαζύγιο και τι πρέπει ακόμα να γίνει. Τι διακανονισμό χρειαζόμαστε να πετύχουμε από τώρα μέχρι την ημερομηνία του Brexit και τι είναι που πρέπει να περάσουμε σαν μήνυμα στο ακροατήριο. Θα το κάνουν αυτό οι διάφοροι εκπρόσωποι σίγουρα. Θα ακούσουμε από διάφορες οργανώσεις για το δικό τους έργο. Θα σας τα πούνε φυσικά οι ίδιοι οι διάφοροι εκπρόσωποι των οργανώσεων, οι ειδικοί κλπ. για εισαγωγή. Θα δώσω το λόγο στη συνάδελφο της ε, Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, την Μαρίτα Ιλκσκόχ, η οποία θα μας ε, πει τη συμμετέχει και εκείνη στη διευθύνουσα ομάδα. δεν ξέρετε, να ξέρετε ότι είναι το κομμάτι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις. Οπότε σας παρακαλώ σε όλους να πείτε ευχαριστούμε για τις διαπραγματεύσεις που κάνουν. Θα ακούσαμε βέβαια μετά και τον Κουαλτιέρη, συμμετέχει και ο κύριος Φερχόφστατ βέβαια, αλλά και η κυρία Ουλσκόκ συμμετέχει για τα θέματα που έχουν να κάνουν με την απασχόληση πιο πολύ. Πρέπει να δούμε λοιπόν τι γίνεται με αυτή την κοινωνική διάσταση που είναι και τόσο σημαντική. Η Μαρίτα λοιπόν παρακαλώ να μας κάνει μια σύντομη εισαγωγή εκ μέρους της Επιτροπής Απασχόλησης. Ευχαριστώ πολύ Κλοντ. Όπως ε, έχετε ήδη καταλάβει, δεν είναι η πρώτη κοινή ακρόαση που κάνουμε μεταξύ μας. Έχουμε ξανακάνει και το Μάιο. για τα δικαιώματα των πολιτών μετά το Brexit. Το Μάιο λοιπόν είχαμε μια πολύ χρήσιμη ακρόαση για μας τους ευρωβουλευτές. Ουσιαστικά ζητούσαμε από τους ευρωβουλευτές να παρακολουθήσουν από κοντά τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ηνωμένου Βασιλείου. Ευρώπης και Ηνωμένου Βασιλείου δηλαδή και να φροντίσουν να στηρίξουν τα δικαιώματα των πολιτών. Αυτό ακριβώς κάναμε και πιστεύω ότι η φωνή μας, η φωνή δηλαδή των πολιτών, των εργαζομένων έχει ακουστεί Και αυτό για θέματα που έχουν να κάνουν με αρμοδιότητα της δικιάς μου επιτροπής ε, των διασυνοριακών εργαζομένων για παράδειγμα θέματα κοινωνικής ασφάλισης και δικαιούχων. Αυτή είναι η αρμοδιότητα της Επιτροπής Απασχόλησης. Είμαστε Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε αρμοδιότητες πολύ περίπλοκες σε σχέση με το Brexit. Οπότε, ως πρόεδρος της Επιτροπής Απασχόλησης, πολύ χαίρομαι για αυτή τη δεύτερη ακρόαση σήμερα, που θα καταγράψει την κατάσταση, θα κάνει έναν απολογισμό. Θα ακούσουμε διάφορες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και ειδικού έτσι θα μπορέσουμε να συζητήσουμε πράγματα τα οποία δεν έχουν ακόμα λυθεί, που όμως θέλουμε να λυθούν με καλό, με αποτελεσματικό τρόπο όσο περισσότερο γίνεται, έχοντας υπόψη μας ένα πράγμα. Τη φιλοδοξία μας να κάνουμε πράγματα καλά και θετικά για τους κοινούς ανθρώπους, για τους πολίτες μας. Τόσο στον Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το πετύχουμε αυτό, σας διαβεβαιώ. Συνεπώς, σας ευχαριστούμε που ήρθατε και προσβλέπω στις παρεμβάσεις σας και στη συζήτηση. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Λέει ο πριν στραφώ στον κύριο Κουαλτιέρη, πρώτα κύριε ε, Σπινέλη αν θέλει να πει κάτι. Παρακαλώ. On behalf of Danuta Hubner, okay. who could not be... Ναι, εκ μέρους της Danuta Hubner που δεν μπορεί να είναι εδώ. I thank all the speakers present today. Ευχαριστώ πολύ όλους τους παρόντες ομιλητές. Θα σας πω κάποια θέματα που είναι προσωπικά, έτσι, δεν εκφράζουν ολόκληρη την Επιτροπή μου. Ακόμα δεν έχουμε διασφαλίσει νομική βεβαιότητα για όλα τα δικαιώματα που περιγράφονται στο κοινοτικό δίκαιο. Συνεπώς δεν είμαι πολύ αισιόδοξη. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι χαίρομαι πολύ που το Συμβούλιο στις κατευθυντήριες γραμμές ξεκαθάρισε κάποια πράγματα για μεταβατική περίοδο κατά την οποία οι πολίτες θα μπορούν να ε, χαίρουν των ίδιων δικαιωμάτων. Η Τερέσα Μέιλ όμως ε, απέρριψε κάτι τέτοιο. Χαίρομαι επίση για αυτά που άκουσα από τον κύριο Μπαρνιέ. Επαρκής πρόοδος δεν σημαίνει πλήρης πρόοδος. Όμως, τα δικαιώματα των πολιτών δεν συμπεριλαμβάνονται στα θέματα αυτά τα οποία παραμένουν σε κρεμότητα, ούτε βάσει των όσων είπε ο Μπαρνιέ στις κατευθυντήριες γραμμές ούτε περιλαμβάνονται στα λιμένα ζητήματα. Και αυτή είναι η ανησυχία μου, ότι αυτό το θέμα θα παρακαμφθεί στο στάδιο αυτό των διαπραγματεύσεων. Και οι δύο πλευρές έκαναν πολύ συγκεκριμένη έκκληση από την αρχή, ότι δεν θα αλλάξει τίποτα για τα εκατομμύρια ανθρώπους. Τώρα λοιπόν υπάρχει μια νέα έκθεση και νομίζω ότι όλοι το καταλαβαίνουμε ότι δεν λύνεται αυτό το πρόβλημα. Ξέρουμε ότι υπάρχουν ζητήματα που παραμένουν σε κρεμότητα και πρέπει να λυθούν. Σίγουρα οι ομιλητέ θα τα αναλύσουν παρετέρω, αλλά ποια είναι, τι γίνεται με τους εταίρους, με τους συντρόφους των ε, πολιτών. Τι γίνεται με το δεσμευτικό χαρακτήρα των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η μελλοντική ελευθερία διακίνησης των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου, η μεταφορά υποχρώσεων και στην πλευρά της Ιρλανδίας. Όλα αυτά αποτελούν ένα μέρος, αλλά είναι σημαντικά θέματα που δεν έχουν επιληθεί ακόμα και πρέπει να γίνουν περισσότερο προκειμένου να καταλήξουμε σε μια συνολική συμφωνία. Για παράδειγμα, σας ζητώ να διαβάσετε το σημείο 58 της κοινή τεχνικής σημείωσης που αναφέρει θέματα που η Επιτροπή θεωρεί εκτός πεδίου της αρμοδιότητάς της όσον αφορά το πρώτο στάδιο των διαπραγματεύσεων. Εγώ θεωρώ ότι αποτελούν αναγκαία στοιχεία προκειμένου να χαίρουν πλήρως οι πολίτες των δικαιωμάτων τους βάσει του ευρωπαϊκού δικαίου. Θυμίζω ότι η Επιβουλή των Λόρδων στην έκθεσή της για το Brexit που είπε ότι τα δικαιώματα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αδιέρετα και δεν είναι δυνατόν να μην μπορεί ένας πολίτης να ζει, να δουλεύει και τα λοιπά σε μια άλλη χώρα. Αν ένα από αυτά καταργηθεί, τότε καταργούνται όλα. Τώρα θέλω να σας πω και κάποια θέματα που πιστεύω ότι θα συζητηθούν σήμερα. Να αποφύγουμε τη διάβρωση των δικαιωμάτων που προσφέρει το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Το άνοιγμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για βήματα που μπορούν να γίνουν στις 27 ε, χώρες, συνταγματικές διαδικασίες δηλαδή, είναι κάτι ιδιαίτερα ανησυχητικό και αντιβαίνει στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Δεύτερον, πρέπει να αποφύγουμε οποιαδήποτε μνήα στο θέμα των επιλογών ζωής γιατί το να είναι, είναι κανείς πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κάτι που απορρέει από ένα νομικό πλαίσιο δεν είναι θέμα επιλογής τα δικαιώματα οπότε πρέπει να μπορεί να ασκήσει κανείς τα δικαιώματά του είναι μια απόλυτα θεμητή προσδοκία και τα δικαιώματα αυτά πρέπει επιμονή μου βάσεως να τυχαίνουν προστασίας Τέλος, επιστήνω την προσοχή σας στην δυνατότητα μη συμφωνίας. Αν κρίνουμε από τις αντιδράσεις της κυρίας Μέης κατευθύνσεις γραμμές του Συμβουλίου, αναρωτιέμαι μήπως θα έπρεπε να προετοιμαστούμε και για ένα τέτοιο σενάριο και να διασφαλίσουμε, αν μη τι άλλο, κάποιες συμφωνίες για τα δικαιώματα των πολιτών και την Ιρλανδία. Σε ευχαριστούμε και φυσικά είναι στην ε, Διευθυντική Επιτροπή του Brexit ε, μέλος η κυρία Ντανίτα Χιούπνε. Αυτό εννοούσα. Ακούμε τους υπέρμαχους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εξ αρχής ε, και εισακούονται αυτά που λένε με δύο τρόπους και το ξέρουν οι βουλευτές που είναι εδώ πέρα. Πρώτον, μέσω των οργανώσεων που το 3 εκατομμύρια Βρετανοί, διάφορες οργανώσεις τώρα εκπροσωπούνται σήμερα και θα τους ακούσουμε. Ε, και στις μεμονωμένες επαφές που είχαμε ως βουλευτές Α, και να πω, παρενθετικά, η Σεσίλια Βίξτρομ ζητά συγγνώμη δεν μπορεί να έρθει και μου ζήτησε να αναφέρω και το ρόλο της Επιτροπής Αναφορών. Είναι κέριος ο ρόλος ε, για την εξέταση των καταγγελιών και θα κάνουμε και μια παρουσίαση. Προβλέπετε στο πρώτο πάνελ ε, ο Γιώργος Παβέντα από την νομική. Ε, ζητά συγγνώμη λοιπόν για την απουσία της Σεσίλια Βίξτρομ. Το Ντίρχαμ. Ε, και επίσης θέλουμε να ακούσουμε ε, για το τι συνέβη στην Διευθυντική Επιτροπή και ε, ποια είναι τα πορίσματα των συζητήσεων και τι πρέπει να κάνουμε. Αυτά είναι τα καλά νέα. Τα κακά νέα είναι ότι σας μοιάζω λίγο αγχωμένος και ανασφαλής. Ε, ξέρετε γιατί, διότι ε, επικαλέστηκε ανωτέρα βία ο Κίφερ Χόφστατ ε, λέγοντας ότι δεν θα μπορέσει κατά πάσα πιθανότητα να έρθει. Όσοι τον ξέρουν, γιατί μας είχε πει ότι θα κάνει μισή ομιλία, 40 λεπτά δηλαδή τουλάχιστον, και θα ξέρουν ότι είναι περίεργο αυτό. και πιστεύω ότι θα καταλάβετε ότι αν είχε επιλογή θα ερχόταν και θα αποντήσουμε φόρο τιμή στο στο έργο του. Αν εμφανιστεί παρελπίδα κάποια στιγμή, ε, φυσικά θα του δώσουμε τη δυνατότητα να μας πει ε, δύο λόγια, αλλά δεν ε, μπορέσε να έρθει και δεν είχε άλλη επιλογή, πιστέψτε μου. Έχουμε παρόλα αυτά από την Διευθυντική Επιτροπή του Brexit ένα μέλος που έχει εργαστεί σκληρότατα και έχει πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα, κυρίως για τα οικογενειακά ζητήματα, γιατί το βίωσα προσωπικά από την Επιτροπή Έκων, ο κ. Γκουαλτιέρη, ε, από τους πιο δραστήριους θα έλεγα στην Επιτροπή Brexit και ε, Και κύριε Γουαλτιέρη, θα σας δώσουμε το λόγο για τα εναρκτήρια σχόλια σας, ε, κυρίως σε σχέση με αυτά που πετύχαμε ε, για τις ρυθμίσεις του διαζυγίου της αποχώρησης και τι πιστεύετε ότι πρέπει να κάνουμε. Κλον, ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια και ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη ΛΥΜΕ, την ΕΜΠΛ, την ε, Χάβκο, ε, που οργανώνουν αυτή την δημόσια ακρόαση. Είναι εξαιρετική ευκαιρία για να κάνουμε έναν απολογισμό για το τι έχουμε από κοινού πετύχει. Θα επανέλθω σε αυτά και να αναφερθούμε σε αυτά που πρέπει ακόμη να γίνουν. Δεν έχει λήξει ο αγώνας μας γιατί εκκρεμούν πολλά βασικά ζητήματα. Όπως ξέρετε ότι ε, σύσσωμο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αναγάγει σε βασική αξία την προστασία των ε, ανθρωπίνων ε, δικαιωμάτων στα προτεραιότητα όχι μόνο στα ψηφίσματά μας αλλά και στις δράσεις που αναλαμβάνουμε, στις διαπραγματεύσεις προκειμένου ξεκαθαρίσαμε ότι ποτέ σε κάποιο περίπτωση δεν θα εγκρίνουμε μια συμφωνία που δεν θα είναι ικανοποιητική ως προς ε, υπό την οπτική γωνία της προστασίας των ε, δικαιωμάτων των πολιτών. Αυτό είναι φιλόδοξο διότι επιδιώκουμε την ε, πλήρη προστασία ή τη διατήρηση του κεκτημένου grandfathering όπως το λέμε ε, για την, ε, τα κοινωνικά δικαιώματα, ε, για εφόρου ζωής, για όλους τους πολίτες που θα υποστούν το, το Brexit. Είναι ιδιαίτερα φιλόδοξο λοιπόν αυτός ο στόχος. Και αρχίζουμε με αυτή την προσφορά του Ηνωμένου Βασιλείου, αυτό εδώ το έγγραφο που σας δείχνω, που πόρο απέχει από αυτό το φιλόδοξο στόχο. Εμείς με πυγμή το διεκδικούμε και η Επιτροπή όμως και τα κράτη-μέλη. Δεν ε, είμαστε μόνοι μας, ασκούμε όμως ιδιαίτερη πίεση και θέλουμε να ευχαριστήσουμε τις οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών που ε, διαδραμάτισαν πολύ σημαντικό ρόλο. Ε, τρία εκατομμύρια Βρετανοί στην Ευρώπη και οι νέοι Ευρωπαίοι. Ε, και άλλες οργανώσεις που θα ακούσουμε στη συνέχεια. Σας ευχαριστούμε ε, που ε, παρουσιάζετε τα ζητήματα και που κάνετε αισθητή την παρουσία σας και τις διεκδικήσεις σας. Και ξαναλέω, ό,τι έχουμε καταφέρει, το έχουμε καταφέρει ως Κοινοβούλιο και όχι σε Επιτροπή Γκρέξη, είτε από τις συναρμόδιες επιτροπές, η ΛΥΜΠΕ ε, που είναι η κυρίως χαρτήλια αρμόδια αλλά και οι άλλες. Η μεταχείριση είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με το Βρετανικό Κοινοβούλιο πάντως και ε, η Επιτροπή Brexit ε, όχι μόνο εξέδωσε μία δήλωση και ε, σε σχέση με τις θέσεις ε, των ε, διαπραγματευόμενων μερών, αλλά και τη σωστή στιγμή όταν είχαμε τις εναλλακτικέ λύσεις μπόρεσε να συμβάλλει στη διαμόρφωση της θέσης φωτέρων των πλευρών και να επηρεάσει την έκβαση των διαπραγματεύσεων. Νομίζω ότι αυτό είναι μια πρότυπη, ένας πρότυπος κοινοβουλευτικός ρόλος. και τα αποτελέσματα είναι επαρκή. Επαρκή θα τα χαρακτήριζα. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι τέλεια. Δεν είμαστε πλήρως ικανοποιημένοι και επαναλαμβάνω ότι παραμένουν ανοιχτά πολλά ζητήματα. Δηλαδή, σε σχέση με την συνεπή εφαρμογή της κοινή ε, έκθεσης και σε σχέση με προσθήκη ζητημάτων που αυτή τη στιγμή απουσιάζουν. Δεν ε, το γιορτάζουμε δηλαδή σήμερα εδώ. Όμως, επειδή ακούω και προπαγάνδα, ε, ότι ήταν με δική τους πρόταση, όχι, δεν έχουμε φτάσει ε, στο επιθυμητό, αλλά έχουμε καταφέρει πολλά. Έχουμε καταφέρει να καλύψουμε όχι μόνο τους πολίτες αλλά και τα μέλη των οικογενειών τους και τα παιδιά που ακόμη δεν έχουν έρθει στον κόσμο. Δεν έχουμε καλύψει ολόκληρο το πεδίο, αλλά σχεδόν. Και το περιεχόμενο, πέρα από την κείμενη νομοθεσία, είναι όχι μόνο τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται στις ε, συνθήκες ε, και στο ευρωπαϊκό δίκαιο, αλλά και στην ομολογία του δικαστηρίου. Δηλαδή, αν κάποια εθνική νομοθεσία, η Βρετανική εννοώ, έτσι, με περίπτωση, αν αποκλίνει από ε, τα την μενή νομοθεσία, έτσι η αναφορά στους κανονισμούς στις οδηγίες στην ονομολογία ε, καθίσταται άκυρη, διότι ε, πρόκειται για άμεση ισχύ, έτσι. Άμεση ισχύ ε, του ενωσιακού δικαίου. Λοιπόν, αυτά τα δικαιώματα κατοχυρώνται δυνάμει του ενωσιακού δικαίου. Κατοχυρώνται μέσα στο δίκαιο και στην νομολογία του δικαστηρίου αυτά τα δικαιώματα η νομολογία κατοχυρώνει ε, φόρου αυτά τα δικαιώματα και μετά έχουμε και την διάταξη ε, εκνοής της ισχύω για, για τα, τις μελλοντικές ε, όμως ε, ε, Όλο το φάσμα των δικαιωμάτων, γιατί και τα κοινωνικά αποζήτησαν στην αρχή. Ασκήσαμε πίεση και τελικά Έχουμε λοιπόν τα κοινωνικά δικαιώματα μετά την πίεση που ασκήσαμε. Έχουμε τα μελλοντικά τέκνα, το είπαμε αυτό. Ήταν αγώνας, μάχη και ε, νίκη που κατήγαγε το κοινοβούλιο. Τώρα έχουμε και τους ανιώντες, γιατί μην τους ξεχνάμε. για μας ε, αυτό το σημείο εκκρεμεί, είναι ανοιχτό. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα. Συνοπτικά, δύο είναι τα τεινά που θα κάνουμε. Πρώτον, θα ελέγξουμε αν το σχέδιο για το οποίο εσείς ε, ελπίζουμε θα δώσετε τη συγκατάθεσή σας ε, συνάδει με αυτά που αναφέρει το τεχνικό σημείωμα και η συνολική συμφωνία. Περιμένουμε λοιπόν. Κάθε γραμμούλα, κόμμα, όλα τα ελέγχουμε επακριβώς. Οτιδήποτε αποκλίνει από αυτά που αναγράφονται στην κοινή έκθεση θα το εντοπίσουμε. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία διότι έχουμε επαρκές επίπεδο λεπτομέρειας και αυτό γιατί, διότι έχουμε, είμαστε μεθοδικοί εμείς, ε, είμαστε ε, συνεκτικοί στην προσέγγιση μας και τώρα τα έχουμε κατοχυρώσει όλα. Δεν τα έχουμε όλα, αλλά ένα μεγάλο κομμάτι. Και τα καταφέραμε διότι στο τελευταίο ψήφισμα λέγαμε ότι όχι, θέλουμε στην ε, συμφωνία αποχώρησης, μέσα στη συνθήκη δηλαδή, αυτό το κομμάτι της συνθήκης αποχώρησης, να, αποχώρησης, να συνταχθεί τώρα. Θέλουμε να δούμε τη διατύπωση, τα άρθρα, τη, τα εδάφια, τα κόμματα, ό,τι θα είναι νομικό δεσμευτικό, γιατί ο μηχανισμός της άμεση ισχύω είναι ακριβώς αυτός που εννοούσαμε και ε, να προβλέπεται ο προσφορότερος ρόλος για το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τη διαδικασία, διοικητική διαδικασία θα επανέλθω σε αυτό. ο, ο ετών θα έχει πάντοτε το πλεονέκτημα ε, σε περίπτωση αμφιβολίας. Αυτό το έχουμε κατοχυρώσει και θα το ε, διευκρινίσουμε. Ε, διότι ξέρουμε ότι η συντακτική δουλειά ε, γίνεται τώρα και ελπίζουμε να περατωθεί σύντομα και φυσικά θα ε, κάνουμε την επαλήθευση με εσάς. Ε, και μέχρι όπου καταλήξουμε σε συμπεράσματα για τη συμφωνία θα προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε και τα επιπρόσθετα σημεία που διεκδικούμε. Η μελλοντική σύζυγη σύντροφοι και η συγκρότηση συγκεκριμένου μηχανισμού για την διοικητική εφαρμογή της Συμφωνίας Αποχώρησης, ε, διότι προβλέπεται πρέπει να προβλέπετε μάλλον ότι πρέπει να είναι ε, σύντομη, απλή φιλική προς το χρήστη και ε, προσαρμοσμένη ως προς τις ανάγκες η διοικητική διαδικασία. Αυτό τι σημαίνει που σας λέω τώρα. Πολλά. Γιατί στο 17 εδάφιο Γ που λέει ότι ωραία, υποβάλλετε εσεί σε αίτημα ή δυνάμει του ενωσιακού δικαίου δικαιούστε να υποβάλλετε έτοιμο. Μάλιστα. Ε, χρειάζεται δήλωση. Πώς θα το εφαρμόσετε αυτό το 17 γ ότι και να πάει στραβά, θα πρέπει να προβλέπει ο μηχανισμό για επανόρθωση. Καταλαβαίνετε. Γι' αυτό πρέπει να έχει χαρακτήρα δήλωση, ε, ε, να μην έχει μόνο χαρακτήρα δήλωση. Διοικητικά, συγκεκριμένα πώ θα εξελιχθεί η διαδικασία. Έχετε πέντε χρόνια για να υποβάλλετε την ε, αίτησή σα. Και αν αυτό επικαλύπτει την ε, μεταβατική περίοδο, τι θα γίνει, πώ ακριβώ, ποια αλληλεπίδραση θα υπάρχει με τη μεταβατική περίοδο, Πώς θα διασφαλίσουμε εμείς ότι όλα καλύπτονται αυτά τα δύο χρόνια που προβλέπονται εδώ πέρα για την υποβολή αίτησης. Ε, ε επίσης, ε, ουσιαστικότατο ζήτημα, η ανεξάρτητη αρχή θέλαμε ε, να εκπροσωπεί και τον ε, ετούντα τον πολίτη ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων και να μπορεί να καταθέσει και προδικαστικό στο δικαστήριο. Όχι μόνο λοιπόν οι πολίτες, δεν θα έχουν μόνο εκείνη τη δυνατότητα να προσφεύγουν στα εθνικά δικαστήρια, αλλά αυτή τη ανεξάρτητη αρχή θα τους εκπροσωπεί και θα πρέπει να έχετε δυνατότητα ενώπιον της δικαιοσύνης να τους εκπροσωπήσει και όχι γενικόλογες δηλώσεις. Πώς θα γίνει αυτό διότι ο... ποιος είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αληθεύει ότι είπαν οι ομόλογοι μας ότι ε, θέλετε να υπάρχει δυνατότητα αλλά να μην είναι υποχρεωτικό. Ναι. Ε, και στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε αυτό το θέμα με τους δικαστές αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Πρέπει να είναι ανεξάρτητος ο φορέας ώστε να εκπροσωπεί τον πολίτη. Και αν κανείς άλλος δεν προσφύγει στα εθνικά δικαστήρια να μπορεί να το κάνει αυτή η ανεξάρτητη αρχή. Και γι' αυτό σα λένε σημαντική η συγκεκριμένη διατύπωση και στην κοινή δήλωση πρέπει να αναφέρεται και να δούμε στην πράξη πώς θα εφαρμοστεί. Άλλα δύο ζητήματα έχουμε εξίσου ουσιαστικά. Ελεύθερη κυκλοφορία στις, ε, στα 27 κράτη-μέλη και εμείς είμαστε υπέρ οι Βρετανοί πολίτες να πηγαίνουν μετακινούνται ελεύθερα. Ξέρετε ότι ε, δεν έχει την ίδια θέση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που σαν καθεν... Ήμασταν ξεκάθαροι και δεν πρόκειται να αλλάξουμε στάση. Και τέλος. Εάν στη μεταβατική περίοδο θα παραταθεί ε, η καθεστική ατάξη, ε, οτιδήποτε άλλο απλώς θα συνεχίσει να ισχύει. Και Τέλη 2020 λέει η οδηγία. Μήπω παραταθεί και αυτή η προθεσμία. τέλο. πάντων, ας μην συζητήσουμε ημερομηνία τώρα, αλλά συζητήσουμε επί τη αρχής. Όλα θα πρέπει να, να παραταθούν. Για να καλυφθεί η ελεύθερη μετακίνηση, ελεύθερη κυκλοφορία των ανθρώπων και όλες αυτές οι διατάξεις και η προκαθορισμένη ημερομηνία, όλα αυτά αναλόγως θα τροποποιηθούν, καταλαβαίνετε ακούσαμε και τη δήλωση Τερέζα Μέη. Αυτή δεν είναι η τοποθέτηση της κυβέρνησης. Έχουμε άλλο ένα ζήτημα να συζητήσουμε. Θα ε, ξαναδείξουμε, ε, θα επιδείξουμε συνέπεια και πυγμή και πάλι ως κοινοβούλιο. Λοιπόν, σε αυτήν την οδηγία που ενέκρινε για τη μετάβαση το Συμβούλιο, μην ξεχνάμε ότι εμεί είμαστε από αυτού που ζητούσαμε από τον Παρνιέ όχι να το βάλει μέσα στην οδηγία η Επιτροπή αυτό το στοιχείο. Δηλαδή ότι κατά τη μετάβαση οι πολίτες θα είναι σε αυτή τη μετάβαση. Δηλαδή το status quo καλύπτει ε, τους πολίτες και όλα παρατείνονται. Και αυτό από θέση του Κοινοβουλίου είναι θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι ομόφωνα εγκρίθηκε από το Συμβούλιο. Τώρα είναι κόκκινη γραμμή, τώρα δεν ε, ανακαλείται αυτό. Και θα επηρεάσει και τα επόμενα βήματα. Αυτά ξεκάθαρα λοιπόν δείχνουν ότι πραγματικά πρέπει να είμαστε περήφανοι γιατί έχουμε πετύχει. Έχουμε επικρίσεις και όλοι μπορούν να βρουν τη λεπτομέρεια που δεν τους αρέσει, αλλά Έχουμε λόγους να είμαστε υπερήφανοι γιατί όλοι τα καταφέραμε μαζί και χωρίς όμως τη συνεπή εφαρμογή των αρχών που είναι στην κοινή έκθεση παρόλα αυτά η συμφωνία δεν θα είναι καλή. Δεν κάναμε ένα πρώτο βήμα μόνο. Και θα είναι αποφασιστική σημασία οι εξελίξει. Χρειάζεται αποφασιστικότητα από το Κοινοβούλιο. Πρέπει να σα ακούσουμε τι έχετε να πείτε. Μα ενδιαφέρουν οι απόψεις γιατί τις επόμενες κρίσιμε εβδομάδες και μήνες αυτά θα μετρήσουν. Σα ευχαριστούμε. Κάποια από αυτά στις πληροφορίες θα βρίσκονται στην ιστοσελίδα μετά από την ακρόαση. Αν εμφανιστεί ο κύριος Φερχόφστατ ε, θα του δώσουμε το λόγο. Ο Ρομπέρτο ανέφερε την διευθύνουσα ομάδα του Brexit και τα επιτέγματά της. Είναι πολύ δύσκολο να τα ζυγίσει κανείς όλα αυτά με τα όσα απομένουν και όλη την αβεβαιότητα και τις ανησυχίες. Εσκεμένα λοιπόν συνδυάσαμε εμείς τη σημερινή ακρόαση με τον αριθμό των ευρωβουλευτών που βρίσκονται εδώ και χαίρομαι που πολλοί κόσμος έχει έρθει εδώ παρότι είναι πέντε απόγευμα. Ζητώ συγγνώμη αλλά έγιναν πολλές οργανωτικές προσπάθειες όπως είπε και ο Ρομπέρτο για να επιτύχουμε όσο επιτύχαμε σε αυτό το πρώτο στάδιο. Πρώτος ομιλητής από το πρώτο πάνελ είναι η κυρία Ανλόρ Σκόη, ιδρυτικό μέλος της ομάδας ε, The Three Million για τους Ευρωπαίους πολίτες ε, που κατοικούν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ανλόρ, αν θέλετε μπορείτε να ξεκινήσετε. Αν μιλήσει ο καθένας για 10 λεπτά ή λιγότερα θα μπορέσουμε να ακούσουμε μετά και τις ερωτήσεις των ε, Ευρωβουλευτών. Όσο πιο συντομίστε τόσο πιο γρήγορα θα μπορέσουμε να κάνουμε και το διάλογο. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, ε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές, ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία που μου δίνετε να σας παρουσιάσω τη σημερινή κατάσταση των Ευρωπαίων πολιτών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, επόμενη διαφάνεια παρακαλώ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ζητήσει πλήρη δικαιώματα ε, των Ευρωπαίων ε, πολιτών όπως έχουν αυτή τη στιγμή να συμπεριληφθούν στη συμφωνία έχει σημειωθεί πρόοδο στην πρώτη φάση ωστόσο ελλειπής σε σχέση με την πλήρη προστασία θα σας δώσω κάποια βασικά σημεία Όσον αφορά τη διαδικασία εγγραφής, ε, ε, ο κανονισμός της 20 Μαΐου 2017 λέει ότι οποιοδήποτε έγγραφο θα επιβεβαιώνει απλά τα δικαιώματα κάποιου ατόμου. Ωστόσο, αυτά που συμφωνήθηκαν το Δεκέμβριο, ότι τα κράτη-μέλη μπορούν είτε να κάνουν μια ε, δήλωση, είτε μια συστατική διαδικασία που σημαίνει ότι θα πρέπει κανεί να, υποβα... να αιτηθεί τα δικαιώματά του. Αυτό δεν υπερβαίνει απλά την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, αλλά δεν βοηθά στην προστασία όλων των δικαιωμάτων. Ε, έτσι λοιπόν ε, θα είναι δύσκολο να επιτευχθεί η μόνιμη εγκατάσταση, το οποίο όχι απλά υπολείπεται των πλήρων δικαιωμάτων, αλλά θα έχει σοβαρέ συνέπειε για όσου ζουν στο, Ευρωπαϊκό, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το πρόβλημα είναι ότι η μόνιμη εγκατάσταση πρέπει να ειδωθεί στο πλαίσιο του μεταναστευτικού νόμου στο Ηνωμένο Βασίλειο. με όποιο τρόπο και να το κοιτάξει κανεί, η μόνιμη εγκατάσταση παρέχει δικαιώματα, δεν τα επιβεβαιώνει. Σύμφωνα με του κανόνε μετανάστευση του Ηνωμένου Βασίλειου, δεν είναι απλά μια δήλωση. Οι συνέπειε τη μη τήρηση όλων των απαιτήσεων ε, τη μόνιμη εγκατάσταση ή κάποιο λάθο ε, στη διαδικασία αίτηση μπορεί να έχει σοβαρέ συνέπειε για του ενδιαφερομένου μπορεί να ρίξει τους ετούντες σε ένα εχθρικό περιβάλλον και με κινδύνο απέλασής τους. Επίσης θα γνωρίζετε ότι το Ρωμανό Βασίλειο, η κυβέρνησή του, έχει εισάγει νομοθεσία με εξαιρέσει ε, για θέματα προστασία δεδομένων. Ε, η πρόσβαση στα δεδομένα που έχει το Υπουργείο Στερικών, η δυνατότητα να κατανοήσει ο πολίτης τα λάθη που έχουν κάνει οι μεταναστευτικές αρχές, ε, δεν θα είναι τέτοια και συνεπώς ε, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα έχει και η κυβέρνηση δεν θα έχει τον, ε, την υποχρέωση να τα χειριστεί όλα αυτά νόμιμα. Αυτό αντίκειται στην προστασία των πολιτικών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίσης, μην ξεχνάμε τον βαθμό σφαλμάτων που έχει πραγματοποιήσει το Υπουργείο Εσωτερικών και φανταστείτε τι θα γίνει με τον αυξανόμενο αριθμό αιτήσεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί όλο αυτό σε ένα διοικητικό εργαλείο το οποίο θα δημιουργήσει προβλήματα σε ανθρώπους που θα χρησιμοποιήσουν την διαδικασία προσφυγών κατά αποφάσεων μεταναστευτικών. Οι έλεγχοι ασφαλείας ε, μας οδηγούν στο ερώτημα ότι πώς ε, θα γίνεται η νέα διαδικασία που αντίκειται στη σημερινή ελεύθερη κυκλοφορία και πώς θα γίνει αυτή η έλεγχη να είναι συστηματική αντίθετα με ό,τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Επίση, έτσι δημιουργείται άλλο ένα στρώμα διοικητικού φόρτου στο Ηνωμένο Βασίλειο, επειδή κάθε ετών θα πρέπει να ελέγχεται εκτενώ. Η οργάνωση The Three Million στην, ε, είναι αντίθετη με την εθελοντική εγγραφή ε, στο σύστημα μόνιμης εγκατάστασης. Δεν έχει νόημα να υπάρχει ένα σύστημα χωρίς νομική ε, ισχύ μέχρι ότου επικυρωθεί η συμφωνία αποχώρησης. Θα υπάρχουν διαφορές μεταξύ του θελοντικού συστήματος και του τελικού κειμένου. Επίσης δεν θα υπάρχει κανένας νομοθετικός μηχανισμός για ετούντε ε, που απορρίφθηκαν. Υπάρχει πιθανότητα όσοι απορρίφθηκαν να αποθαρρυνθούν από το να ξαναετηθούν αναξάρτητα από το σύστημα που θα έχουμε τελικά διότι θα φοβούνται την απόρριψη. Το οποίο σημαίνει ότι μπορεί να ε, αποτελέσουν παράνομους μετανάστες με ε, κίνδυνο απέλασης. Όσον αφορά την νόμιμη κατοικία ε, υπάρχει πολύ ασάφεια και σύγχυση για το πώς το Ηνωμένο Βασίλειο ερμηνεύει αυτά τα κριτήρια. Υπάρχει πιθανότητα και εκεί απορρίψης αιτήσεων. Με όλα αυτά δεδομένα. Υπάρχει κίνδυνος πολλές ομάδες πολλά άτομα να μείνουν πίσω για διάφορου λόγου. Το πρώτο είναι θέμα δικαιωμάτων. Πολλές κατηγορίε δεν καλύπτονται όπως ε, ε, συγγενείς που επιστρέφουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, ε, κόσμος που έλειπε από την τοποκατοικία του την ημέρα του Brexit κτλ. Το άλλο είναι ζήτημα διεκπαιρεωτικό. Ηλικιωμένοι άνθρωποι με αναπηρίες, παιδιά, θύματα εμπορίας, άστεγοι, όλοι έχουν κινδυνό να μείνουν πίσω διότι θα είναι δύσκολο να αποδείξουν ότι είχαν νόμιμη κατοικία. Η πρακτική βοήθεια που προτείνει το όνομα Βασιλείο είναι ανεπαρκής και ε, από τη φυστής και σε απόψη αντικειμένου. Το πώ το Home Office θα ασχοληθεί με αυτά τα ζητήματα δεν μα εμπνέει η εμπιστοσύνη. Ενώ θα έπρεπε, θα θέλαμε να υπάρχει ομαλή αντιμετώπιση, διαφανή αντιμετώπιση και ισότιμη. Ωστόσο υπάρχει μία λύση. Η εναλλακτική πρόταση των 3 million δείχνει ότι υπάρχει ένα πιο δίκαιο, απλούστερο και πιο ευέλικτος τρόπος, εναλλακτικός ε, σε σχέση με το settled status στην μόνιμη εγκατάσταση. Η οργάνωσή μα ανησυχεί για την ερμηνεία που πιστεύει ότι είναι λανθασμένη από το Ηνωμένο Βασίλειο ε, και ότι αυτό θα συνεχιστεί όταν θα αναχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεπώς θα απαιτηθεί ιδιαίτερη προστασία των δικαιωμάτων μα. Πρώτα απ' όλα θέλουμε να προστατεύσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο τα δικαιώματά μα. Θέλουμε λοιπόν να ασκήσετε πίεση Επίσης, η σημερινή νομική βοήθεια στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι ε, ιδιαίτερα δύσκολη για ανθρώπους περιορισμένων εισοδημάτων. Τρίτον, χρειάζεται παρακολούθηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε το ε, Βρετανικά δικαστήρια να ερμηνεύουν σωστά τα κομμάτια που αφορούν τους πολίτες στη Συμφωνία Αποχώρησης. Τι γίνεται με τις μελλοντικέ ε, με τους μελλοντικούς συντρόφους, οι οποίοι θα πρέπει να προστατεύονται. Αυτό θα πρέπει να ισχύει και για τους 27 ε, εθνικότητες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τους Βρετανούς πολίτες στην Ευρώπη που μπορεί να θέλουν να επιστρέψουν στο μέλλον με ε, εταίρου, με συντρόφους τους στο Ενωμένο Βασίλειο. Οι επιπτώσει θα είναι τεράστιε δυσανάλογε για τι νέε γενιέ, Το ίδιο και για του πολίτε, οι οποίοι μετά από ένα διαζύγιο ή το θάνατο των συντρόφων του θα θελήσουν να ξαναπαντρευτούν μετά από τον Brexit. Όλα αυτά μας οδηγούν να θυμηθούμε τα θεμελιώδη στοιχεία της ευρωπαϊκής ηθαγένειας. Το Ηνωμένο Βασίλειο ισχυρίζεται ότι θα έχει ίση πρόσβαση ε, στα δικαιώματα και στις υπηρεσίες μετά τον Brexit, αλλά υπάρχει πολλή αβεβαιότητα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Όλο και περισσότεροι πολίτες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης μας λένε ότι έχουν δυσκολίες ε, να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και πρέπει να αποδείξουν το δικαίωμα κατοικίας τους επίσης βλέπουν περιορισμό της ε, ελευθερίας ε, κυκλοφορίας. Βλέπουμε με λύπη μας ότι η πραγματική άσκηση των δικαιωμάτων βασίζεται σε κάποιες επιλογές σε απαρελθούσες της ζωής. Αυτό είναι λάθος. Δεν θα έπρεπε να γίνεται έτσι. Θα έπρεπε οι αποφάσεις να λαμβάνονται βάσει μελλοντικών επιλογών, όχι αντίστροφα. Υπάρχει ένα τεράστιο ερωτηματικό όσον αφορά τις τα επαγγελματικά και ακαδημαϊκά προσόντα μετά τον Brexit. Ποιοι θα έχουν τη δυνατότητα να δουλέψουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην, Ηνωμένη, στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να συμμετέχει στο μηχανισμό Μπολόνια μετά τον Brexit κάποια στιγμή, αλλά τι θα γίνει μέχρι τότε. Πολλά από τα προνόμια της ελευθερίας κυκλοφορίας σχετίζονται περισσότερο με την χώρα κατοικίας και όχι με την εθνικότητα. Η Ευρωπαίοι πολίτες που θα ζουν στο ΕΒ μετά από τον Brexit θα χάνουν πολλές ευκαιρίες διότι το Ηνωμένο θα έχει γίνει τρίτη χώρα η συμφωνία αποχώρησης θα πρέπει να μας προστατεύει να μην γίνουμε πολίτες τρίτης χώρας ακόμη και μετά την αναχώρηση. Συνοπτικά, στη φάση ανασυνοηθήκαμε ε, πράγματα τα οποία δεν θα μας προστατεύουν επαρκώς. Υπάρχουν διάφορες ε, διάφορα σκοτεινά σημεία, οπότε δικαιώματα των Ευρωπαίων στο Ηνωμένο θα είναι περιορισμένα. Η μόνιμη εγκατάσταση θα μας ρίξει σε ένα εχθρικό περιβάλλον, θέτοντας εκατοντάδες χιλιάδες Ευρωπαίους πολίτες σε κίνδυνο που και μπορεί να μην ε, τους επιτρέπεται να παραμείνουν στο Ρωμανοβασίλειο. Βασίλειο. Μην ξεχνάμε ότι η πρώτη αρχή βάσει της οποίας πρέπει να γίνουν διαπραγματεύσεις για τα δικαιώματα των πολιτών, αφορά πρωταρχικά τις ζωές των ανθρώπων πριν από οποιαδήποτε εμπορική συμφωνία και πριν από οποιαδήποτε διαδικασία. Πρέπει να βασιστούμε στα δικαιώματά, δικαιώματά μας όπως θεσπίζονται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, στην προστασία τους ώστε να συνεχίσουμε να ζούμε όπως ζούσαμε μέχρι σήμερα. Όπως πολλές φορές έχουν δηλώσει και το ΕΒ και η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από το δημοψήφισμα. Ευχαριστούμε. Uh, Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίασή σας αυτή. Και ο κύριος Έλμαρ Μπροκ ήρθε, που και αυτό συμμετέχει στη Διευθύνουσα Επιτροπή για τον Brexit. Δεν το είπα στην αρχή. Όχι, δεν φταίτε εσείς, είσαστε ευπρόσδεκτος και ελάτε και εδώ. Θα πάρετε το λόγο αργότερα. Μιλάω για την διευθύνουσα αυτή ομάδα, γιατί όσοι συμμετέχουν σε αυτή περνάνε ώρες και ώρες προσπαθώντας να βοηθήσουν και να δουν τι πρέπει να γίνει ακόμα εν ώψη του Brexit, όπως τα ακούσαμε και από την οργάνωση 3 Million. Τώρα, θα ακούσουμε την Jane Golding, που είναι πρόεδρος της οργάνωσης Βρετανή την Ευρώπη. Αποτελείται από 10 ομάδες Βρετανών πολιτών που ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε και κύριοι Ευρωβουλευτές. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ευκαιρία που μας δώσατε σήμερα. 1,2 εκατομμύρια Βρετανοί ζουν στην Ευρώπη σήμερα. 80% αυτών βρίσκονται σε ηλικία εργασίας. Το 1 τρίτο είναι στην ηλικία 30 με 49. Όπως και από την οργάνωση 3 Million που ακούσαμε όλοι οι Ευρωπαίοι, οι παιδιά της Ευρώπης που εποφεληθήκαμε από όλες τις ευκαιρίες που απορρέουν από τα δικαιώματα όταν έχει κανείς την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια. Και περιμένουμε από εσά και την Ευρωπαϊκή Ένωση να προστατεύσει τα δικαιώματά μας και χαιρόμαστε για την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις διαπραγματεύσεις όσον αφορά τις αρχές. Άρχισαν λοιπόν οι διαπραγματεύσεις και βέβαια αναπόφευκτα κατέληξαν σε επιδείνωση τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τα δικαιώματά μας, δεδομένου ότι και το Ηνωμένο Βασίλειο από τη δική του την πλευρά έκανε τις δικές του προτάσεις και χρειάστηκε να καταλήξουμε σε συμβασμούς. Όμως, όπως είπε και ο κύριος Γκολτιέρη, έγινε κάποια πρόοδος για τα δικαιώματα των πολιτών το 2017 που οδήγησε στην κοινή έκθεση της 8 Δεκεμβρίου. Αυτό όμως που είναι γνωστό της πάση σήμερα είναι ότι έχει υπάρξει κάποια πρόοδος προκειμένου να μπορέσουμε να περάσουμε στο δεύτερο στάδιο των διαπραγματεύσεων αφήνοντας πολλά θεμελιώδη ζητήματα ανοιχτά ακόμα. Θα επαναλάβω αυτά που είπε και η συνάδελφος, η Αν Λόρ Ντόσκο από την οργάνωση 3 Million, ότι είμαστε απογοτευμένοι από την κοινή έκδοση, γιατί εκεί τα δικαιώματά μας προσδιορίζονται ως βασισμένα σε επιλογές ζωής αυτό ε, επειδή στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις οδηγίες διαπραγματεύσεων της 23ης Μαΐου του 2017 ήταν η προστασία ε, του καθεστώτος και των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ενωσιακή νομοθεσία την ημέρα της αποχώρησης. Οπότε τα δικαιώματά μας πρέπει να προστατεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι τις επιλογές της ζωής μας. Όπως είπε και η Άννα Λόρ, τα δικαιώματα οδηγούν σε επιλογές ζωής. Συνεπώς, ε, όλα αυτά πού μας πηγαίνουν στις διαπραγματεύσεις, πώς θα προστατευτούν τα δικαιώματά μας. Έχει υπάρξει κάποια πρόοδος όπως είπαμε, υπάρχει συμφωνία σε διάφορα τεχνικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αμοιβαιότητα της ε, υγειονομικής περίθαλψης και της κοινωνικής περίθαλψης. Όμως αυτά έχουν να κάνουν με τους ανθρώπους που είναι οικονομικά ανενεργοί, που είναι μόνο το 20% των Βρετανών στην Ευρώπη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πολλά θεμελιώδη ζητήματα παραμένουν ανοιχτά, κυρίως για τους πιο νέους. Και αυτό έχει να κάνει και με τους Βρετανούς και με εδώ και με τους Ευρωπαίους στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κάνει ψήφισμα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 13 Δεκεμβρίου όπου αναφέρθηκε σε πολλά από αυτά. Ένα από αυτά είναι το κατά πόσο οι Βρετανοί στην Ευρώπη θα εξακολουθούν να έχουν το δικαίωμα ελεύθερη κυκλοφορία. Πολλοί βασίζονται σε αυτή την ελευθερία διακίνηση, γιατί δουλεύουν αλλού, ζουν αλλού και αναρωτιόνται τι θα γίνει και πώς θα κερδίσουν το ψωμί τους μετά το Brexit. Πρέπει να υπάρχει ελεύθερη κυκλοφορία και μετά, γιατί οι Βρετανοί πολλές φορές δουλεύουν στο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά σε διάφορες χώρες. Πώς θα κατοχυρωθεί αυτό το δικαίωμα και μετά. Οι επιπτώσεις της μείωσης της ελεύθερης κυκλοφορίας ε, θα πλήξει επαγγελματικά προσόντα, οικονομικά δικαιώματα και σημαίνει ότι κάποια επαγγέλματα δεν θα αναγνωρίζονται καν πια και αυτά που θα αναγνωρίζονται ε, θα είναι πιο περιορισμένα. Πολλοί Βρετανοί πολίτες πήγαν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες ακριβώς επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια επικράτεια χωρίς εσωτερικά σύνορα. Και δεν πρόκειται μόνο για τους δικηγόρους εδώ ή τους ε, ε, οδηγούς φορτηγών ή αυτούς που απασχολούνται στην πληροφορική έχει να κάνει με πάρα πολλούς. Επίσης μετά από αυτά που είπε η Ανλόρ, η συμφωνία που επετέφθηκε για το πώς θα διασφαλίσει το καθεστώ τους οι πολίτες μετά την ε, αποχώρηση ε, τι κάνει, δέχεται την πρόταση του Ηνωμένου Βασιλείου, δηλαδή να μπαίνουν όροι δεν επιμένει δηλαδή σε μία σαφή δήλωση για τα δικαιώματα αυτά. Δηλαδή θα είναι οι πολίτες οι οποίοι θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι έχουν ε, κάποια δικαιώματα. Κάτι το οποίο μπορεί να καταστεί πάρα πολύ δύσκολο για ορισμένου που βρίσκονται σε μια χώρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και έπειτα υπάρχει και η γραφειοκρατία που και αυτή κάνει λάθη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 μπορεί να επιβάλλει στους ε, Βρετανούς επίσης περιορισμούς. Και αυτό ήταν κάτι που προσθέθηκε τελευταία στιγμή, χωρίς να υπάρξει διαβούλευση προηγουμένω. Νιώθουμε λοιπόν ότι το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τη 13η Δεκεμβρίου σωστά έλεγε ότι θα έπρεπε να το ξαναδούμε. Και οι Βρετανοί πολίτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εντελώ στο σκοτάδι για το κατά πόσο τελικά θα εφαρμοστεί όχι αυτή η επιλογή. Όπως επίση είπε η Ανλό, θα υπάρξουν περιορισμοί και στην επανένωση οικογενειών για τα μελλοντικά μέλη των οικογενειών και στις δύο περιπτώσεις. Και τι θα γίνει με αυτούς που επιστρέφουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις οικογένειές τους. Και μια που μιλάμε και για τις πιο νέες γενιές, δεν έχει αποσαφανιστεί τι θα γίνει με τους φοιτητές. Δεξιότητες, ε, προσόντα, διπλώματα κλπ. μετά το Brexit. Και επιπλέον από όλα αυτά τα ουσιαστικά ζητήματα, όπως έχουμε ήδη πει, τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί αν δεν συμφωνηθούν όλα. Και πώς θα κατοχυρωθούν τα δικαιώματα των πολιτών στο υπόλοιπο των διαπραγματεύσεων εφόσον ε, τώρα παραμένουν σε κρεμότητα. Τέλος, σε αντίθεση με ό,τι γίνεται για την Ιρλανδία, δεν υπάρχει σαφής ε, διευκρίνηση ότι θα συνεχιστούν διαπραγματεύσεις για τα δικαιώματα των ε, πολιτών. Οπότε πολύ πιθανόν το θέμα αυτό να ξεχαστεί, να παρακαθεί. Αυτές είναι οι νομικές και οι πολιτικές επιτυχίες των διαπραγματεύσεων όσον αφορά τα δικαιώματα των πολιτών που ανέφερα μέχρι τώρα. Τι γίνεται όμως με την ανθρώπινη πτυχή, με τις κοινωνικές πτυχές των ε, Βρετανών ε, και των υπόλοιπων Ευρωπαίων. Το ευρωπαϊκό σχέδιο βασίζεται στην ειρήνη, τη συνεργασία, την ελεγγύη και την κοινωνική διάσταση. Η καγκελάριος Μέρκελ στον Ταβός μίλησε την προηγούμενη εβδομάδα για τη συνεργασία, την αλληλεγγύη. Και εγώ θέλω να μιλήσω για την Ευρώπη σαν μια ένωση ανθρώπων. Το 1945 ο πατέρας μου που ήταν τότε 20 ετών ήρθε στην Ευρώπη με τις συμμαχικές δυνάμεις και την ίδια χρονιά ο πεθερός μου που τότε ήταν 16 επέζησε το βομβαρδισμό της Δρέζης. Δεν συναντήθηκαν ποτέ, αλλά και οι δύο με διαφορετικό τρόπο ελπίζανε σε μια καλύτερη Ευρώπη για τα παιδιά τους και τα γόνια τους. 50 χρόνια αργότερα ο, πατέ... ο πεθερός μου έφερε τον άντρα μου στις Βρυξέλλες μέσα σε ένα λάντα για να έρθει και να ακολουθήσει την ίδια μαθητεία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που παρακολουθούσα κι εγώ. Και έτσι γνωριστήκαμε. Ήταν η δεύτερη φουρνιά Ανατολικογερμανών μετά την κατάρρευση του τείχους του Βερολίνου. Εκεί γνωριστήκαμε. Τα παιδιά μας είναι τυχερά, δεν θα χάσουν την ευρωπαϊκή Ιθαγένεια αλλά δεν ε, ανήκουν όλα τα παιδιά σε αυτή την κατηγορία προστατευμένων παιδιών και το αν τελικά είναι τυχερά ή δεν είναι, είναι εντελώ τυχαίο υπάρχει ομάδα ανθρώπων που καλή την πίστη ε, μετακόμισε, μετακινήθηκε πιστεύοντας στα δικαιώματα που του προσέφερε η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Οικοδόμημα. Η αλληλεγγύη, η αίσθηση του ανήκειν σε μία ομάδα ακριβώς είναι έκφραση του ευρωπαϊκού σχεδίου. Πρόκειται για μια κοινότητα Ευρωπαίων που έχουν ένα κοινό μέλλον, ένα μέλλον που τους ενώνει κάπου. Και αυτό είναι τα δικαιώματά τους. Τώρα πρέπει να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών και όχι να τα αποδυναμώσουμε. Αν απογοητευτούμε τώρα, καταλαβαίνετε ότι πάνε οι ελπίδε μας, τα όνειρά μας και τόσων Ευρωπαίων πολιτών που πιστεύουν στο μέλλον. Και στέλνουμε το μήνυμα ότι η ευρωπαϊκή θαγένεια βρίσκεται σε κίνδυνο, ότι μπορεί να σα αφαιρεθεί με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Κι όμως η Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια αποτελεί ένα ξεκάθαρο καθεστώς και πρέπει να προστατεύεται και να προστατευτεί και τώρα σε αυτήν την χωρίς προηγούμενο κατάσταση. Και αν δεν γίνει αυτό τώρα, πότε θα γίνει. Πολύ ευχαριστώ. Πολύ συγκινητική η παρουσίασή σας. Τρίτη βασική οργάνωση Ρότζερ Κασάλη, είστε πρόεδρος των New Europeans, ε, οργανώση για την προστασία των ε, πολιτικών δικαιωμάτων, ε, για την αρχή της μη διάκρισης, για την αλληλεγγύη στην Ευρώπη. Αυτές είναι οι αρχές που υπερασπίζεστε μέσα από την οργάνωσή σας. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε Μπρόκ, αγαπητοί εξέτοιμοι βουλευτές, Ευχαριστώ που μου δίνετε την ε, δυνατότητα να ανταλλάξουμε απόψη αυτό το σημαντικό ζήτημα και όπως και και οι 3 Millions ε, ανησυχούν ε, για τα δικαιώματα των 3 εκατομμυρίων Βρετανών που ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. έτσι και θα πρέπει να μας απασχολούν εκατομμύρια των Βρετανών στο Ηνωμένο Βασίλειο που ανησυχούν γιατί χάνουν το δικαίωμα Ιθαγένειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλουν να διατηρήσουν, να διαφυλάξουν κάποια δικαιώματα. Και επίσης ε, τα δικαιώματα των μεταναστών, των προσφύγων, το δικαίωμα τη ελεύθερη μετακίνησης, ε, το settle status ε, που μπορούν να έχουν το καθεστώς, το ρυθμιμένο καθεστώ. Αυτό δεν σημαίνει δικαίωμα μόνιμη διαμονή. Και η ερώτηση που ακούμε, τι θα συμβεί με τους Βρετανούς που ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το αντίστροφο, εάν, έτσι, εάν, γιατί δεν είναι αναπόφευκτο. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι ε, αναπόφευκτο, ε, μπορεί να πιστεύουμε ότι ε, θα συμβεί, αλλά θέλω να καταγραφεί ότι δεν πιστεύω ότι είναι αναπόφευκτο. Λοιπόν, τα αυτά τα 5 εκατομμύρια, νομίζω ότι είναι λιδία αλήθως για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν θέλουμε να μιλάμε για την Ευρώπη των πολιτών στο μέλλον για ένα ασφαλές χώρο δικαιωμάτων για τους πολίτες, για την προστασία και ε, το σεβασμό των δικαιωμάτων θα είναι λιδία λίθος αυτό που σημαίνει. Ε, λοιπόν, μιλάμε ε, για την περίοδο μέχρι το 2020. Ανησυχούμε τι θα συμβεί με την ενδεχόμενη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Τι θα γίνει με τα δικαιώματα. Αυτό είναι το ερώτημα που μας απασχολεί σήμερα. Και μετά από πέντε χρόνια δεν έχουμε πλησιάσει καθόλου μια μονιμότερη λύση. Και βέβαια ε, ε, τι μου θυμίζει αν τα ξέρω που λέμε άντε φτάσαμε. Όχι δεν φτάσαμε λοιπόν. Ε, διότι ε, και είναι περίεργο αυτό διότι στο Ηνωμένο Βασίλειο ανέκαθεν ναι, και πιστεύω αυτό θα εξακολουθήσει να ισχύει, υπάρχει ευρεία συνένεση εδώ ε, εξω κοινοβουλευτικά ότι ε, θα πρέπει αμελητή να υπάρχει μονομερής εγγύηση για η διαφύλαξη των, και κατοχήρωση των δικαιωμάτων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, όλοι αναγνωρίζουν την ανάγκη να γίνει αυτό. Εντάξει, κάποιοι θέλουν να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν αλλάζει τίποτα και κάποιοι δεν δεν μπόρεσαν να, ε, καν να ψηφίσουν και είναι σε αυτό το λίμπο, αυτή την ανασφάλεια. Ε, και με την ε, πριν από το δημοψήφισμα μία οργάνωση που είναι κατά της μετανάστευσης ε, παρά το όνομά της, λέγεται Migration, είπε ότι θα πρέπει να υπάρχει αυτή η εγγύηση προτού εκείνη κάνει το δημοψήφισμα. Πού είναι αυτή η εγγύηση. Πολλοί το πιστεύουν. Αυτοί που ψήφισαν ότι πρέπει να αποχωρήσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούν ότι άμεσα θα πρέπει να υπάρξουν χέγγια, να διαφυλάτονται τα δικαιώματα. Ε, όλες οι επιτροπές, όλοι, η σύσσωμη αντιπολίτευση, όλοι το ζητάνε και εξακολουθεί αυτή ε, η κατάσταση ανασφάλειας που οξύνεται τόσο πολύ όπως δείχνουμε και με τις μελέτες μας που σας έχουμε δώσει την Επιτροπή ε, που συνιστά αυτό παραβίαση της ε, ε, Σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή δεν έχουν δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης σχεδόν κατοχυρωμένο και αυτό ισχύει για 5 εκατομμύρια Ευρωπαίων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Λοιπόν πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι θα πρέπει να κάνουμε για να σταματήσει αυτό. Αύριο πρέπει να σταματήσει από την Βρετανική κυβέρνηση και με μονομερή δράση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί λοιπόν συμβαίνει αυτό. Τρεις βασική ε, λόγοι, γιατί δεν ακούγεται η φωνή τους. Αυτό το χειριζόμαστε, διότι μετά το δημοψήφισμα ε, οι 3 Millions, in Britain Europe, διάφορες οργανώσεις έχουν ε, συγκροτηθεί και είναι πολύ αποτελεσματικές ε, και τους έχουμε σταθεί μαζί τους, τους υποστηρίζουμε και χαίρομαι πάρα πολύ ε, για την δέσμευση που έχουν αναλάβει, την αναγνώριση της οποίας χαίρουν και δεν, είναι μόνο, δεν είσαστε εσείς, υπάρχουν και άλλες οργανώσεις που υπερασπίζονται τα δικαιώματα, δεν έχουν την ίδια εκπροσώπηση, αλλά χαιρόμαστε γιατί ακούγονται αυτές οι φωνές και γίνεται lobbying για τα δικαιώματα ε, των Ευρωπαίων και ε, ε, ενώνουμε τις δυνάμεις μας και οπότε ακούγονται οι φωνές. αυτού. Ε, το έχουμε καταφέρει. Αλλά πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ανταπροσωπευτικότητα και μεγαλύτερη διασύνδεση με τα θεσμικά όργανα. Ε, έχει, υπάρχει μια διακοινοβουλευτική ομάδα και μια ομάδα φιλίας ονομάζεται στο Βρετανικό Κοινοβούλιο για να ε, υπάρχει λογοδοσία, διαφάνεια, να είναι ανοιχτές αυτές οι ομάδε, ούτω ώστε να συσπηρωθούν όλε αυτές οι νέες οργανώσεις για να υπάρχει πρόσβαση σε όλους. Λοιπόν, αυτά έχουν συμβεί και είναι σημαντικό να συνεχίσουν. Αλλά υπάρχει κι άλλος φραγμός. Η ίδια η Βρετανική κυβέρνηση, διότι ξέρουμε πως η Τερέζα Μπέι θέλει να διαπραγματευτεί και όχι να νομοθετήσει. Πρέπει να σταματήσει λοιπόν να διαπραγματεύεται και να αρχίσει να νομοθετεί. Ε, το, η νομοθεσία για την μετανάστευση θα, ε, ε, θα, φτάσει στο κοινοβούλιο και ήρθε η στιγμή να κάνει το σωστό Βρετανική κυβέρνηση. Αμελητή να δώσει τις μονομερίες, τα μονομερή εχέγγυα για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων ε, των πολιτών τη Ευρωπαϊκή Ένωση του ΕΒ και θα ασκούμε πίεση γι' αυτό. Για κάτι άλλο που ίσω δεν γνωρίζετε ήδη, να σα πω, ε, και κάτι που δεν είναι διαδεδομένο. Η Βρετανική κυβέρνηση δεν ασχολείται με τους ε, Βρετανούς που είναι στην Αλοδαπή, όπως και για τους Ευρωπαίους, πόλους Ευρωπαίους που είναι στο Ενωμένο Βασίλειο και το ξέρουμε διότι για τις ε, κοινοβουλευτικές εκλογές ε, θέλαν να δώσουν σε 17χρονους ε, το δικαίωμα ψήφου για το δημοψήφιο. Τέλος το πήραν πίσω αυτό, τους εμποδίσαμε. Ε, λοιπόν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι από την πλευρά των δικαίων, αλλά ε, μην ξεχνάμε τι γίνεται με τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα. Αλλά ε, λένε κάποιοι, α, δεν είναι δικό μου το πρόβλημα, εκείνοι θέλουν να φύγουν. Ε, ζητάμε συγγνώμη που ε, έχουν μπλεχτεί σε αυτό το πράγμα, σε αυτήν την ανακατοσούρα, γιατί τι έχουν κερδίσει τώρα οι Βρετανοί υπήκοοι μέχρι στιγμή τίποτα. Ε, και όπω είπε ο κ. Σταρ, δεν είναι το θέμα ε, ποιον θα κατηγορήσουμε και ποιον θα κληροδεικτούμε. το θέμα είναι τι θα γίνει, το θέμα ευθύνη, γιατί μπορεί να μην είστε υπεύθυνοι για αυτό που συνέβη, αλλά είστε υπεύθυνοι για αυτό που θα γίνει στο μέλλον. Αυτά που κάνει τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κατοχυρώσουν ή όχι τα δικαιώματα μελλοντικά. Λοιπόν, και μα λέει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί έχουμε επαφέ μαζί τη, α ζητούμε συγγνώμη, δεν έχουμε νομική βάση και δεν έχουμε διαπραγματευτική εντολή για να μπορέσουμε να χορηγήσουμε δικαίωμα ελεύθερη μετακίνηση στου πολίτε του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σα παρα... Σας ζητούμε λοιπόν να επανέλθετε στο Συμβούλιο να διαζητήσετε την τροποποίηση τη εντολή σα. Το, δεν είναι ο δικό σας ρόλος να ορθώνετε νέα εμπόδια ε, και προσκόμματα ε, στον δρόμο των πολιτών, αλλά να βρίσκετε τρόπο να υπερπηδείτε τα εμπόδια, να δείξετε ε, ποιον ηγετικό ρόλο μπορείτε να έχετε, γιατί η μεγαλύτερη οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξαναλέω, είναι λιδία λίθος για την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό που συμβαίνει. Άλλο τώρα που τίθεται ως θέμα και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πώς ε, θα ξαναδώσουμε το δικαίωμα ελεύθερη μετακίνηση στους Βρετανούς. Ε, το Κοινοβούλιο έχει αναλάβει δέσμευση να ε, δώσει ας το ψήφισμα έτσι του Δεκεμβρίου να δώσει, επιστρέψει αυτό το δικαίωμα ελεύθερη μετακίνηση. Πώς θα γίνει αυτό όμως στην πράξη. Ε, πώς θα μεριμνήσετε ώστε να το έχουν οι Βρετανοί. Προς το παρόν ε, δεν έχουμε ακούσει κανένα στοιχείο απάντησης. Δεν έχω χρόνο τώρα για να σας κάνω όλη αυτή την παρουσίαση PowerPoint, αλλά ούτως ή άλλως ε, θα επισυναυθεί στα πρακτικά, πειράζει. Ε, έχουμε, έχει, έχει κερδίσει και βραβείο αυτή η αλλω θα επισυναυθει στα πρακτικα δεν πειραζει εχουμε εχει Από τους Financial Times ε, υπήρχε ε, ολόκληρο άρθρο για την έκδοση πράσινης κάρτας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πακέτο δηλαδή ε, δικαιωμάτων ηθαγένειας ε, που πάνε πακέτο με το διαβατήριο. Δηλαδή μετά την αποχώρηση της Βρετανία θα μπορούν να διαμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιο αποτέλεσμα έχει αυτό. Η πολίτες, πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο με το που διευκρινιστεί το καθεστώς διαμονής ε, θα τύχουν τις ίδιες μεταχειρήσεις σαν να ήταν ακόμη κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο από πλευράς ε, ηθαγένειας. Όλο το πακέτο έτσι, δικαίωμα στη ψήφου, στις τοπικές εκλογές, δικαίωμα μη διακριτικής μεταχείρισης κτλ. Και αυτό για τους υπηκόρους τρίτων χωρών, εν χρόνο. Λοιπόν, κλείνω και ζητώ από εσά. Η Ντανίτα Χίμνερ μα ζήτησε να συντάξουμε μια σύντομη μελέτη για την ΑΦΚΟ. Ε, θα είναι ε, αυτός ο σκέντος που μόλι ακούσατε. Διότι Ωραία. Ε, έχει αναλάβει τη δέσμευση μετά την αποχώρηση της Βρετανία να έχουν τα δικαιώματα οι πολίτες. Όμως, εντάξει, πρέπει να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση με συγκεκριμένες προτάσεις από εσάς πώς θα γίνει αυτό και ελπίζουμε αυτή την πρόταση που σα κάνουμε να την εξετάσετε μεταξύ άλλων ε, που θα προκύψουν στο άμεσο μέλλον. Σας ευχαριστούμε. Okay, so the final part of this panel before us. Ε, ο τελευταίος ομιλητής ε, πριν να ζητήσω από τους ευρωβουλευτές να κάνουν ερωτήσεις βλέπω και κάποιον που φεύγει αν θέλετε να μιλήσετε τώρα λοιπόν για 10 λεπτά και μόλις τελειώσουμε αυτό το κομμάτι θα ακούσουμε και ερωτήσεις ε, προς ε, τους οργανισμούς από τους ευρωβουλευτές. Θα ζητήσω λοιπόν από την καθηγήτρια Λενό, Παβέντα από το νομική σχολή του Ντερχάμ να μας κάνει μια παρουσίαση της επικαιροποίησης της μελέτης που ζήτησε η Επιτροπή Αναφορών και που αφορά τις επιπτώσεις του Brexit σε σχέση με το δικαίωμα αναφορά. Παρακαλώ, περιοριστείτε στα 10 λεπτά, αλλιώ θα έχουν φύγει όλοι οι ευρωβουλευτέ. Οπότε, εναπόκειται σε εσά, μην περάσετε τα 10 παρακαλώ, γιατί ούτω ή άλλω η παρουσίαση σα θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα. Θέλω ε, κάποιοι ευρωβουλευτέ και αυτοί που δεν είναι από το Ηνωμένο Βασίλειο, ιδιαίτερα που αφιέρωσαν το χρόνο του εδώ, να σα κάνουν ερωτήσει. Και ζητώ συγγνώμη για όλα τα προβλήματα επικοινωνία που υπήρξαν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε εδώ. Θα είμαι πολύ σύντομη. Ευχαριστώ ο Πρόεδρος και τον κύριο Μπρόκ για όλες τις προσπάθειες που έκανε. Η κυρία Σπαβέντα, Όταν έγραψα πριν από έξι μήνες τη μελέτη μου, εντόπισα κάποιους κινδύνους που κατά την απόψή μου ήταν ρεαλιστικοί για Ευρωπαίους πολίτες του ΕΒ και για πολίτες του ΕΒ στην Ευρώπη αντίστοιχα. Οι περισσότεροι από αυτούς τους κινδύνους δεν έχουν εξεταστεί ούτε αναλύονται στην κοινή έκθεση. Ελπίζω να τους εξετάσουμε αργότερα. Το βασικότερο πρόβλημα, πιστεύω εγώ, είναι το ότι βασιζόμαστε υπερβολικά στην ιδέα της νόμιμης κατοικίας, διότι σκοπός ε, της ενωσιακής ηθαγένειας είναι να δημιουργηθεί ένα χώρο όπου μπορεί να μετακινηθεί, να κυκλοφορήσει ελεύθερα ο πολίτης και επειδή αφαιρούμε αυτήν ε, την, ε, την κατάσταση, μπορεί ο πολίτης να μην νομίζει ότι πρέπει να κάνει κάτι. Να σα δώσω ένα παράδειγμα. Ένας εργαζόμενος που θέλει να παραμείνει εργαζόμενο κάτι σημαντικό για τα δικαιώματά του, θα πρέπει να εγγραφεί στο Γραφείο ενεργεια. Οι περισσότεροι πολίτες, ειδικότερα οι νέοι, όταν η ζωή τους ε, είναι έτσι αβέβαιη, άλλες φορές δουλεύουν, άλλες όχι, δεν θα το γνωρίζουν αυτό. Δεν θα καλύπτονται δηλαδή από τη συμφωνία ως έχει, παρότι θα έχουν ε, καλόβουλα ε, μετακομίσει. Δεν θα έχουν κάνει κάτι κακό, απλά δεν γνωρίζουν πώς γίνεται. Το ίδιο θα γίνει και με τις ασφάλειες κτλ. Το Ηνωμένο Βασίλειο, όπως λέει σήμερα, θα άρει την απέτηση για υποχρεωτική ε, ασφάλιση υγείας, αλλά στην έκθεση αναφέρεται κάτι σχετικό μόνο για τους ηλικιωμένους που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Καρτά Υγείας. Δεν καλύπτονται όλοι οι γυναίκες. Οι γυναίκες δεν έχουν συμπεριληφθεί σε αυτή τη συμφωνία. Γιατί δεν υπάρχει εκτίμηση των επιπτώσεων αυτής της συμφωνίας βάσει του φύλου. Να δώσω άλλο ένα παράδειγμα. Αν είμαι μετανάστρια, εργαζομένη στο Ηνωμένο Βασίλειο και έχω παιδί, οικονομικά μπορεί να μου είναι αδύνατο να πάω να δουλέψω λόγω του κόστους ε, του παιδικού σταθμού ή μπορεί να αποφασίσω να μένω σπίτι. Και σε αυτή την περίπτωση δεν με προστατεύει πια η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ούτε αυτή η συμφωνία. Μιλάμε τώρα για τι γυναίκε που φροντίζουν τα παιδιά του, Δεν αποκλείω και το ενδεχόμενο ένα άντρα να φροντίζει το παιδί του. Μιλάμε όμω κυρίω για γυναίκε, αναπήρου και ηλικιωμένου. Αυτοί αποκλείονται. Τα παιδιά, τα παιδιά δεν αναφέρονται σε αυτή τη συμφωνία τα δικαιώματα του παιδιού δεν αναφέρονται, ο χάρτης δεν θα εφαρμόζεται σε αυτή τη συμφωνία και πού αφήνει αυτό τις πιο ευάλωτες κατηγορίες ε, της κοινωνίας, παιδιά τα οποία δεν έχουν λάβει καμία απόφαση. Δεν έχουν κανένα δικαίωμα να συνεχίσουν να βρίσκονται στην εκπαίδευση όπως ε, υπάρχει αυτή τη στιγμή υπό την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Δεν θα υπάρχει τέτοιο ε, δικαίωμα. Δεν αναφέρεται κάτι τέτοιο στην κοινή έκθεση. Οι ε, σύζυγοι ε, από τρίτες χώρες θα προστατεύονται αν είναι ήδη νομίμοι κάτοικοι, αλλά υπό το ευρωπαϊκό δίκαιο ο νόμιμος κάτοικος, ο μόνιμος κάτοικος δεν αποτελεί προϋπόθεση για τέτοια προστασία. Αυτό είναι απόκληση από το κεκτημένο που δεν αναγνωρίζεται καν στην έκθεση και θα παρότρινα το Κοινοβούλιο να απαιτήσει οποιαδήποτε απόκληση από το κεκτημένο να ορίζεται και να εξηγείται καθαρά. Διότι είναι τόσο περίπλοκη η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία που πολλοί κόσμος μπορεί να μην γνωρίζει ότι υπάρχει απόκληση από το κεκτημένο. Με ανησυχούν ιδιαίτερα τα δικαιώματα των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου που θα επιστρέφουν στο Ηνωμένο Βασίλειο λόγω των πολύ αυστηρών μεταναστευτικών κανόνων ε, για τα μέλη των οικογενειών τους. Δεν έχουν αντιμετωπιστεί αυτά τα ζητήματα, αλλά δύο λεπτά μου. Επίση ανησυχώ ιδιαίτερα όσον αφορά την υλοποίηση αυτής της συμφωνίας. Γιατί, διότι όλη η συμφωνία βασίζεται στην οδηγία 38-2004 και όχι στην άσκηση των δικαιωμάτων της συνθήκης. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι αν δεν πληρείται το γράμμα του νόμου είναι έξω. Δεν υπάρχει αναλογικότητα, δεν υπάρχει αξιολόγηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ένα παραδείγμα από το Ηνωμένο Βασίλειο να σας δώσω επειδή αυτό το σύστημα γνωρίζω καλύτερα. Το Ηνωμένο Βασίλειο από το 2017 και μετά έχει εισηγαγεί μια νέα ιδέα κατάχρηση των ευρωπαϊκών δικαιωμάτων. Κάτι άγνωστο στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Η οδηγια 2438 μιλά για κατάχρηση ευρωπαϊκών δικαιωμάτων. Εάν καταχράται κάποιο τέτοιων δικαιωμάτων που του παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, και το παράδειγμα στην οδηγία δημιουργεί πρόβλημα, διότι ουσιαστικά λέει ότι αν μπει και βγει κανεί ε, διαρκώ, αν μπαίνει και βγαίνει διαρκώ στο όνομα Βασίλειο, θα αποτελεί αυτό κατάχρηση των δικαιωμάτων. Μπορεί κανεί ε, έτσι να εκδιωχθεί για 12 μήνε από το όνομα Βασίλειο, να μην μπορεί να ξαναμπεί. Σα ε, προκαλώ να βρείτε ένα νομικό στην Ευρώπη που θεωρεί ότι αυτό είναι συμβατό με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Αυτό σα δίνει μία ένδειξη του ότι ο τρόπο με τον οποίο το Ηνωμένο Βασίλειο προσεγγίζει το Brexit ε, δημιουργεί πρόβλημα όσον αφορά την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Τώρα η κοινή συμφωνία ε, διαθέτει μια ρήτρα που λέει ότι σε περίπτωση κατάχρησης των δικαιωμάτων του ένας πολίτης χάνει το δικαίωμα να παραμείνει στην χώρα υποδοχής ε, αναμένοντας ε, το αποτέλεσμα της προσφυγής. Αν τα βάλετε αυτά μαζί, αντιλαμβάνεστε σε πόσο τοξική κατάσταση βρισκόμαστε, σε τι κίνδυνο βρισκόμαστε, γιατί το Ηνωμένο μπορεί να ε, αποφασίσει να ερμηνεύει πολύ ε, γενικόλογα όλο αυτό το ζήτημα της καταχρήσης των δικαιωμάτων και να αναγκάσει ανθρώπους να φύγουν. Επίσης με ανησυχεί το εχθρικό αυτό περιβάλλον που νιώθουμε στο Ηνωμένο και το γεγονό ότι θα εφαρμοστεί αυτό εις βάρος των Ευρωπαίων πολιτών. Δεν θέλω απλά να επικρίνω πράγματα. Δεν είναι μόνο αυτό που θέλω να κάνω. Απλά είναι νομικά προβλήματα αυτά τα οποία είναι δυσεπίλητα. Πρέπει να γίνει μια προσπάθεια να εξετάσουμε τα σημερινά ε, καθεστώτα μετανάστευση σε όλα τα κρατημελικές στο Ηνωμένο Βασίλειο και να αξιολογήσουμε τι θα γίνει όταν αυτά θα εφαρμοστούν στους πολίτες του Brexit, έτσι αναφέρομαι σε αυτούς, κατά πόσο θα είναι συμβατά με το πνεύμα και το γράμμα της συμφωνίας. Και το πρόβλημα δεν είναι μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, διότι γνωρίζουμε για παράδειγμα ότι ε, εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης δεν θα έχουν το δικαίωμα ε, ελεύθερης μετακίνησης νομίζω στο τουλάχιστον τα μισά κράτη-μέλη. Λοιπόν, πριν τελειώσω να πω, ναι, ε, είναι μια καλή αφετηρία, αλλά ανησυχώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ε, τελικός κανονισμός αυτό. Αυτή η συμφωνία είναι εντάξει για έναν ε, εργαζόμενο πλούσιο απασχόλησης που ανέκαθεν δούλευε full, αλλά δεν είναι έτσι οι περισσότεροι άνθρωποι. Πολλές συμβάσεις υπάρχουν που ορίζουν ώρες εργασίας και όχι μόνο με απασχόληση. Οπότε θα πρέπει να προσέξουμε, να προστατεύσουμε όλους ε, και όχι μόνο όσους ε, ε, ανήκουν σε μια συγκεκριμένη κατηγορία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Σπαβέντα. Όλη σας η παρουσίαση με τα slide θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Μπορούμε τώρα να ακούσουμε κάποιες ερωτήσεις και να δοθούν κάποιες απαντήσεις διότι βλέπω ότι έχει αρχίσει να φεύγει ο κόσμος και θέλω να έχουμε κάποια άλλη επίδραση. Είχαμε πει ότι οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις θα γίνουν στο τέλος και των δύο πάνελ, αλλά ε, μέχρι τότε θα έχουν φύγει όλα τα μέλη. Βέβαια θα έχουν έρθει και κάποια άλλη. Λοιπόν, ας ε, ακούσουμε λοιπόν κάποιες αντιδράσεις από τα μέλη και να ζητήσουμε από το πάνελ, από τους ομιλητές που μόλις ακούσαμε, να απαντήσουν. Και ο κ. Γκουαλτιέρη θέλει να αντιδράσει σε κάποια από τα πράγματα που ακούσαμε. Πρώτα απ' όλα, κυρία Χιμένες Μπεθερέλ. Ένα-δύο λεπτά παρακαλώ καθένας, έτσι όχι παραπάνω. Μετά ο Ρομπέρτο. Και μετά η Τζούθι Κάρτον Ντάρλινγκ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Από αυτά που ακούω, είχα κάποια ιδέα για τις διαπραγματεύσεις και έχω ακούσει διάφορα πράγματα και μια προοπτική έτσι πιο μακρινή. Δεν ξέρω αν μου έχουν πει την αλήθεια μέχρι τώρα, πάντως από αυτά που άκουσα εγώ ακούσει λέξεις όπως είναι ανησυχία, προδοσία, φόβος, ε, θλίψη, αβεβαιότητα. Εμείς που εκπροσωπούμε τους Ευρωπαίους πολίτες πρέπει λοιπόν να τους προσφέρουμε ακριβώς το αντίθετο από αυτό. Εμπιστοσύνη, ηρεμία, βεβαιότητα και αν όχι χαρά, τουλάχιστον να μπορούν να ζουν και να δουλεύουν με ηρεμία και ειρήνη. Τρία εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες είπατε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και Βρετανοί σε διάφορες χώρες όπως τη δικιά μου. 270.000 φαίνεται στην Ισπανία, αν και στην πραγματικότητα είναι πάνω από 800.000. Είμαι από την Ανδαλουσία εγώ και σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε λέει ότι είναι 80.000 μόνο στη Μάλαγα εγκαταστημένοι Βρετανοί, έτσι. Αν και στην πραγματικότητα είναι πάνω από 100.000. Άσε πια στην Αλικάντε, στη Μούρθια κλπ. που είναι πάρα πολύ. Ήμουνα σε μια συνάντηση μαζί του και τους είπαμε ότι για δύο χρόνια είναι κειμένα τα δικαιώματά του, Αν από αυτά που λέτε εσεί φαίνεται ότι δεν είναι απόλυτο αυτό, τουλάχιστον για υγεία, περίθαλψη, εκπαίδευση κλπ. Τι με ρωτούσανε. Με ρωτούσαν κάτι πολύ σημαντικό για αυτούς. Το δικαίωμα ψήφου των πολιτών αυτών στους Δήμους. Σε ένα μισή χρόνο, ένα σχεδόν, θα έχουμε ε, εκλογέ δημοτικές εκεί. Οπότε έχετε να μας πείτε τίποτα εσείς για το δικαίωμα αυτό ψήφου των Βρετανών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Θα ακούσουμε τρεις-τέσσερις ερωτήσεις και μετά να απαντήσετε εσείς, έτσι, το πάνελ. Ρομπέρτο τώρα, σύντομα παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ναι, θέλω να αντιδράσω σε κάποια από αυτά που ακούσαμε. Φυσικά, τα γνωρίζω, είναι αναπόφευκτο να υπάρχει ανησυχία Όταν έχουμε να κάνουμε με τέτοια πράγματα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πίσω από κάθε πράξη, διάταξη, διατύπωση υπάρχουν άνθρωποι. Γι' αυτά που είπα Σπαβέντα, ναι υπάρχουν προβλήματα πολύ δύσκολα για να βρεθεί λύση. Και γι' αυτό είναι πολύ περίπλοκο να προστατεύσουμε τα δικαιώματα σε ένα διαφορετικό συνταγματικό πλαίσιο. Τώρα, από αυτά που υπόθηκαν, στη θεωρία τουλάχιστον πολλά από αυτά καλύπτονται. Να δούμε βέβαια στην πράξη πώς θα εφαρμοστούν. Και υπάρχουν και άλλα που δεν καλύπτονται και θα έπρεπε να καλυφθούν. Ε, για το λάθος που λέτε. Κάνει κάποιος κάποιο λάθος και πρέπει να φύγει. Λέτε ότι πρέπει να δούμε πώς το 17ΒΓ συντάσσεται, γιατί η διατύπωση εδώ είναι ότι όταν κάνετε κάποιο λάθος ε, πρέπει να έχετε τη δυνατότητα να το διορθώσετε και όχι να ε, σας διώξουν. Αυτό το λέει το Ηνωμένο Βασίλειο. Οπότε αυτή είναι μια μάχη που πρέπει να δώσουμε γιατί έχουμε εδώ μια βάση να βασιστούμε πάνω. Τώρα αυτό πρέπει να το διασταυρώσουμε και μάλλα. Λέτε ότι οι αποφάσεις δεν θα εφαρμοστούν όχι σύμφωνα με την παράγραφο 18 που λέει εφόσον εκκρεμεί μια τελική απόφαση και είναι σημαντικό. Τότε ισχύουν τα δικαιώματα. Δηλαδή δεν μπορεί να σας διώξει κανείς αν δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Παραμένετε, το λέει εδώ. Πρέπει να εφαρμοστεί φυσικά. Δηλαδή αν υπάρχει λάθος έχετε τη δυνατότητα να το διορθώσετε. Αν σας πούνε όχι δεν γίνεται και εσείς κάνετε προσφυγέφυση κτλ. Έχετε δικαίωμα να παραμείνετε μέχρι να τελεσιδικήσει υπόθεση. Και επίσης έχετε δύο χρόνια για να κάνετε την αίτηση. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί κανείς να σας διώξει με τίποτα, παρά μόνο αν περάσουν τα δύο χρόνια. Έχετε κάνει την αίτησή σας, απορριφθεί, έχετε κάνει την προσφυγή σας και απορριφθεί και αυτή. Μόνο τότε, έτσι λέει εδώ, μέχρι τότε δεν μπορεί να σας διώξει κανείς. Συμφωνώ μαζί σας, πρόκειται για δύο γραμμές το κείμενο. Πρέπει να δούμε πώς θα τεθεί σε εφαρμογή αυτό που λέει εδώ. Τώρα έλεγχο τη εγκληματικότητα, ναι, δεν είναι όπως το θέλαμε. Είναι διατυπωμένο έτσι, λέει, αν διαβάσετε προσεκτικά, ότι όπως και να έχει το πράγμα, εφαρμόζονται τα άρθρα 17 και 18. Ακόμα δηλαδή και αν υπάρξει έλεγχος για εγκληματικότητα δεν μπορούν να σας διώξουν γιατί αν εσείς προσφύγετε πρέπει να περιμένουν να τελεσυδικήσει η υπόθεσή σας. Αλλά πράγματι είναι εκεί που δεν ήμασταν και τόσο ευτυχισμένοι. Πρέπει να δούμε στην εφαρμογή πώς θα προχωρήσουν αυτά τα θέματα. Εφαρμογή. Το λέει η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλάει για εφαρμογή. Υπάρχει αυτή η λέξη, όρος. Τι δώσαμε τη μάχη. Θέλαμε να υπάρχουν δηλώσεις, δήλωση, δήλωση, δήλωση, αλλά Τέλος πάντων, το δέχτηκε η Επιτροπή γιατί υπάρχει στο ευρωπαϊκό δίκαιο ο όρος εφαρμογή. Θα έπρεπε όμως ε, να πρόκειται για δήλωση. Το νόημα να είναι δηλωτικού χαρακτήρα. Και θα έπρεπε αυτόματα να μετατρέπεται σε δηλωτικό Θέλουμε ενία εφαρμογή. πανέ, το θέμα της επανένωσης οικογενειών θα εξεταστεί μαζί. Τι σημαίνει μαζί, σημαίνει ένα ενιαίο έγγραφο. Δεν μπορεί να πάρει κανείς διαφορετική απάντηση ε, στη μία ή την άλλη περίπτωση επανένωσης οικογενειών. Και τέλος, συμφωνώ απόλυτα το θέμα των επιλογών. μόνο για τα μελλοντικά μέλη της οικογένειας γι' αυτό. Και αυτό είναι που θέλουμε εμείς να πολεμήσουμε. Γιατί το μόνο επιχείρημα που χρησιμοποιούν κατά των μελλοντικών μελών είναι ότι λένε «Μα πρόκειται για μελλοντική επιλογή». Όχι, εγώ λέω ότι εφόσον ε, έχω το δικαίωμα μπορεί να επιλέξω στο μέλλον να έχω μια επιλογή. Δεν πρέπει να βασίζεται στις ε, επιλογές, έχετε απόλυτα δίκιο σε αυτό που είπατε πώς πάμε από τα δικαιώματα στην επιλογή ζωής, ότι δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Έχετε δίκιο. Είναι ένα κενό, σύμφωνο... και γι' αυτό ακριβώς παραμένει ανοιχτό αυτό το θέμα και θα φροντίσουμε να καλύψουμε και τα μελλοντικά μέλη, εκτός αν δεν το θέλετε βέβαια. Δεν μπορούμε να βάλουμε ότι υπάρχει μια επιλογή που έχει ημερομηνία λήξη, το δικαίωμα είναι δικαίωμα, λέει και παύλα. Παρακαλώ, κυρία Κάρτον Ντάρλινγκ. Ευχαριστώ, θα είμαι σύντομη. Συμμετέχω στην Επιτροπή Αναφορών. Και γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να πούμε πως τα τελευταία χρόνια ο αριθμός ε, αναφορών από το Ηνωμένο Βασίλειο έχει διπλασιαστεί. Και η Επιτροπή Αναφορών έχει αποτελέσει άνισμα το μέσο για τους ε, Βρετανούς για να καταλάβουν καλύτερα τα πράγματα που αφορούν τη ζωή τους. Μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι καλή την πίστη ε, θέλησαν να χρησιμοποιήσουν τα δικαιώματα που τους προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση και μετακινήθηκαν προς τη μία την άλλη κατεύθυνση. Και τώρα τιμωρούνται από το Brexit. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να επανέλθω σε αυτό που είπε η Jane Golding. η δουλειά που κάνουμε εμείς εδώ ε, δεν πρέπει να ξεχνάμε τη συνεργασία. Και είναι πολύ σημαντική αυτή που γίνεται και από τις οργανώσεις 3 ε, Million ε, και την άλλη της κυρίας Golding. Χαίρομαι που η Ισπανίδα συνάδελφος επίσης έθεσε το θέμα των πολιτικών δικαιωμάτων που απουσιάζει πλήρως από το πρώτο στάδιο και δεν πρόκειται μόνο για το δικαίωμα ψήφου που πρέπει να μπορούν και να είναι υποψήφοι οι Βρετανοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ευρωπαίοι πολίτες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχουμε και τις τοπικές εκλογές Κλοντ που είναι στο Λονδίνο το Μάιο, οπότε υπάρχει νομικό ζήτημα εδώ θα μπορούν να είναι υποψήφοι ε, κάποιοι μη Βρετανοί ε, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ζουν ε, στο Λονδίνο και αν ναι θα μπορέσουν να φέρουν σε πέρα στη θητεία τους. Πρέπει λοιπόν πρώτα απ' όλα να εντοπίσουμε πού βρίσκονται αυτοί και έτσι θα ήταν καλό οι οργανώσεις να ασχοληθούν και με αυτό. Έπειτα, το θέμα της διάστασης του φύλου. Και αυτή είναι πολύ σημαντική. Έλα να αναρωτιέμαι, θα μπορούσαμε να βρούμε τι ακριβώς διακυδεύεται εδώ για αυτό το θέμα. Γιατί στον Ηνωμένο Βασίλειο ακούμε ας πούμε για μητέρα που παντρεύτηκε κάποιον άλλον, ήρθε και αυτό στο Ηνωμένο και διαπίστωσαν ότι τελικά είναι υποχρεωμένες να μετακομίσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση εκτός Ηνωμένου Βασιλείου και η νομική τους κατάσταση είναι πολύ μπερδεμένη. Μα για μένα η Ευρώπη δεν βασίζεται μόνο στην αλληλεγγύη, αλλά και στην ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Αναφέρεται στη συνθήκη της Ρώμης. Οπότε μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και αυτό. Τέλος. Ένα μικρό σχόλιο που έκανες, Τζέιν, αλλά που και αυτό είναι ζωτικής σημασία. Οι φοιτητέ, τι θα γίνει με αυτού. Δεν υπάρχει σαφήνεια για τους φοιτητέ. Και τα στοιχεία των ιατρικών ε, υπηρεσιών λένε ότι λίγοι φοιτητέ πάνε και θα έχουμε πρόβλημα με το εθνικό μας σύστημα υγείας. Γιατί δεν θα έχουμε γιατρούς. Θα πρέπει να το προσέξουμε πολύ περισσότερο κατά τη γνώμη μου. Ήθελα να το επαναλάβω αυτό γιατί το έπεσε έτσι κάπως στα γρήγορα. Να ξέρετε ότι εμείς θα συνεχίσουμε να πιέσουμε ώστε η δικιά σας η φωνή να εισακουστεί σε αυτή τη διαδικασία και η ανθρώπινη μορφή του Brexit να παραμείνει ζωντανή. Τέλος, να ξέρετε ότι ντρέπομαι για τη δράση της κυβέρνησής μου στον Ηνωμένο σήμερα. Ο κόσμος βρίσκεται ήδη σε πολύ δύσκολη κατάσταση, νιώθει ευάλωτος και αν του προσθέσουμε και άλλη αβεβαιότητα, που, σε ανθρώπους που τελικά δεν μπορούν να πειράσουν καθόλου αυτή τη διαδικασία, είναι τροπή και δεν θα ήθελα να με συνδυάσει κανείς με τις δράσεις αυτές της κυβέρνησής μου. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ, θα πω κάτι βαρετό και πολύ κοινότυπο σε σχέση με αυτά που ακούμε. Η Μαρτίνα Κιτζίν. Θέλετε να είσαστε πρώτες που θα κάνετε ερωτήσεις στο επόμενο πάνελ. Εντάξει. Θα με βοηθήσετε. Βλέπετε κάνουμε διαπραγματεύσεις και εμείς μέσα στο κοινοβούλιο. Λοιπόν, ευχαριστούμε Μαρτίνα και Τζίνη. Ξέρω ότι θα κάνετε καλές ερωτήσεις. Λοιπόν, σύντομες ε, αντιδράσεις, αν θέλετε να αντιδράσετε σε αυτά που ακούσατε. Σε αυτά που ακούσατε και από εμά και από τους άλλους. Δεν είναι υποχρεωτικό, αν θέλετε, να αντιδράσετε, να απαντήσετε. Ευχαριστώ. Στη παράγραφο 17βγ που λέει ότι αν έχουμε κάνει λάθος μπορούμε να το διορθώσουμε. Ναι, αλλά αν δεν έχουμε πρόσβαση στα στοιχεία και τα διαθέτει το Υπουργείο Εσωτερικών, πώς θα κάνουμε αυτή τη διόρθωση. Αυτό είναι ένα σχόλιο. Για την παράγραφο 18. Ναι. Έχουμε δύο χρόνια να κάνουμε προσφυγή αλλά πού θα καταλήξουμε σε κάποιο κέντρο κράτηση. Και ξέρουμε τι κατάσταση επικρατεί εκεί. Άνθρωποι αυτοκτονούν εκεί, πεθαίνουν, ε, τους κακομεταχειρίζονται κλπ. κλπ. Όσον αφορά την ε, εφαρμογή κατά δήλωση, πρέπει να είναι δηλωτικού χαρακτήρα η εφαρμογή. η γραφειοκρατία και στη Γαλλία για παράδειγμα απόλυτα, αλλά εκεί δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Ας γίνει λοιπόν και για μας για το νέο καθεστώς που θα έχουμε. Να μην βάλουμε εφαρμογή, γιατί εφαρμογή σημαίνει όρη. Και για τους φοιτητέ ε, και για τη διάσταση του φίλου συμφωνώ. Για τους φοιτητέ πιο συγκεκριμένα, δύο είναι τα ζητήματα. Ξέρουμε και το λέει σαφώς ότι αν αρχίσουμε το δίπλωμα πριν το Brexit έχουμε τα ίδια δικαιώματα. Αν μετά το Brexit δεν έχουμε ιδέα. Μπορεί να είμαστε σαν τρίτη χώρα. χώρας. Αν θέλουμε τώρα μετά το Brexit να σπουδάσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είπα και νωρίτερα, θα θεωρηθούμε υπήκοοι τρίτης χώρας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πληρώνουμε. Δεν έχει να κάνει με την εθνικότητα ή τη χώρα διαμονής. Θα πρέπει να πληρώσω όπως πληρώνουν αυτοί που είναι από την Ασία, για παράδειγμα, φοιτητές. Σύντομα, παρακαλώ. Ναι, ναι, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομα και εγώ για τα πολιτικά δικαιώματα. Εμείς καταλαβαίνουμε ότι δεν θα καλυφθεί από την συμφωνία. Και το Ηνωμένο Βασίλειο σε διμερή βάση θα διαπραγματευτεί βάση εθνικού δικαίου. Για τα πολιτικά δικαιώματα, ναι, πολλοί έχουν εκφράσει ανησυχία. Δημοτική Σύμβουλη κυρίως στην Ισπανία και μας ρώτησαν για τη μεταβατική περίοδο, πώς επηρεάζει τα δικαιώματα των Δημοτικών Συμβούλων, αν θα μπορέσουν να παραμείνουν στη μεταβατική περίοδο Δημοτική Συμβουλή όχι. Για τα άλλα που είπε ο κύριος Γκουαλτιέρη, δεν θα πω πολλά γιατί έχουν να κάνουν με αυτά που ακούσαμε από το 3 Million. Προφανώς όμως όλα αυτά τα θέματα θέλουμε να διατυπωθούν πολύ συγκεκριμένα και να εφαρμοστούν καλά οι κανόνες πρέπει να είναι πιο ξεκάθαροι. Αν υπάρξει διαφωνία, αν υπάρχει μια διαδικασία επίλυσης διαφορών και βέβαια κυρώσεις. Χαίρομαι που λέτε ότι πρέπει να προστατεύονται τα δικαιώματά μας και όχι οι επιλογές ζωής μας. Και η ελεύθερη διακίνηση είναι ένα δικαίωμα. Συμφωνώ με το όσο υπόθηκαν για την ισότητα των φύλων. Και τέλος, για τους φοιτητές. Έχουμε το ίδιο θέμα με παιδιά Βρετανών που ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που πληρώνουν δίδακτρα. Και υπάρχει ζήτημα και με την αναγνώριση των διπλωμάτων που μπορεί να έχουν αρχίσει πριν το Brexit, αλλά να τελειώσουν μετά. Αν φύγουν από τη χώρα διαμονή τους θα χάσουν τα δικαιώματα που έχουν συλλέξει στη χώρα διαμονή τους. Αν λείψουν πολλά χρόνια. Παρακαλώ. Σύντομο. Ναι. Για το θέμα της μεταφοράς. Αν υπήρξε κάποια κατάχρηση, θα πρέπει να περιμένει κανείς να δική υπόθεση. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό να υπάρχει στη συμφωνία. Δεδομένε της ερμηνεία που δίνει το Ηνωμένο Βασίλειο που δεν είναι στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, είναι επικίνδυνα τα πράγματα εδώ. Για τα πολιτικά δικαιώματα είναι θέμα αρμοδιότητας. Τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, μέλη πρέπει να δώσουν τα πολιτικά αυτά δικαιώματα. Αλλά υπάρχει και το ζήτημα κατά πόσο έτσι υπάρχει διάκριση με άλλους. Γιατί αν είναι τρίτη χώρα, το Ηνωμένο Βασίλειο, τότε τίθεται το ζήτημα πώς ε, μεταχειρίζεστε ανθρώπους που μπορεί να βρίσκονται σε αντίστοιχη κατάσταση. Για τους φοιτητές θέλω να επαναλάβω ότι για τα πανεπιστήμια αυτό είναι ένα πρόβλημα και είναι και οικονομικό ζήτημα. Είμαστε ένας πολύ σημαντικός κλάδος της οικονομίας του Ηνωμένου Βασίλειου τα πανεπιστήμια. Τέλος, παρακαλώ. Βάλτε κάτι και για την διπλή υπηκότητα. Το δικαστήριο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο διευκρίνησε ότι αυτοί που έχουν και την υπηκότητα της χώρας στην οποία διαμένουν προστατεύονται από το ευρωπαϊκό δίκαιο. Να διευκρινιστεί. Γιατί πολλοί βιάζονται να πάρουν μια άλλη υπηκότητα για να τύχουν αυτή τη προστασία. Αλλά πρέπει να μπει στην συμφωνία αυτό. Ευχαριστούμε. Να μείνει η πόρτα ανοιχτή, Ρομπέρτο, για όποιον θέλει να μείνει στον Ηνωμένο Βασίλειο για την προστασία των δικαιωμάτων. Να υπάρχουν στο και μονομερείς εγγύσει και πώς όλα αυτά θα γίνουν νομοθεσία. Στη δουλειά μας, στη Βουλή των Κοινοτήτων, το έχουμε υπόψη μας. Το Υπουργείο Εσωτερικών διαβουλεύεται Υπάρχει μια ευκαιρία, Ρομπέρτο, νομίζω ότι δεν είναι ακριβώ έτσι όπως νομίζεις. Πρέπει να δούμε πώς θα καλυφθούν τα κενά. Θέλουμε κι εμείς, δηλαδή στον εσωτερικό να υπάρχει κάτι πλήρες και να γίνει τώρα. Να μιλήσουμε με τους δικούς τους εμπειρογνώμονες και να ξέρουμε τι πρέπει να γίνει. Υπάρχει δηλαδή μια ευκαιρία να γίνει αυτή η λεπτομερή δουλειά τώρα. Έτσι κι αλλιώς, ό,τι γίνει με τα δικαιώματα θα πρέπει να υπάρξει προς τα πάνω ομοιομορφία, όχι προς τα κάτω. Δεν θα πρέπει να υπάρξει απώλεια δικαιωμάτων, πολιτικών δικαιωμάτων κτλ. Ό,τι είναι διαπραγματευτούν, να το διαπραγματευτούν προς τα πάνω, όχι προς τα κάτω, για να βελτιωθούν τα δικαιώματα αυτά και όχι να χειροτερέψουν. Θέλουμε να υπάρξει ισότιμη μεταχείριση προς τα πάνω, όχι προς τα κάτω. Και γι' αυτό στρεφόμαστε προ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που πιστεύουμε ότι ακριβώ αυτό θέλει. Ευχαριστώ όλους σας ε, τα μέλη του πάνελ, ευχαριστώ και τους ευρωβουλευτές. Είναι φιάλτηση η πέμπτη το απόγευμα. Ξέρετε όταν κάνουμε τέτοια πράγματα πρέπει να προβλέπουμε και το άγχος που προκαλεί αυτό. Ήδη μου έχει στείλει ένα μήνυμα η οικογένειά μου ότι δεν είμαι ευπρόσδεκτο αύριο ή το Σαββατοκύριακο. Χαίρομαι όμως που μείνατε όλοι εδώ. Είναι πολύ σημαντικό και ιδιαίτερα τα άτομα που θα λάβουν μέρος στο επόμενο πάνελ. Ευχαριστώ για την υπομονή σας και περνάμε στο επόμενο πάνελ. Ε, μείνετε παρακαλώ όσο μπορείτε περισσότερο, μας βοηθάτε ιδιαίτερω θα ακούσουμε κάποια ενδιαφέροντα πράγματα. Θα ξεκινήσουμε με τον Τζαν Ντέρφελ, ο οποίος είναι δικηγόρος για θέματα αλλοδαπών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Θα παρατηρήσατε ότι αυτό το τμήμα το έχουμε ε, επεκτείνει σε διάφορους εμπειρογνώμονες. Ε, ξέρω ότι αυτό θα δημιουργήσει τώρα λίγο χάος. Μπορείτε να μην ε, εξαντλήσετε τα 10 λεπτά, μπορείτε λίγο λιγότερο λίγο λιγότερο γιατί δεν έχουμε χρόνο ώστε να προλάβει και ο καθηγητής κ. Πίρες να πει δύο λόγια. Ας είστε συναδελφικοί παρακαλώ. Αλλά και για να ακούσουμε και κάποιες ερωτήσεις ε, θα μας κάνετε μεγάλο χατήρι αν το κάνετε αυτό. Όλες οι παρουσιάσεις ούτως ή άλλως θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα. Πιστέψτε με, οι ευρωβουλευτές ε, παρακολουθούν ε, την απευθείας μετάδοση, μας παρακολουθούν. Έχει μεγάλη προβολή τη σημερινή συζήτηση. Ευχαριστώ την Επιτροπή ΛΥΜΕ και εύχομαι για την πρόσκληση. Ε, ήμουν εδώ και το Μάιο, την περασμένη ακρόαση. Ευχαριστώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως είπε και ο κύριος Γκουαλτιέρη, όλοι μπορεί να είσαστε ιδιαίτερα περήφανοι για τα επιτεύγματα. Αυτά είναι που βλέπετε σε αυτή τη διαφάνεια. Και ούτε που θα το είχα μοιρευτεί εγώ το Μάιο που ήμουν εδώ ότι θα τα καταφέρναμε όλα αυτά. Ε, το δικαίωμα για μελλοντική οικογενειακή επανένωση εξαρτώμενα μέλη στους ανιώντες. Ε, το ανέφερε ο καθηγητής και το είπα και εγώ στην προηγούμενη παρουσίασή μου. Είναι ιδιαίτεροι αυστηροί κανόνες ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο και εμποδίζουν ε, ουσιαστικά την οικογενειακή επανένωση με ε, ενήλικα εξαρτώμενα μέλη στην ανιούσα γραμμή. και αυτό το ξέρουμε διότι οι δύο δαπάνες έχουν προσπαθήσει πάρα πολύ βάσει του Βρετανικού δικαίου και δεν τα έχουν καταφέρει ε, στο παρελθόν. Ε, φυσικά θα πρέπει να υπάρξει μια αρρωγή για την απόδειξη ε, ε της επιλεξιμότητας όταν βλέπουμε κάτι που ξέρουν ήδη οι δικηγόροι ότι το η Υπουργείο Ιστορικών Υποθέσεων βρίσκει τεχνητά λόγους για να απορρίψει αιτήσει, ε, ε, καταλαβαίνουμε πόσο επαναστατικό είναι αυτό το επίτευγμα. Για να περάσουμε στην επόμενη διαφάνεια για να περάσουμε και σε κάποιες λεπτομέρειες. Σάριντερ Σίνγκ, Βλέπουμε ε, ότι το δικαστήριο αναγνωρίζει το δικαίωμα επιστροφής για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν προβλέπεται στην τωρινή συμφωνία. Όσοι έχουν ε, δουλέψει σε κάποια άλλη χώρα θα πρέπει να τύχουν σύνδεση μεταχείριση όπως οποιοδήποτε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι ε, δηλαδή να έχουν την ίδια μεταχείριση με Βρετανούς πολίτες ποτέ δεν είχαν εργαστεί στην Αλλοδαπή. Όμως δεν καλύπτονται και άρα δεν έχουν δικαίωμα για μελλοντική οικογενειακή επανένωση παρά μόνο βάσει τη ιδιαίτερα εθνική εθνικής νομοθεσίας. Ε, και αυτό δεν καλύπτει μόνο τα μέλη που είναι στο Ηνωμένο Βασίλειο, που δεν έχουν ε, τέτοιο καθεστώς μετά το Brexit, ε, διότι δεν καλύπτονται μέσα στην κοινή δήλωση. Αλλά αυτό επηρεάζει και τα μελλοντικά μέλη οικογένειας καθώς και τους υπηκόους που θα επανέλθουν μετά το Brexit αφού έχουν εργαστεί σε κάποια άλλη χώρα και Έχω είχα τέτοιες υποθέσεις, δεν είναι θεωρητική περίπτωση. Πάει κάποιος Βρετανός, πάει στη Μάλτα, έρχεται η Ρωσίδα μητέρα της, γιατί εμένα είναι πολιτογραφημένη, έτσι, αυτή η Βρετανή υπήκος. Και η μητέρα της πάει η Ρωσίδα στη Μάλτα, στο Ηνωμένο Βασίλειο όμως δεν μπορεί να έρθει λόγω αυτής της υπόθεσης Σαρίντερ Σινγκ. Όμως με τη νέα διάταξη θα μπορέσει να επανενωθεί η οικογένεια ε, και για πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου, ξέρετε, θα έχουν αποκλειστεί οι Βρετανοί υπήκοοι σε άλλα κράτη-μέλη. Αυτό είναι η διακριτική μεταχείριση λόγω ηθαγένειας πολίτη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. μόνο και μόνο επειδή δηλαδή είναι Βρετανοί, δεν έχουν την ίδια μεταχείριση όπω άλλοι πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. The, the, the point that όπως είπε η κυρία Μπάρμπαρα Σπινέλη, τα δικαιώματα είναι αναφέρετα και αδιέρετα. Και όταν μιλάμε για derivative rights, αυτό, ε, για, για παράγωγα δικαιώματα, derivative rights, αυτό εννοούμε. Ε, δηλαδή, αυτό είναι στον πυρήνα της ελεύθερης κυκλοφορίας, σε βάση του άρθρου 21. Όμως αυτό επηρεάζει και τα δικαιώματα ηθαγένεια. Άρθρο 20. Θέλει το Ηνωμένο Βασίλειο να αποκλείσει οτιδήποτε απορρέει από το άρθρο 20 γιατί λέει είναι όλοι Βρετανοί. Όχι. Αυτό είναι πλημελές. Και δεύτερον, όσοι έχουν εργαστεί στην Αλλοδαπή πρέπει να έχουν την ίδια μεταχείριση. Όπως πολίτες, οποιοδήποτε πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράγωγα δικαιώματα. Καλύπτει αυτούς που τους περιθάλπουν, τους συγγενείς και τους κηδεμόνες. Δεν περιορίζεται αυτό από την οδηγία 2004-38 γιατί κρίνεται κατά περίπτωση. Γιατί όταν χρειάζεται την περίθαλψη και την αυτού του ατόμου ένας Βρετανό υπηκό. έτσι, γιατί αλλιώς πρέπει να αποχωρήσουν. Και αυτό δεν καλύπτει μόνο ε, την περίπτωση Ζαμπράνο, ε, δηλαδή οι Βρετανοί υπήκοοι που οι γονεί είναι ε, από την Κολομβία, παραδείγματος χάρη, αλλά και ένα, ε, ε, ένα παιδί που, Γερμανών που γεννήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο και επειδή δεν έχει ε, κατοχυρωμένη συνθήκη δικαιώματα και εξαρτάται από τους γονείς πρέπει να φύγει, γιατί μπορεί να είναι υπήκοοι των χωρών. Δηλαδή, ένα παιδί, η μητέρα του είναι Πακιστανή, έχει εκείνο η γερμανική υπηκότητα. Για περάστε στην επόμενη διαφάνεια. Αχμετ Έιμος, έτσι. Ε, στην νομολογία ε, δικαστηρίων του Ηνωμένου ε, Βασιλείου. Πατρεύεται ένας Γερμανός, μία Πακιστανή, χωρίζουν, αλλά στο μεταξύ ζούσαν στο Ηνωμένο Βασίλειο και έχουν δύο παιδιά με γερμανική υπηκότητα και ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και και λέει η, μητέρα ότι άμα δεν μπορούν να μείνουν τα παιδιά μου, δεν, δεν θα μείνω ούτε εγώ. Και λέει το, το δικαστήριο ότι εσείς ε, μπορεί να επικαλεστείτε το άρθρο 20 ε, για το δικαίωμα ηθαγένειας. Για τέλος θα πρέπει να φύγετε ε, και να φύγουν και τα παιδιά σας. Και αυτό είναι άρθρο 20 και όχι 21. Και αυτό δεν υπάρχει καθόλου μέσα στην κοινή δήλωση. Και το ίδιο ε, και για τα παιδιά όσων, ε, των νοσηλευτών παραδείγματος χαρή, όσων περιθάλπουν ηλικιωμένα άτομα. Ή παιδιά. Ε, αυτά εννοούσε η κυρία ε, Σπινέλη. Ένα λιθαράκι να βγάλετε καταραίει όλο το σπίτι και γι' αυτό μιλάμε για τα δικαιώματα και την ερμηνεία τους από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, λένε ότι ισχυρίζονται ότι δεν πρέπει να συμπεριληφθούν ή να συμπεριληφθούν μόνο τα μέλη της οικογένειας οδηγίας. Μα όχι, όχι. Γιατί μπορεί να είναι μία θεία, μπορεί να είναι σύντροφος, ε, κατά περίπτωση θα πρέπει να κρίνεται. Επόμενη διαφάνεια Λοιπόν, ε, ε, ό,τι προκύπτει από το άρθρο 7 του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων ε, οι οικογένειες μένουν εκτός χώρας υποδοχή Νομίζω δεν υπάρχει πρόβλημα, διότι είναι εξαρτώμενα μέλη, μέλη του ε, νοικοκυριού. Ε, και θέλω να απευθυνθώ στην Επιτροπή Brexit για τα παιδιά και να πω ότι Νομίζω ότι υπάρχει και είναι κατανοητό ε, βασική λήψη εμπιστοσύνη για τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου διαπραγματεύσει. Εγώ μπορώ να σα αποδείξω το αντίθετο, διότι όσα παιδιά έχουν αυτά τα παράγωγα δικαιώματα, ε, βάσει της απόφαση Τσέντε Σέιρα θα πρέπει να καλυφθούν ναι, και όχι γιατί τώρα περιορίζεται αυτό στη διάρκεια της εκπαίδευσης. Με το που ε, σταματήσει η φίτηση δεν μπορούν ε, να ζητήσουν παράταση ε, του δικαιώματος γιατί μπαίνουν σε άλλη κατηγορία. Αλλιώς θα μπορούσαν να μείνουν άλλη μία πενταετία. Ε, θα με πιάσει κατάθλιψη αν δεν τα καταφέρουμε. Πολύ θα ήθελα να ανατραπεί αυτό. θα πρέπει να σε αντιμετωπίζει ως αντι, ανεξάρτητους φορείς δικαιωμάτων ε, για να αναγνωριστεί το καθεστώς της μόνης διαμονής ή ένα αντίστοιχο δικαίωμα. Επόμενο. Ε, τι θα συμβεί σε αυτά τα άτομα που αποκλείονται, όπως σας έλεγα. Λοιπόν, βάσει της εταιρείας γίνονται παράνομοι γιατί πρέπει να νομιμοποιήσουν το καθεστώς τους. Και ε, από τη από, επειδή προέρχεται από το Υπουργείο Ιστορικών Υποθέσεων, αυτό ακριβώς εννοεί, έτσι. Και τι σημαίνει αυτό, πολύ ακριβές αιτήσει και Όλα αυτά που προαναφέραμε ε, έχουν μεγάλη σημασία διότι ε, ε, μιλάμε για δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, δικαίωμα στην οικογενειακή επανένωση, είναι η νομοθεσία περί μετανάστευσης. Αυτή είναι η εθρική ατμόσφαιρα και δεν είναι εύκολες υποθέσεις το άρθρο 7. Ε, α, γιατί να τη ποια είναι, ποιο είναι το τέλος. Ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, δυόμιση ε, χρόνια έχουν ε, και έχουν και κοστίζουν 93 λίρες και μετά από δυόμιση χρόνια ξανά τέσσερις φορές και μετά από 10 χρόνια τότε μπορούν να ζητήσουν επαόριστο αίτηση. 269 λίρες και Δύο φορές 65 λίρες, ε, ε, ε, άμα υπολογίσουμε και τα μέλη της οικογένειας. Ε, οπότε όταν ζητάνε 10 χρόνια, αυτό είναι ένα πρόβλημα, κόστους επίσης. Και τι γίνεται με αυτή την υπόσχεση ότι δεν θα ζητήσουν εγγύηση, ότι δεν ε, εξετάζουμε ε, τα πραγματικά χρόνια απασχόλησης. Αυτό θα πρέπει να το διατυπώσουμε και να το συμπεριλάβουμε. Ε, και η οδηγία άρθρο 34. Η 2004-38, έτσι, λέει ότι τα κράτη-μέλη θα διαδίδουν πληροφορίες σε σχέση με τα δικαιώματα και τις ε, υποχρεώσεις ε, όπου προβλέπονται από αυτή την οδηγία κυρίως μέσα από εκστρατείες ε, ευαισθητοποίησης μέσω τοπικών και περιφερειακών ΜΜΕ και άλλων επικοινωνιακών μέσων. Δεν το έχουν κάνει αυτό και δεν χρειάζεται να καταχωρηθεί κάποιος και αυτό δεν το ξέρουν οι άνθρωποι και αυτό είναι παγίδα. Μπορεί να λένε άλλο να, ε, να ζητάμε ε, κατά γράμμα να εφαρμοστεί η νομοθεσία και άλλο να ζητάς να προσυμμορφωθεί κάποιος με κάτι που δεν γνωρίζει. Και μετά γιατί ε, η προσωπική ζωή αυτό είναι πρόσκομα διότι 20 χρόνια χρειάζεστε χωρίς κανένα παράνομο κομμάτι αυτό για τα παιδιά και είναι πολύ, υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικά εμπόδια για την εσωμάτωσή σας στη χώρα προέλευσης. Δηλαδή, αν δεν τους καλύπτει η συμφωνία αυτοί οι άνθρωποι, είναι πολύ δύσκολο, ζωφερή προοπτική, ακριβή και τίποτα δεν τους ε, εγγυάται μια ευτυχή έκβαση στο διάβημά τους. Θα ήθελα λοιπόν να χαρώ και πάλι, είναι εξαιρετικά τα επιτέγματά σας και ε, συμφωνώ και άλλα μπορείτε να πετύχετε ε, και εδώ είμαστε. Θα σας βοηθήσουμε με όποιο τρόπο το χρειάζεται. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ήθελα απλά να πω στην Ανλόρα, είπατε νωρίτερα την εξαίρεση στο, για το GDPR. Η Guardian θα γράψει ένα άρθρο γι' αυτό. Υπάρχει κίνδυνος. Υπάρχει κίνδυνος ε, με προκάλημα διαπραγματεύσεις ε, ε, τώρα η συμφωνία να έχει πολλούς περιορισμούς θα το δημοσιεύσουν σήμερα ήθελα απλά να σας ενημερώσω να ξέρετε πού βρίσκονται οι ευρωβουλευτές να ξέρετε ότι τα ξέρουμε όλα αυτά τώρα για το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, τα, προκαλού, τα παρακολουθούμε. Ευχαριστούμε για την ανάλυση. Πάμε στην Έστερ Λέιν, είναι γραμματέας για το Brexit στο ETC. ETUC. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ που δίνετε την ευκαιρία στους εργαζόμενους στα Συνδικάτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πούμε τις δικές μας απόψεις ε, για αυτό το δικό σας εγχείρημα απολογισμού των διαπραγματεύσεων. Οι εργαζόμενοι στην Ευρώπη αρχίζουν να ανησυχούν όλο και περισσότερο. Ο λόγος είναι ότι εξακολουθούμε να μην έχουμε λάβει σαφείς απαντήσεις. Από τη μία πλευρά έχουμε κάτι εξαιρετικές αρχές, ότι θα συνεχιστεί το δικαίωμα διαβίωσης και εργασίας, αλλά όταν συναντά κανείς εργαζομένους ε, ε, και με ρωτούν είναι για πάντα και εγώ ως νομικός λέω μπα δεν είμαι βέβαιη και εγώ μίλησα πρόσφατα με έναν εργαζόμενο ε, Βρετανό που ζει στην Πρατισλάβα ε, και εργάζεται στην Αυστρία διαμεθοριακός δηλαδή διασυνοριακός εργαζόμενος μου λέει θα μπορέσω να συνεχίσω να το κάνω αυτό τι θα γίνει με την κοινωνική μου ασφάλιση η οικογένεια μου θα μπορεί να είναι μαζί μου Όλοι φωνάζουν και κανείς δεν έχει συμφωνήσει τίποτα. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο για τους εργαζομένους να λάβουν διάφορες αποφάσεις, να πάρω την προαγωγή, να μετακομίσω, εάν επενδύσω σε σπουδές θα μοναγνωριστούν ε, τα επαγγελματικά προσόντα και αυτά έχει τραβήξει τώρα πάνω από χρόνο και δεν φαίνεται να σταματά σύντομα. Οπότε το πρώτο που έχω να πω όσον αφορά τον απολογισμό... είναι ότι πρέπει να δούμε τα πράγματα πιο ρεαλιστικά και να αρχίσουμε να παρέχουμε στους ανθρώπους την ασφάλεια που χρειάζονται για να πάρουν τις αποφάσεις της ζωής τους. Τις αποφάσεις που πρέπει για τη ζωή τους. Το δεύτερο μήνυμα που ήθελα να σας μεταφέρω είναι ότι είναι λίγο επιφανειακές οι συζητήσεις μέχρι στιγμής. Κάτι που δεν βοηθά την κατάσταση. Ναι, μεν θέλουμε μια συμφωνία ε, που λέει ότι θα υπάρχει στις συνθήκες ε, για όλους ε, αλλά μακράν απέχει ακόμα μια νομοθεσία που να το θεσπίζει αυτό που θα επιβάλλει σε έναν εργοδότη να τηρεί κάποιους κανόνες. Πρέπει να φτάσουμε σε τέτοιο επίπεδο λεπτομέρειας οι προηγούμενοι ομιλητέ ε, κατέδειξαν τα προβλήματα στι προτάσει. Από τη δική μου άποψη, απέχουμε μακράν από τέτοιου είδου ε, ρυθμίσει στι προτάσει. Όχι μόνο είναι επιφανειακέ οι προτάσει, αλλά εγώ ανησυχώ όλο και περισσότερο για μια πιθανή παρανόηση ε, του πιο δίκαιο θα ισχύει στους χώρους εργασίας και στους εργαζομένους. Να το πω σύντομα τώρα γιατί μου ζητήσατε να περικόψω την παρουσίαση. Ε, λοιπόν, φανταστείτε τώρα ε, να έχουμε κάποιον άνθρωπο που εργάζεται σε ένα βενζινάδικο όπου σταματάμε στον αυτοκινητόδρομο. Αυτός η όροι βάσει των οποίων εργάζεται διέπονται από ε, την ομοθεσία για τα χημικά, διότι υπάρχουν χημικά εκεί, για τα φαγητά, διότι πουλάει σάντουιτς ενδεχομένω, ε, ασφαλεία, διότι υπάρχει κίνδυνο έκρηξη, ε, κοινωνική ασφάλιση. Μπορεί να δουλεύουν νύχτα οπότε, και να σπουδάζουν την ημέρα, οπότε θα έχουν τα δικαιώματα φοιτητών. Μπορεί να είναι μουσική και να θέλουν να περάσουν τα σύνορα με τα κουβάλλοντα στα αργανά Όλα αυτά ε, καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Όπως είπε η κυρία Σπινέλη, δεν μπορούμε να λέμε ότι με το ένα με το άλλο η νομοθεσία θα λειτουργήσει. Αποκλείται να γίνει αυτό. Θα καταρρεύσει ακόμη και στα πιο βασικά. Η Έχουμε την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για το χώρο εργασία, για τι συνθήκε εργασία, όπω είπαν και οι προλαλήσαντε, και πάνω από αυτό έχουμε όλου του κανόνε που αφορούν την απασχόληση. Και εγώ σκέφτηκα λοιπόν να πάω να διαβάσω την νομοθεσία για να αποκτήσω μια ιδέα του πόσο μακριά είμαστε από οποιαδήποτε ε, λύση. Ξέρετε και μόνο αν διαβάσουμε τα ονόματα ε, των διαφόρων νομοθεσιών που αφορούν όλα αυτά τα θέματα, δεν μας στάνουν τα 10 λεπτά. Οπότε είμαστε τελείως απροετοίμαστοι. Χρειάζεται να εξετάσουμε πάρα πολλά θέματα για να διασφαλίσουμε ε, αυτή την αρχή, αυτές τις αρχές υψηλού επίπεδου που είναι εξαιρετικές μένως αρχές αλλά πρέπει να μπούμε σε λεπτομέρειες για να βεβαιωθούμε ότι θα υπάρχουν απαραίτητες νομοθεσίες και άμα γίνει αυτό μετά τι γίνεται πώ θα εφαρμοστούν αυτέ τι νομοθεσίε είναι το θέμα, διότι θα πρέπει να μπορούν να υποβάλουν προσφυγέ οι εργαζομένοι και κυρίω κατά των εργοδοτών του. Δεν μπορούμε ρεαλιστικά να σκεφτόμαστε ότι θα έχουμε μια συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών με κάποιε όμορφε αρχέ ε, που θα λένε όλα είναι καλά. Δεν θα ανταγωνιζόμαστε όσον αφορά του όρου εργασία. θα σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Από εμπειρία μου, εγώ ως εξωματούχος συνδικάτων, έχω σύρει σε δικαστήρια κυβερνήσει ώστε να τηρούν τις βασικές αρχές της ίσης αμοιβή για τους εργαζομένους. Οπότε χρειάζεται μια πραγματική νομοθεσία που να μπορούν να, ε, να χρησιμοποιήσουν οι εργαζομένοι, να μπορούν να στραφούν κατά των δράσεων των εργοδοτών τους και πολύ συχνά κατά των δράσεων του κράτους ω εργοδότη. Και τέλο ε, θα πρέπει να έχουμε απόλυτη αντίληψη του ότι για τους εργαζομένους ε, ε, πολλά πράγματα στην Ευρώπη δεν λειτουργούν σωστά. Η υποστήριξή μας λοιπόν του ευρωπαϊκού οικοδομήματος ε, βασίζεται στην προσπάθεια εξάλληψης της εκμετάλλευσης. Δεν είναι ότι θα δημιουργηθεί αυτή η εκμετάλλευση αν ε, δεν είναι επαρκής η όρηση αυτής της συμφωνίας εδώ. Το πρόβλημα είναι ότι σε ολόκληρη την Ευρώπη πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρχει εκμετάλλευση των εργαζομένων. Και εγώ μιλώντας ως μητέρα με Ιρλανδό πατέρα και Αγγλίδα μητέρα δεν μπορώ να μην αναφέρω τέλος τα σύνορα της Βόρειας Ιρλανδίας τόσο ριζική σημασία. Το σύνορα αυτά τα οποία δεν πρέπει να επανέλθουν. Πολλοί κόσμος, λένε, πολλοί κόσμος λέει αν δεν υπάρξουν διαπέρατα ε, σύνορα τα πράγματα θα είναι εντάξει. Μόλις θα υπάρξει κάποιος με στολή, πιθανότατα με ένα όπλο, σε ε, ένα φυλάκιο που θα χωρίζει τη Βόρεια και μόνο αυτό θα μας πάει πίσω. Γι' αυτό είχαμε μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είμαστε Ευρωπαίοι, για να σταματήσουν να υπάρχουν τέτοιου είδους διαφορές. Ευχαριστώ. Thank you Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα μας είπατε. Ευχαριστούμε. Τώρα με ιδιαίτερη χαρά θα σας παρουσιάσω την ε, Τζούλια Όσλο Κόουλ που είναι επικεφαλής προσταμένη του Τμήματος Παγκόσμιας Μετανάστευσης στην Price Waterhouse Coopers. Για πολύ καιρό ασχολείται με αυτά τα θέματα και πολύ χαίρομαι που βρίσκεται εδώ σήμερα μαζί μας. Τζούλια, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ, Κλοντ. Και εγώ χαίρομαι πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να μοιραστώ μαζί σας τις εμπειρίες μου. Είναι πολύ σημαντικό οι ευρωβουλευτές να συμμετέχουν στον διάλογο που συνεχίζεται για να μην υπάρχουν κενά για τις επιχειρήσεις. Θα μιλήσω λοιπόν από την οπτική γωνία ακριβώ των επιχειρήσεων. Τώρα επιπλέον ότι είμαι επικεφαλής στην παγκόσμια μετανάστευση, στην PwC, είμαι και στο Δημαρχείο υπεύθυνη του Λονδίνου, υπεύθυνη για τα θέματα του Brexit και πρόσφατα ε, ορίστηκα και στο Υπουργείο Εσωτερικών στο θέμα της ε, μετανάστευσης ε, και εργοδοτών. Έχουμε πάρα πολλές ε, αιτήσει για θέματα μετανάστευσης και από τον ρόλο που έχω εγώ αντιλαμβάνομαι πολύ καλά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο επιχειρηματικό κόσμος σε σχέση με το Brexit. Και μετά το δημοψήφισμα συζητάω με επιχειρήσεις πολλών κλάδων από startups μέχρι μεγάλες πολυεθνικές για να καταλάβω τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν εκείνοι, εργοδότες και εργαζομένοι τους. Από την τελευταία φορά που ήρθε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει υπάρξει βέβαια πρόοδος όσον αφορά τους πολίτες και οι επιχειρήσεις χαίρονται για την ε, κοινή έκθεση. Πρέπει όμως ε, να πούμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών είχε πολλές δυσκολίες προκειμένου να αντιμετωπίσει τις συνέπειες του Brexit. Και νομίζω ότι ένα από τα πράγματα που πρέπει να πούμε εδώ ότι το Υπουργείο Εσωτερικών δημοσίευσε ε, πολλά, πολλές ειδήσει για το πώς αντιμετωπίσει τις δυσκολίες και τις προκλήσεις αυτές και αυτό είναι κάτι πολύ θετικό. Αν δούμε τα στοιχεία, πριν από το δημοψήφισμα, οι αιτήσει που είχαμε για μόνιμη ε, διαμονή ήταν 24.000 τρίμηνο Το πρώτο τρίμηνο του 2017 όμως έλαβαν πάνω από 127.000 127.500 αιτήσει και το προσωπικό αντίστοιχα αυξήθηκε μόνο κατά 5%. Το Υπουργείο Εσωτερικών λοιπόν εξετάζει πώς θα σχεδιάσει το νέο σύστημα καταγραφής των αιτήσεων αυτών για να διευκολύνει τους Ευρωπαίους πολίτες και να μην τους φορτώνει με πολλή γραφειοκρατία. Όπως είπε και κάποιος άλλος νωρίτερα, σήμερα είμαστε απέναντι σε μια μεγάλη ευκαιρία. Το Υπουργείο Εσωτερικών προσπαθεί να διασφαλίσει ότι θα πρόκειται για ένα εντελώ νέο σύστημα που θα συνδέεται και με άλλα τμήματα κυβερνητικά, έτσι ώστε να μπορούν από μόνοι του να βρίσκουν πληροφορίε και να μην χρειάζεται να τι απαιτήσουν από του πολίτε. Και έχω δει μια πρώτη εκδοχή του νέου αυτού συστήματο και πραγματικά πιστεύω ότι ανταποκρίνεται στι προσδοκίε μα όσον αφορά την απλοποίηση. Επιπλέον ξέρω ότι το Υπουργείο Εσωτερικών συνεργάζεται με τους ενδιαφερόμενους και με διάφορες ομάδες ενδιαφερομένων με ιδιαίτερη προσοχή στην βελτίωση της επικοινωνίας, κάτι το οποίο χρειάζονται και οι Ευρωπαίοι πολίτες και οι επιχειρήσεις. Παρόλη αυτή τη δουλειά όμως και την πρόοδο, αυτό που διαπιστώνουμε από τις επιχειρήσεις, από όλες τις επιχειρήσεις, όλο τον επιχειρηματικό κόσμο, είναι ότι νιώθουν μεγάλη ανησυχία και είναι μπερδεμένοι και δεν ξέρουν τι πρέπει να αποφασίσουν, να μείνουν, να φύγουν από το Ηνωμένο Βασίλειο. Και είναι κάτι το οποίο επηρεάζει τελικά και την καθημερινότητά του, να δουλέψουν σε καθημερινή βάση. Έχει επιπτώσεις στη ζωή του. Και το είδα και αυτό από πρώτο χέρι πώς επηρεάζονται και οι επενδύσεις των επιχειρήσεων, κυρίως στους κλάδους εκείνους που βασίζονται πολύ στο ευρωπαϊκό εργατικό δυναμικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε λοιπόν, στις διάφορες εκθέσεις φαίνεται ότι όλοι ανησυχούν για το μέλλον τους και γι' αυτό είναι ζωτική σημασία να υπάρξει σαφής επικοινωνία ώστε να ενημερώνονται σωστά και επιχειρήσεις και οι Ευρωπαίοι πολίτες καθώς επίσης και οι πολίτες οι Βρετανοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και άλλη φορά είχα πει εδώ ότι ο ΠΟΕ είχε, μάλλον συγγνώμη, ότι η PwC είχε, πάρει, είχε κάνει πολλές έρευνες και έχουμε και την κοινή έκθεση με την London First με τίτλο Facing Facts. Εκεί κοιτάξαμε τι γίνεται με το εργατικό δυναμικό στο Λονδίνο 10 χρόνια και διαπιστώσαμε ότι κάθε μετανάστη συνεισφέρει με 46.000 λίρες το χρόνο σε καθάριστη αξία το έτος και έχουμε 1,8 εκατομμύρια μετανάστες που προσφέρουν συνολικά 83 δισεκατομμύρια που είναι ουσιαστικά το 1 τέταρτο του του Λονδίνου. Επίσης, κάναμε μια έρευνα και στον Ταβός όπου ρωτήσαμε διευθύνοντες συμβούλους, 1.300 συγκεκριμένα και όλοι μας εξέφρασαν τις ανησυχίες τους ε, τους τελευταίους 12 μήνες. Το 80% από αυτούς είπαν ότι ανησυχούν ιδιαίτερα για το κατά πόσο θα μπορέσουν να διατηρηθούν οι δεξιότητες και κυρίως Βρετανοί ε, διευθύνονται σύμβουλοι το είπαν αυτό. Και είναι ενδιαφέρον να δούμε ότι το 2013 η η ανησυχία τους ε, αυξήθηκε πάρα πολύ σε σχέση με σήμερα. Φοβούνται δηλαδή ότι δεν θα υπάρχουν αρκετά προσόντα στο εργατικό δυναμικό μετά το Brexit. 88% αυτών των ε, διευθυνόντων συμβούλων παρόλα αυτά πιστεύουν ότι θα διαβριθούν οι επιχειρήσεις τους, θα μεγαλώσουν. Αν δούμε λοιπόν όλους αυτούς ε, τους δείκτες για την ανάπτυξη, την ε, ανεργία, τον πληθωρισμό και όλα αυτά, ε, διαπιστώνουμε πόσο μεγάλη είναι η ανησυχία στα πλαίσια μάλιστα και της οικονομικής κρίσης που μόλις περάσαμε. Οπότε δεν μας εκπλήσει το γεγονός ότι θέλουν οι διευθύντες αυτοί σύμβουλοι να βρούνε προσόντα και δεξιότητες στον κόσμο για να αναπτυχθούν ακόμα περισσότερο. Είναι σημαντικό λοιπόν να πούμε ξανά ότι χρειαζόμαστε καλή στρατηγική επικοινωνίας Ελπίζουμε ότι θα διαλυθούν κάποιες από τις αβεβαιότητες που υπάρχουν σήμερα. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, επιχειρήσεις ε, κοιτούν μπροστά και περιμένουν να δούνε τι θα αποφασιστεί για τη μεταβατική περίοδο και τι θα συμβεί μετά την μεταβατική αυτή περίοδο. Επίσης, οι επιχειρήσεις θέλουν οι Ευρωπαίοι πολίτες που μπαίνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου θα έχουν τα ίδια δικαιώματα όπως και εκείνοι οι οποίοι μπήκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν από τον Brexit. Αυτό θα βοηθήσει να υπάρχει βεβαιότητα για αυτούς. Οπότε θα ολοκληρώσω λέγοντας ότι η μεταβατική περίοδος, οι διευθετήσεις για αυτήν και Όλα αυτά θα διευκρινιστούν πολύ σύντομα με όσο γίνεται λιγότερα προβλήματα για τους Βρετανούς που ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους Ευρωπαίους που ζουν στον Ηνωμένο Βασίλειο. Για παράδειγμα, σε απασχολούν θέματα που έχουν να κάνουν με τον αυτοματισμό, τη ρομποτική και τις θέσεις απασχόλησης του μέλλοντος. Πρέπει να υπάρξει συμφωνία για την περίπτωση αυτών των πολιτών όσο γίνεται πιο γρήγορα και αυτό να είναι προτεραιότητα για μας. Ευχαριστούμε. Τώρα περνάμε στους δύο τελευταίους ομιλητές, μόνο στον τελευταίο ομιλητή, στον Τζόναθαν Πόρτες, τον καθηγητή. Έχουμε κι άλλον ένα έκδοση μετά. Είναι καθηγητές και δύο. Αλλά κάτι παραπάνω από καθηγητές. Συνεισφέρουν πάρα πολύ στην στρατηγική μας και στην ανάλυση για τα θέματα που μας απασχολούν. Ο κύριος Πόρτες ο καθηγητής οικονομικών από το King's College. Αναλυτής για θέματα μεταναστευτικής πολιτικής. Θα σχολιάσει για το Brexit, σίγουρα με έναν ιδιαίτερα καλό τρόπο. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Τζόναθαν. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια και ευχαριστώ και για την πρόσκληση. Χαίρομαι που ήρθα Θέλω να είμαι σύντομο και θα παραλείψω κάποια πράγματα, ώστε να προσπαθήσω να δώσω μια μελλοντική προοπτική σε σχέση με τη συμφωνία του Δεκεμβρίου. Πιστεύω ότι οι λαλίσαντε μα κάλυψαν για πάρα πολλά πράγματα, χρειάζεται να τα επαναλάβω. Επόμενη διαφάνεια. Λοιπόν, η συμφωνία του Δεκεμβρίου. Ε, ε, εγώ δεν μπορώ να σας δώσω τόσο λεπτομέρειες όσο οι προηγούμενοι ομιλητές, οπότε πάμε στο επόμενο. Σε τι πρέπει να εστιάσει την προσοχή το Κοινοβούλιο. Οι τρεις πρώτες τελείωσε καλύφθηκαν από τους προραλίσαντες, αλλά την τελευταία δεν νομίζω να την ανέφερε κανείς. Και εσύ. Το καθεστώς δηλαδή της ανεξάρτητης Εθνική Αρχή. Αυτό αναφέρεται στη Συμφωνία του Δεκεμβρίου. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή η ανεξάρτητη αρχή να έχει ξεκάθαρο νομικό καθεστώ, να είναι πραγματικά ανεξάρτητη και να εκπροσωπεί τα συμφέροντα και τα δικαιώματα των πολιτών και να έχει ουσιαστικέ εξουσίε. Mm-hmm. τα τελευταία χρόνια το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει πολύ ε, καλά αποτελέσματα. Ε, σε αυτό το τομέα δηλαδή ε, σε σχέση με τι ανεξαρτητέ αρχές θα χρειαζόμαστε λοιπόν την κλίση ασφαλείας για να μην μπορέσει η Βρετανική κυβέρνηση να το αγνοήσει. Ε, δεν είναι ένα από τα ζητήματα που ακούγονται περισσότερο αλλά θα έχει μακροπρόθεσμη επιπτώσει σε σχέση με την εφαρμογή της ε, συμφωνίας. Είναι πάρα πολύ κέριο αυτό το πολιτικό ζήτημα με το που κλείσει, κλειδώσει η συμφωνία ο, οποιοδήποτε ε, θα έχει στις Βρυξέλλες πάρα πολύ ε, περιορισμένες δυνατότητες πλέον επιρροής. Ε, δηλαδή θα μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα στις σχέσεις του ΕΒ Βασιλείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά σε πρωτογενές και δευτερογενές επίπεδο, δηλαδή στην εφαρμογή της συμφωνίας στη νομική και διοικητική δομή του ΕΒ δεν θα υπάρχει δυνατότητα επιρροής επόμενη διαφάνεια, το Standstill Agreement, ε, η μεταβατική περίοδος, ε, όπως έγραψαν και στο tweet από, την, ε, από το επιτελείο του κύριου Μπαρνιέ, δηλαδή η διατήρηση του status quo είναι το αντίθετο της μετάβασης. Και εδώ μιλάμε για διατήρηση του status quo και όχι για μετάβαση. Πώς συμφιλιώνεται λοιπόν τις δύο απόψεις, ε, πολιτική και νομική, ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ε, του Ηνωμένου Βασιλείου. Τι γίνεται για να φτάσουμε μετά το Brexit, μετά το πέρασε την εκνοή αυτής της περίοδου διατήρησης του κεκτημένου και μετά από αυτή την περίοδο λοιπόν ε, Μετάβαση μπορούν να διαμείνουν και μπορούν, θα έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν ε, μόνιμη διαμονή. Ε, να σας δώσω κάποια στοιχεία απάντησης. Ε, η θέση του Ηνωμένου Βασιλείου ε, έχει ε, κάποια λογική. Όσοι έρχονται μετά τον Brexit δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα με αυτούς που υπακούν σε συγκεκριμένες κανόνες όσο ήταν κράτος μέλος του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί οι κανόνες σε αυτή τη μεταβατική περίοδο ούτως ή άλλως θα έχουν προκαθοριστεί πριν τις 29 Μαρτίου 2019. Όλοι θα τους ξέρουν τους κανόνες δηλαδή ξέρουμε όμως ότι δεν είναι στην πράξη δεν είναι δύσκολο εφαρμόζεται αυτή η θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και θα οδηγήσει σε μεγάλη σύγχυση και χάος. Ε, όποιος έρχεται κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περίοδου, τι θα κάνει δηλαδή μετά, θα είναι σε λίμπο, σε μια ε, αδιευκρίνηστη νομική θέση μετά την εκπνοή της περίοδου. Ε, και αυτά θα διευκρινιστούν πολύ αργότερα και ε, κατά πάσα πιθανότητα πολύ μετά την έναρξη αυτής της μεταβατικής ε, περίοδου διότι ε, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν λέει πολλά σε σχέση με το σύστημα όπως θα ισχύει μετά το, το, Brexit. Οπότε όσοι θέλουν μετά το Brexit ναι, από τα 27 κράτη-μέλη να πάνε στο Ηνωμένο Βασίλειο για οικογενειακή επανένωση, για δουλειά, για οποιοδήποτε λόγο, αλλά δεν ξέρουν ποιο θα, ποιο θα είναι το νομικό καθεστώς του μετά από 2,5 χρόνια. δεν είναι απαραίτητο αυτό και για τους πολίτε και για τις οικογένειές τους και για τους τους ε, εργοδότες. Από πλευρά ε, του ακαδημαϊκού κόσμου, του Πανεπιστημίου, παραδείγματο χάρη, προσπαθούμε να προσελκύσουμε ανθρώπους. Θα αρχίσουμε έτσι ε, του χρόνου και του παραχρόνου. Τι θα τους πούμε ότι μετά από 18-20 μήνες δεν ξέρουμε τι καθεστώς θα έχουν. Ναι, δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό. Το ίδιο και για τον τομέα υγείας λοιπά. Ε, αν θέλει αλλακτική το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να δώσει κάποιες πρακτικές αλλακτικές ε, λύσεις ε, για να διαφύγουμε αυτή την κατάσταση και προς το παρόν δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Επόμενη διαφάνεια. Λοιπόν, δεν θέλω τώρα να περάσω το χρόνο που μου έχει απομείνει γιατί δεν σχετίζεται με τα δικαιώματα, δηλαδή το πλαίσιο για τις μελλοντικές σχέσεις, διότι αν όλα πάνε καλά και συνεχίσουν τι πρόοδο στι συνομιλίες. Πολύ σύντομα θα ε, εγγραφεί στο θεματολόγιο αυτό και πρέπει να ε, διαμορφώσει θέση στο Κοινοβούλιο. Από πλευρά των 27 ε, και το Ηνωμένο Βασιλείου. Δεν ξέρω αν κάποιοι θέλουν να μιλήσουν για την ε, ε, κινητικότητα του εργατικού δυναμικού και για τη μετανάστευση. Υπάρχουν συγκεκριμένα οικονομικά πλεονεκτήματα για τη συμπερίληψη τη κινητικότητα του εργατικού δυναμικού σε αυτό το πλαίσιο. Ξέρουμε κυρίω σε σχέση με εμπορικέ υπηρεσίε. Έτσι, γιατί υπάρχουν ε, ε, κοινά στοιχεία, ακόμη και η ΣΥΤΑ η συμφωνία έχει κάποια ε, στοιχεία, διότι σχετίζεται με πολυεθνικές επιχειρήσεις και άρα συμπεριλαμβάνει ζητήματα κινητικότητα ε, ε, στο εργατικό δυναμικό, αλλά όχι μόνο. Και λοιπόν ξεκάθαρα θα είναι υποφελές να υπάρχει αυτή η κινητικότητα εργατικού δυναμικού και ε, στις δύο πλευρές ε, αλλά μπορεί και να μην συμπεριληφθεί. Οι μετανάστε είναι πολύ πιο προβληματικοί από πολιτική σκοπιά ε, σκοπιάς ε, και πολύ ευκολότερο είναι καμία πλευρά να μην φέρει τη μετανάστευση σε αυτές τις ε, συζητήσεις που νομικός, νομικός και τεχνικό θα είναι εξαιρετικά περίπλοκες. Ε, και άλλοι ξέρουν καλύτερα και από μένα ότι υπάρχουν ιδιαίτερε νομικέ περιπλοκέ ε, αν ε, επεκτείνουμε το καθεστώ στου μετανάστε, κυρίω είναι αρμοδιότητα εθνική. Και όταν μιλάμε για συμφωνίε με επιχειρήσει που έχουν την έδρα του σε τρίτη χώρα, καταλαβαίνετε πόσο περιπλέκεται αυτό. Έχει κάνει χρήσιμε αξιολογίε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά για αυτό το θέμα, ποιο θα είναι ο οικονομικό αντίκτυπο συγκεκριμένων ελεκτικών λύσεων για την κινητικότητα του δυναμικού Οικονομικού ε, Συμμελλοντική Συμφωνία. Αυτό πρέπει να ε, ε, βιληφθεί αυτό το ζητήμα άμεσα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί θα προκύψει σύντομα. Επόμενο. Επίση πιστεύω και αυτό σχετίζεται με αυτό που μα είπε και ο Ρότζερ προηγουμένω. Πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να αλλάξει γνώμη το Ηνωμένο Βασίλειο. Όχι μόνο για, ε, όχι απαραίτητα για το Brexit, αλλά για την ελεύθερη κυκλοφορία. Δύσκολο και ακαθόδεσαι αυτό το ζήτημα από πολιτική σκοπιά. μπορούμε μόνο να υποθέσουμε ότι το είναι κυβέρνηση, τον είναι πρωθυπουργό ε, και η, τον είναι για τι διαπραγματεύσει ε, θα παραμείνουν στην εξουσία. Μπορεί, ναι, μπορεί και όχι όμω. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα ανέβει άλλο κόμμα στην εξουσία. Δεν το ξέρει κανεί αυτό. Υπάρχουν διάφορα πολιτικά σενάρια. Όμως το ότι το, το, το, το κυβερνών κόμμα έχει ε, αποκλείσει την ελεύθερη μετακίνηση, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι αμετάκλητα μετακίνητη θέση, μια πλειοψηφία στο κοινοβούλιο και στο εκλογικό σώμα, ενδεχομένω να ε, διαφωνήσει. Οπότε ας ετοιμάσουμε ένα πλάν B, ένα εφεδρικό σχέδιο, αν το Ηνωμένο Βασίλειο αποφασίσει να ε, κάνει reset στη διαπραγματεύσεις και να ε, ακολουθήσει αυτές τις γραμμές. Ναι, ναι, ε, ψηφίσαμε για τον Brexit, θα φύγουμε, αλλά ε, απειχώντας τις απόψεις στο Ηνωμένο Βασίλειο ότι ε, η πολιτική του Ηνωμένου Βασιλείου είναι ασύμβατη με την πολιτική δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως θέλουμε να διατηρήσουμε τις ε, ε εμπορικές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε τις κόκκινες γραμμές του Μαΐου, της ε, Τερέζα Μέη. και, αυτό τι σημαίνει για τα εμπορικά ζητήματα ελεύθερη κυκλοφορία. Αν ε, αυτό γίνει και ε, επανδημορφωθούν διαπραγματεύσεις, τότε θα πρέπει να αποφασίσουμε ακριβώς ποια μορφή ελεύθερης κυκλοφορίας σε συνάδει με ε, τα πρωτόκολλα και τις δομές του, της ενίας αγοράς, γιατί έχουμε και την Ελβεδία και το Λίχτενστάιν αναγνωρίζουν όλοι την, επί της αρχής ε, το δικαίωμα ελεύθερης ε, ε κυκλοφορίας, αλλά έχουν πολύ διαφορετικό νομικό πλαίσιο για την εφαρμογή του ε, για τους υπηκόρους των 27. Πολύ δύσκολα και πολυδιάστατα και πολυσύνθετα νομικά προβλήματα. Μπορεί να μην συμβεί αυτό, όμως εάν φτάσουμε σε αυτό το σημείο θα είναι εξαιρετικά ατυχές να μην έχουμε κάνει την απαιτούμενη προβασκευαστική εργασία, τόσο ώστε και από τις δύο πλευρές να είναι έτοιμοι οι διαπραγματευτές. Σε περίπτωση έτσι που επανέλθουν στις θέσεις τους και εγγραφεί αυτό το θέμα, ε, που είναι ραγδαίες εξελίξεις ε, πολιτικές ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο, το, είπαμε, το είδαμε αυτό τα τελευταία χρόνια. Έχω σε μία μελέτη παραθέσει τις διάφορες εναλλακτικέ, αλλά πρέπει να μελετηθούν περαιτέρω. Αυτά και σταματάω. Βλέπετε τι επίπεδο είναι οι ομιλητέ εδώ. Αξίζει τον κόπο μια επίσκεψη στην ιστοσελίδα. Εμείς θα μεριμνήσουμε όλες οι παρουσιάσεις εδώ να διαβιβαστούν και στην διευθυντική ομάδα του Brexit και στο προσωπικό κατά τη συζήτηση. Ο κ. Γκουαλτιέρη ανέφερε ότι όλα αυτά του είναι χρήσιμα. Αυτό είναι και ο σκοπό τη ακρόαση, να φτάσουν στην Διευθύνουσα Επιτροπή του Brexit όλα αυτά και στου ε, ευρωβουλευτέ που δραστηριοποιούνται στον τομέα. Αυτό είναι κρίσιμη σημασία. Θα μεριμνήσουμε λοιπόν να διαβαστούν και στου ευρωβουλευτέ που δεν είναι παρόντε. Τελευταίο ομιλητή, ε, υπό το ίδιο πνεύμα, εξέχων ακαδημαϊκός ε, ε, στον τομέα. Αν δεν τον ακολουθείτε στο Twitter, ε, σας προτείνω να το κάνετε. Παρότι έχει αρκετούς ακολουθούς, είναι ο καθηγητής Steve Pierce. Ε, Steve, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για την περιγραφή σας του ατόμου μου. Θέλω να εστιαστώ στη συμφωνία αποχώρησης, παρότι δεν έχουμε δει ακόμα το προσχέδιο. Διότι αυτό αναπόφευκτα θα αποτελεί στο επίκεντρο των συζητήσεων. Και αυτό θα επικυρωθεί ως βάση νομική για πολλά χρόνια στο μέλλον. Ε, όταν θα έχουμε ξεχάσει τις κοινέ εκθέσεις και τις κατευθύνες ε, γραμμές για διαπραγμάτευση, η συμφωνία απαχώρησης θα είναι το βασικό νομικό κείμενο στο τέλος και θέλω να σας πω και δύο λόγια για το κατά πόσο θα πρέπει να υπάρχει μονομερής ευρωπαϊκή νομοθεσία για το ζήτημα των Βρετανών πολιτών. Για τη συμφωνία αποχωρησής υπάρχει ένας κίνδυνος. Μόλις εμφανιστεί κάποιο προσχέδιο, ακόμη και πριν, αν κυκλοφορήσει οποιοδήποτε προσχέδιο, ακόμη και αν δεν έχει δημοσιοποιηθεί, όλη η προσοχή θα πάει στο ζήτημα των συνόρων με τη Βόρεια Ιρλανδία. Διότι αν διαβάσετε τι διάφορε εκθέσει, το κομμάτι για του πολίτε, τι οικονομικέ αποζημιώσει, όλα αυτά μπορούν να μεταφραστούν σε νομικό κείμενο εύκολο. Το Ιρλανδικό, τα Ιρλανδικά σύνορα είναι κάτι. Ε, είναι ένα επίμαχο θέμα, ένα θέμα που πονάει. Είναι πολύ δύσκολο να το συντάξει κανεί ω νομικό κείμενο. Γι' αυτό το λόγο δικαίω ε, λαμβάνει τεράστια προσοχή. Είναι πολύ σημαντικό, αλλά μην ξεχνάμε το ζήτημα των πολιτών Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ενωμένου Βασιλείου, διότι και αυτοί θα αναφέρονται σε αυτή τη συμφωνία αποχώρηση. Τα βασικά στοιχεία, τα βασικά νομικά στοιχεία για αυτού θα βρίσκονται εκεί. Να επισημάνω κάποια βασικά ζητήματα. Πρώτα απ' όλα το γενικό ερώτημα, πώ μπορούμε να επηρεάσουμε τη συμφωνία αποχώρηση. Δεν ξέρω τι γίνεται στη διευθύνουσα του Brexit. Έχετε δει κάποιο προσχέδιο, μπορείτε να κάνετε συστάσει αυτή τη στιγμή. Κάποια στιγμή θα δημοσιοποιηθεί το κείμενο και εμεί εξωτερικοί θα μπορέσουμε να αρχίσουμε να σχολιάζουμε και να κάνουμε και συστάσεις για τροποποιήσεις ε, που ευχόμαστε να τις δείτε και εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο. Θα υπάρξει αυτή η διαδικασία και πολλοί εμείς ε, εξωτερικοί έχουμε ήδη προετοιμάσει κάποια κείμενα για τροποποιήσεις γιατί έχουμε και ψηδές για το τι πρέπει να αναφέρεται στη συμφωνία αποχώρησης. Ποια είναι τα βασικά ζητήματα. Πρώτα απ' όλα η οποπτική αρχή Βάσει τον, είπε, είπε όσων είπε ο κ. Πόρτε, συνεχίζω λέγοντα είναι σημαντικό ζήτημα, χαρακτηρίζεται από τρία στοιχεία. Αυτονομία, εξουσίε και πόροι του εποπτικού οργανισμού για του ε, Βρετανού ε, πολίτε που θα, που θα ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ελπίζουμε ότι και η Κομισιόν θα κάνει τη δουλειά τη όσον αφορά τα δικαιώματα των Βρεταμονών πολιτών ε, στι 27 χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εκεί θα πρέπει να υπάρχει κάποιο κείμενο. Αλλά για τα ζητήματα αυτά για αυτό τον νέο οργανισμό στο Ενωμένο Βασίλειο είναι σημαντικό να διασφαλίζεται πρώτα απ' όλα η αυτονομία του ε, Στη 31 Δεκεμβρίου ε, προσπάθησε να κάνει το Ενωμένο Βασιλείο έναν τελείως λάθος διορισμό στη ρυθμιστική αρχή του Ενωμένου Βασιλείου ε, να βάλει κάποιον τελείως ακατάλληλο ως, αξιωματούχο της ρυθμιστικής αρχής κάποιον που είπε κάτι για νομολογία περί αρχών η εξουσία αυτού του οργανισμού θα πρέπει να αποφασιστεί να μην είναι απλά συμβουλευτικό. Είναι σημαντικό να αποφασίσουμε αν θα έχει τι εξουσίε που έχει και μια αρχή προστασία δεδομένων. Θα λέει δηλαδή στην κυβέρνηση τι να κάνει. Και αν θα έχει το δικαίωμα να προσφύγει στα δικαστήρια. Αυτό μα οδηγεί στο ζήτημα των πόρων. Είτε λαμβάνει απόφασεις, είτε ε, καταφεύγει κατά της ε, κυβέρνησης εκ μέρου των ε, πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να έχει πόρους. Δεν θέλουμε να φτάσουμε στην κατάσταση της, Ευρωπαϊκής, της Ιρλανδικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων που ουσιαστικά είναι λειτουργεί μόνο με στο Facebook, έτσι φαίνεται. Δεν θέλουμε να φτάσουμε σε τέτοια κατάσταση. Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα είναι η εγγραφή. Κατά πόσο θα εγγράφει τους πολίτες σε Μητρό το Ηνωμένο Βασίλειο, τους πολίτες της το ερώτημα είναι θα συμμορφωθεί το νομό Βασίλειο με τους περιορισμούς αυτής της οδηγίας που θέτει κάποια όρια για το τι μπορεί να κάνει κανείς με την εγγραφή για ε, Ευρωπαίων πολιτών ως αλλοδαπών. Πρέπει να φροντίσουμε λοιπόν η συμφωνία που χωρίς να αναφέρει ρητά αυτά τα, αυτούς τους περιορισμούς εγγραφής. Ε, ένα άλλο ερώτημα είναι οι ρυθμίσει για τη μόνιμη εγκατάσταση για του πολίτε τη Ευρώπη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και εδώ υπάρχει πρόβλημα. Γίνεται αναφορά σε κάποιο εσωτερικό έγγραφο του Ηνωμένου Βασιλείου και δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια πρόθεση να γίνουν νομικώ δεσμευτικέ οι δεσμεύσει του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτά είναι βασικά ζητήματα που θα παίξουν σημαντικό ρόλο στι ζωέ πολλών ανθρώπων. Για παράδειγμα, έλεγχοι ποινικού του Ηνωμένου Βασιλείου ήδη έχει κακό μητρό για τους δικαίους του ε, πολίτες. Ο καθένας μας πρέπει να έχει ποινικό μητρό. Η γυναίκα μου είχε ένα πρόβλημα γιατί δεν διαχειρίστηκε σωστά τον έλεγχο η τοπική αρχή και χρειάστηκε να διαμαρτυρηθούμε. Αν το συγκρίνετε αυτό και δείτε το πόσα εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται ήδη στο Ηνωμένο Βασίλειο, αν δεν τα καταφέρνει με τόσο μικρό αριθμό το κράτος μας, καταλαβαίνετε τι πρόβλημα θα δημιουργηθεί. Πρέπει να δούμε λοιπόν πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό. και η αποποίηση της απέτηση ε, ολικής ε, ασφαλής υγείας. Ε, και εκεί και το ζήτημα της, του φίλου και οι γονείς που παραμένουν στο σπίτι. Για κάποιο τρόπο πρέπει να λάβει το Ηνωμένο Βασίλειο κάποια δέσμευση. Θέλει το Ηνωμένο Βασίλειο να υπάρχει και κάποια αναφορά στη συμφωνία για τη μελλοντική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι λογικό Αναφέρεται και στο άρθρο 50 κάτι παρόμοιο, αλλά θα πρέπει να γίνονται και νομικώς δεσμευτικά εσύ δεσμεύσει του Ηνωμένου Βασιλείου με κάποιο τρόπο. Για να αναφερθώ σε κάποια άλλα σημαντικά ζητήματα, η κατάσταση ε, όπως την υπόθεση της Ρέγγια οι άνθρωποι που φεύγουν και ξαναέρχονται, ε, Έχουμε και την υπόθεση ενό Ολλανδού πολίτη που πήγε στον Ηνωμένο και επέστρεψε στην Ολλανδία. Πρέπει να είναι αμφίδρομη δηλαδή ε, η κάλυψη. Έχουμε έτσι υποθέσει Ζεμπράνου, Βρεταν, ε, παιδιά που έχουν βρετανική υπηκότητα χωρί Βρετανού γονεί και αυτά πρέπει να καλυφθούν και στη μεταβατική συμφωνία. Υπάρχει κίνδυνο να παραληφθούν τα παιδιά αυτά και οι γονεί του. Διότι το δικαίωμα βασίζεται σε ηθαγένεια και όχι στη νομοθεσία ελεύθερη κυκλοφορία. Οπότε επιχείρημα θα είναι ότι αφού δεν είναι πλέον το νομοβασίλειο κράτο οι Βρετανοί πολίτες δεν είναι πλέον πολίτες της Ένωσης. Οπότε θα πρέπει να βρεθούν συγκεκριμένα λόγια, συγκεκριμένα κείμενα για να καλυφθούν όλα αυτά. Και η Judith Κιόρτον Darling αναφέρθηκε στην Ιθαγέρια σε σχέση με τα δικαιώματα ψηφοφορίας και τα δικαιώματα ε, να εκλεγεί κάπου. Κάποιος ε, είναι το ίδιο είδους ζήτημα. Ε, διατήρηση δηλαδή κάποια μορφή ηθαγένεια ακόμη και μετά, Ευρωπαϊκή ηθαγένεια ακόμη και μετά από την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου. Και μετά ήθελα να σας παροτρύνω να σκεφτείτε κατά πόσο θα έπρεπε να υπάρχει νομοθεσία ευρωπαϊκή για τους Βρετανούς πολιτέ σε δύο περιπτώσεις. Πρώτον, σε περίπτωση που ε, εξακολουθήσει να υπάρχει το δικαίωμα ελεύθερη κυκλοφορία επειδή είναι διασυνοριακό το ζήτημα, θα είναι δύσκολη η διαχείρισή του εκτό αν υπάρχει νομοθεσία, εκτό αν υπάρχουν λεπτομερεί κανόνε στη συμφωνία αποχώρηση. Μπορεί αυτοί να αρκούν. Αλλά σε περίπτωση που δεν υπάρχουν, αλλά ακόμη και αν υπάρχουν, καλό θα ήταν να υπάρχει και εσωτερική νομοθεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το ζήτημα αυτό. Και το χειρότερο σενάριο είναι το να μην υπάρξει καμία συμφωνία. Σε αυτή την περίπτωση είναι απολύτω απαραίτητο για την Ευρωπαϊκή Ένωση να δράσει μονομερό για να προστατεύσει τη θέση των Βρετανών πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να είναι έτοιμη να το πράξει αυτό. Ούτω ή άλλω η χρονική στιγμή είναι δύσκολη όσον αφορά το Ευρωκοινοβούλιο, διότι εκείνη την εποχή ακριβώ θα έχετε τι νέε εκλογέ αμέσω μετά από την ημέρα του Brexit. Δεν νομίζω θα να συνεδριάσετε τον Απριλίο του 2019, οπότε θα πρέπει να δράσετε με τη διαδικασία κατεπήγοντο. Όχι μόνο για το ζήτημα τη ηθαγένεια, αλλά και ένα σωρό άλλα ζητήματα θα πρέπει να σκεφτείτε πώ μπορεί να δράσει πολύ γρήγορα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή και άλλα θεσμικά όργανα για να ασχοληθούν με όλα αυτά τα πολυάριθμα ζητήματα που είναι δυνατόν να εμφανιστούν τον Απρίλιο 2019 ε, δημιουργώντας προβλήματα σε πάρα πολλά επίπεδα και για πάρα πολλές κατηγορίες πολιτών. Και μετά το άλλο, ο εφεδρικός μηχανισμός είναι να υπάρχει μια ξεχωριστή συμφωνία για τους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και τους Ευρωπαίους πολίτες που να μπορεί να βγάλει κανείς από το σιρτάρι αν όλα πάνε ε, άσχημα. Να έχουμε δηλαδή κάτι στα χέρια μα σε περίπτωση που δεν υπάρχει τελικά συμφωνία ε, γι' αυτό θα θέλαμε το Ευρωκοινοβούλιο να δείξει κάποια βούληση να ασχοληθεί και με αυτό. Ευχαριστώ. Thank uh, Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Θα στραφώ τώρα στους ευρωβουλευτές για ερωτήσεις. Μαρτίνα και Τζίνι είπαμε θα είναι οι πρώτες, μετά η Κάτριν. Και μετά μπορείτε να επανέλθετε βέβαια αν θέλετε. Έχουμε χρόνο. Η Μαρτίνα Άντερσον πρώτα. Ευχαριστώ Κλώτ και συμπρόεδροι. και σας ευχαριστώ εσάς ε, όλους που ήρθατε εδώ σήμερα να μας μιλήσετε για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Θα πρέπει να φύγω να πάρω την πτήση μου αργότερα, αλλά θα συνεχίσουμε και ελπίζω και οι άλλοι που έχουν φύγει για να πάρουν τις δικές τους πτήσεις θα παρακολουθήσουν στην ιστοσελίδα, οπότε να ξέρετε ότι θα πιάσουν τόπο αυτά που είπατε. Εγώ συνεργάζομαι ε, με την ε, Μπάρμπαρα Σπινέλη ε, από την ομάδα Γκουε. Είμαστε δυο μας και συνεργαζόμαστε για τα θέματα του Brexit και τα παρακολουθούμε. Και χαίρομαι που είναι εδώ όλοι αυτοί οι ευρωβουλευτές που συμμετέχουν στη διευθύνουσα ομάδα για το Brexit. Ό,τι και αν λέει εκείνη η έκθεση και ότι η πρόοδος, αν θέλετε να την πείτε έτσι, έχει επιτευχθεί, σίγουρα υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια. Γιατί υπάρχει μεγάλη αμφισημία και ασάφεια. Και αυτό πρέπει να το ακούσει και η διευθύνουσα ομάδα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ολόκληρο, ξεκάθαρα. Γιατί δεν προσφέρει την ε, προστασία που θέλουν οι πολίτες. Τα δικαιώματα των πολιτών δεν είναι καμία παραχώρηση, είναι μια εγγύηση που πρέπει να έχουν. Και πρέπει να ισχύει και για τα 3 εκατομμύρια στο Ηνωμένο Βασίλειο και τα 2,5 στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση Βρετανών. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βασιζόμενοι σε αυτά τα δικαιώματα μετακινήθηκαν. Και το ίδιο ισχύει και στη Βόρεια Ιρλανδία, έτσι. Και εδώ έχουμε δικαίωμα να είμαστε είτε Βρετανοί είτε Ιρλανδοί. Ή υπάρχουν διεθνείς συμφωνίες που τα προβλέπουν όλα αυτά. Οπότε εδώ υπάρχουν δυσκολίες σε περίπτωση που υπάρξει το λεγόμενο σκληρό σύνορο ανάμεσα στη Βόρεια Ιρλανδία και την Ιρλανδία. Και όπως κι άλλοι, και εγώ θέλω να διασφαλίσω ότι ευρωβουλευτές από τις άλλες χώρες μέλη θα ξέρουν τι σημαίνει η Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής και να καταλάβουν τι διακυδεύεται για τα δικαιώματα των ε, πολιτών στη Βόρεια Ιρλανδία. Οπότε, Όταν μιλάτε για την προστασία των Ευρωπαίων πολιτών, λάβετε υπόψη σας και αυτούς στην Βόρεια Ιρλανδία. 1,8 εκατομμύρια που έχουν βρετανικό διαβατήριο σήμερα. Η εμφυσιμία, όπως σας είπα πριν, υπάρχει. Το Ηνωμένο Βασίλειο λέει θα υπάρχει τελωνιακή ένωση. Είπε στην αρχή ότι δεν θα υπάρχουν έλεγχοι, ότι δεν θα υπάρχουν σκληρά σύνορα, ότι θα ισχύει κάτι διαφορετικό για μας. Όμως η διευθύνουσα ομάδα και όλοι οι διαπραγματευτές και κυρίως ο Μισελ Παρνιέ πρέπει να ξέρουν ότι κανείς δεν ξέρει τους Βρετανούς καλύτερα από εμά τους Βόρειο Ιρλανδούς και τι σημαίνουν οι τακτικές τους διαπραγμάτευσης. Σήμερα, την επόμενη μέρα μετά την κοινή έκθεση, έχουμε και πάλι δηλώσεις. Και είπαν ότι πρόκειται για δήλωση προθέσεων. Και όλα είπε σήμερα ότι η μεταβατική περίοδος δεν θα ισχύει για τους ανθρώπους που μπαίνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο τότε. Οπότε παραμένει ασάφεια, το λέω και το τονίζω. Οι Βρετανοί στις διαπραγματεύσεις, άπαξ και εσείς βάλετε ε, τα όρια σας, αρχίζουν με καινούρια. Είναι τακτική τους. και δεν θα υπάρξει στήριξη για τα δικαιώματα των πολιτών που έχουν δικαιώματα. Δεν είναι παραχωρήσεις, είναι δικαιώματα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν πρέπει να τα πετύσει αυτά. Όλοι εσείς να ξέρετε ότι έχετε εμάς να σας στηρίξουμε. Πιέστε λοιπόν. Πιέστε τον κάθε ευρωβουλευτή της χώρας σας. Μόνο έτσι. Μόνο τους πιέσετε όλους τους ευρωβουλευτές για να ψηφίσουν με τον τρόπο που θέλετε, μόνο τότε θα υπάρξει αυτή η προστασία. Αλλιώς όχι. Δεν θα έχετε την προστασία που θέλετε και όλοι μας εμείς οι ευρωβουλευτές δεν θα είμαστε εδώ. Εσείς πρέπει να μας πρόξετε, να μας πιέσετε για να σας προστατεύσουμε. Εσείς πρέπει να μας βάλετε σε πίεση από τις χώρες σας, από όπου έρχεστε. Μόνο τότε θα τα καταφέρουμε. Πρέπει να στριμώξετε τους ευρωβουλευτές. Και αν κάποιος από εμά δεν ψηφίσει όπως θα έπρεπε να ψηφίσει, να πάτε να τον ε, βγάλετε να φανεί αυτό, να τα πείτε. σε εθαρρύνω λοιπόν αυτό να κάνετε, να μας εκθέσετε στις χώρες μας αν δεν κάνουμε αυτό που πρέπει. Γίνεται lobbying και οι ευρωβουλευτές θα αντιδράσουν όπως πρέπει μόνο αν έχουν, τους έχει γίνει κατανοητό από τα δικά σας την πίεση ότι θα εκτεθούν στις χώρες τους. Συνεχίστε λοιπόν το πολύτιμο έργο σας. Και ευχαριστώ πολύ και τον ε, πρόεδρο που μου επέτρεψα πάρω το λόγο. Ναι, μίλησα πολύ, αλλά νομίζω ότι... Ναι, ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος. Θα επανέλθεις. Ναι, ευχαριστούμε Μαρτίνα. Πολλοί αλλάζουν τα πρόγραμματά τους, κάποιοι που ήρθαν και στην αρχή της συζήτησης. Ε, συνάδελφοι, απλώς να επισημάνω ότι πολλοί το έκαναν γιατί είναι νεκρή ζώνη η πέμπτη το απόγευμα και πολλοί άλλαξαν τα σχέδιά τους για να είναι εδώ. Μαρτίνα, σου ευχαριστούμε. Και κάποια άλλη που άλλαξε τα σχέδια είναι η Τζιν Ευχαριστώ και ευχαριστώ όλους τους ομιλητές διότι παρουσιάσατε με ευκρίνεια και με λεπτομέρειες πολλά ζητήματα ε, τα οποία θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ε, για να κλειδώσουμε, για να διαφυλάξουμε, να κατοχυρώσουμε τα δικαιώματα στο μέτρο του δυνατό. Εγώ είμαι στην Επιτροπή Λίμπε και Απασχόλησης και σε αυτές ε, τις επιτροπές ε, υπάρχουν κοινά ζητήματα, κυρίως ό,τι έχει σχέση με διώματα υπηκών τρίτων χωρών. Και ε, οφείλω να πω ότι με ανησυχεί πάρα πολύ ε, ότι τεκμέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά πάσα περίπτωση για κάποια κάτι μέλη ότι αυτό το δρόμο πρέπει να ακολουθήσουμε για τους Βρετανούς που ασκούν το δικαίωμα ελεύθερης μετακίνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το αντίστροφο. Ε, η χώρα με το Ηνωμένο Βασίλειο και με ιδιαίτερη περιφέρεια εκπροσωπώ το Λονδίνο εδώ και επειδή ακούγονται διάφορα μην ξεχνάμε ότι ε, ο Δήμαρχος του Λονδίνου κάνει πάρα πολλά πράγματα εσείς ε, εξάλλου είσαστε και στη Σχετική Επιτροπή μας το είπατε. Λοιπόν, για τα ε, διάφορα που ακούσαμε ε, και τα όσα όλοι τεκμένουν θα ήθελα ε, να ρωτήσω το εξής. Για τους 27. Τελικά, ποια είναι η κοινή βάση, η κοινή θέση των 27 και συμφωνώ με τη Μαρτίνα για αυτά που κάνουμε στο ε, κοινοβούλιο. Πρέπει να μιλάμε και στα εθνικά κοινοβούλια, γιατί δεν μιλάμε μόνο για το Ηνωμένο Βασίλειο. Λοιπόν, υπάρχει συνένεση, υπάρχει συμφωνία σε σχέση με ποια δικαιώματα θα πρέπει να διατηρηθούν, όχι μόνο για όλους όσους ε, θα παραμείνουν στη χώρα όπου διαμένουν, αλλά και για αυτούς που θα ασκήσουν το δικαίωμα ελεύθερης ε, κυκλοφορίας υπηκόους τρίτων χρόνων Από, επιτροπή, την Επιτροπή Λίμπα θα πούμε ότι δεν έχουμε συνεκτική πολιτική. Είσαστε στην Ισπανία και θέλετε να πάτε στη Γαλλία γιατί βρήκατε νέα δουλειά ε, και τι αίτηση θα κάνετε, τη μπλε κάρτα γιατί έχετε υψηλέ ε, δεξιότητε. Ο Κλόντ είναι εισηγητή τώρα. Προ, προ, προσπαθώ να το κρύψω. Υπάρχουν λοιπόν διαφορετικά δικαιώματα ανάλογα με τα κράτη-μέλη για υπηκόους τρίτων χωρών. Βλέπω τον κατάλογο θέματα οικογενειακής επανένωσης, πρόσβαση στην εκπαίδευση, διάφορα πράγματα. Για τους αυτά απασχολούμενους, ε, τα κράτη-μέλη έχουν διαφορετικές προϋποθέσεις ε, για την είσοδο και την καταχώρηση υπηκών τρίτων χωρών. Ε, δηλαδή, τι κεφάλαιο πρέπει να έχουν για να ανοίξουν δική τους δουλειά, τι εκπαίδευση κτλ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, λοιπόν, σε επίπεδο 27 λειτουργεί ως ομάδα και γενικότερα. Δηλαδή θέλω να πω όταν ε, είναι εύκολο όταν ε, έχεις κάποιον ε, απέναντί σου, συγκεκριμένη περίπτωση του να λειτουργεί σαν ομάδα. Αλλά μεταξύ τους τα κράτη-μέλη λειτουργούν τελικά ως ομάδα. Και ε, τώρα να μην το πω να μου καταλόγει τα ψωνιά, μία, ένα ε, κατάλογο για το τι πράγματα πρέπει να κάνουμε για να μπορέσουμε να έχουμε μία κοινή προσέγγιση. Ευχαριστώ. Θέλω να πω ε, μόνο για να ξέρετε όλοι τι συμβαίνει. Ο Ρομπέρτο πρέπει να φύγει έχει πτήσει, έχει οικογένεια που τον περιμένει, εκλογέ, για χαμό, όλα τα έχει, πρέπει να φύγει. Αλλά επειδή είναι στην ε, Διευθυντική Επιτροπή, θέλω να τη δώσω το λόγο. Η Κάθριν Μπίρντερ, ε, ξέρετε τώρα ότι δραστηριοποιείται ιδιαίτερα. Και μετά η Τζούτ. Ε, απλά τα λέω για να ξέρετε ποιος, με ποια σειρά θα μιλήσετε. Ε, ε αν, αν συμφωνείς, έτσι μόνο να ακούσουμε τον Ρομπέρτο. Ε, Ευχαριστώ τους ομιλητές για την πολύτιμη συνεισφορά τους και θέλω να παραμείνουμε σε ε, επαφή για να εξετάσουμε ε, και τα νομικά κείμενα και με προσοχή να εξετάσουμε κάποιες συγκεκριμένες ιδέες. Λοιπόν, Σούρινγκ ε, the Sing, δεν καλύπτεται αυτή η περίπτωση. Θα, θα κλείσουμε αυτό το παράθυρο, αυτή την πόρτα μάλλον. Ε, για την ε, θέσπιση της ε, Εθνικής Ανεξάρτητης Ορχής. Το παρακολουθούμε εκ του σύνεγγης. Είναι στο ραντάρ μας, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Και εξετάζουμε όλα τα σενάρια. Μιλάω τώρα για τον καθηγητή Πόρτες. Ε, γιατί... Ε, πρέπει να ξέρουμε τι διατάξει ισχύουν για ένα κράτο μέλο. Δεν μπορούμε να έχουμε διαφορέ ε, και με όσο πιο όμοιε είναι οι διατάξει, ε, τόσο το καλύτερο. εάν αλλάξουν οι κόκκινες γραμμές, μια δι... ακρατική συμφωνία είναι καλύτερη εναλλακτική για μας, για τέτοια πράγματα εννοώ. Λοιπόν, θέλουμε με κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις και όσο πιο ε, στενή είναι η σύγκληση τόσο το καλύτερο αλλά φυσικά υποαίρεση και αυτό σχετίζεται με αυτό που είπατε και παρότι αποκλείεται τώρα από τη θέση τη Βρετανική κυβέρνηση είναι ένα σενάριο. Ρομπέρτο, ε, ευχαριστώ και ξέρω ότι θα είσαι επαφή με τους συναδέλφους ε, που ήρθαν στα πλαίσια της ε, ομάδας για το Brexit και εδώ. Η Κάθριν Μπίρντερ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ θα ήθελα να προσθέσω τις ευχαριστίες μου για όλους τους ομιλητές που ήρθαν εδώ για να συμμετέχουν στο πάνελ και τα μέλη της Διευθυνούσης Επιτροπής που μας μίλησαν 587 ημέρες έχουν περάσει από το δημοψήφισμα. Κάθε μια από αυτές τις μέρες ε, είναι απελπιστική για τους πολίτες του Brexit, τους Βρετανούς πολίτες που ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ονομάζονται πολίτες του πουθενά από τη δική τους Πρωθυπουργό η οποία απορρίπτει αυτό το δικαίωμα για αυτούς τους πολίτες που ζουν εκτός του Νόμου Βασιλείου να ψηφίσουν ε, για ε, το Brexit. Έχουμε δηλαδή μια κυβέρνηση που ήδη δεν εκτιμά επαρκώς ε, την κατάσταση. Και επίσης, και πρέπει να σημειωθεί αυτό, αντιλαμβάνομαι αυτά που λέτε για πέμπτη απόγευμα είναι δύσκολο για τους ευρωβουλευτές, αλλά πολλοί από εμάς καταφέραμε να είμαστε εδώ γιατί είναι κάτι σημαντικό μας εκλέγουν πολίτες, εκπροσωπούμε πολίτες στο Ευρωκοινοβούλιο. Ούτε ένας βουλευτής από το UKIP συντηρητικός δεν βρίσκεται εδώ για να συμβάλλει στη συζήτηση. Θα πρέπει λοιπόν να το αναφέρουμε αυτό ρητά. Είναι ντροπή τους. Είναι αναμφίβολο κατά την απόψη μου ότι οι Ευρωπαίοι πολίτε στον Ηνωμένο Βασίλειο αισθάνονται ότι βρίσκονται σε ευάλωτη θέση. Και το ίδιο ισχύει και για του Βρετανού που ζουν στην υπηρετική Ευρώπη. Και ειδικότερα για του πολίτε που βρίσκονται και εδώ, του εκπροσώπου του. Υπάρχουν πολλά εκκρεμή ζητήματα. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι οι κόκκινε γραμμέ ε, θα πρέπει να τι λαμβάνουν υπόψη οι διαπραγματευτέ ε, αποκλείται να υπογραφεί η συμφωνία χωρίς να υπάρχουν σαφείς τέτοιες γραμμές. Είχαμε ήδη... Πρέπει να έχουμε νομική βεβαιότητα και για τα σύνορα στη Βόρεια Μιλάμε για ανθρώπινα όντα. Ε, δεν μπορούμε να αποφασίζουμε έτσι για τις ζωές τους δεν είναι ότι το Ευρωκοινοβούλιο κάνει το δύσκολο. Είναι η δουλειά μα αυτή. Υπερασπιζόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα και διασφαλίζουμε την εφαρμογή του. Σε ε, αμφότερε τι πλευρέ ε, τη συζήτηση. Έχω μια ερώτηση προ του ε, νομικού εκπροσώπου που είχαμε εδώ. Οι κατευθυντήριε γραμμέ για τη μεταβατική περίοδο λένε ότι το ΕΒ πρέπει να δεχτεί ολόκληρο το κεκτημένο Δηλαδή θα ήταν νόμιμο το Ηνωμένο Βασίλειο να εισάγει αυτή τη στιγμή ένα σύστημα εγγραφή, κάτι που έπρεπε να έχει γίνει εδώ και χρόνια για του Ευρωπαίου πολίτε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι νομικό το θέμα. Και επίση, ε, όσον αφορά την επέκταση τη εποπτεία ε, του δικαστηρίου, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου πέραν τη πενταετία, και η πρόταση για την ανεξάρτητη εθνική αρχή ώστε η συμφωνία να εφαρμοστεί σωστά και να μην απομειωθούν τα δικαιώματα από μελλοντικέ κυβερνήσει. Όλα είναι καλά άμα το υπογράφει η συντηρητική κυβέρνηση με ένα, αλλά πρέπει να θεσπίζεται με απόλυτους όρους όλο αυτό το νέο καθεστώς των Ευρωπαίων πολιτών στο Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να είναι ένα σύστημα εγγραφής δηλωτικού χαρακτήρα που να επιβεβαιώνει και να θεσπίζει τα δικαιώματα. Εμεί πρέπει να είμαστε μετακίνητοι σε αυτό. Η αίτηση πρέπει να είναι απλή, ψηφιακή και κυρίω δωρεάν. Η ηθαγένεια δεν εξαρτάται από την ικανότητα κάποιου να την αγοράσει. Επίση πρέπει να διασφαλιστεί η κάλυψη ομάδων που δεν δίνανται να συμπληρώσουν μια ψηφιακή αίτηση διότι δεν μπορούν να το κάνουν ε, λόγω σωματικών ικανοτήτων, γλωσσικών ικανοτήτων ή διότι έχουν άλλε ευθύνε. Ε, το ζήτημα των γυναικών που αναφέραμε όταν μεγαλώνουν παιδιά και τέλος η οικογενειακή πανένωση θα πρέπει να περιλαμβάνει και τους μελλοντικού ε, συντρόφους και συζύγους αν τους εξαιρέσουμε θα επηρεαστεί η νεότερη γενιά δυσανάλογα καθώς και τους πολίτες που μετά από θάνατο ή διαζύγιο επιθυμούν ενδεχομένω να ξαναπαντρευτούν μετά τον Brexit. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Οι ευρωβουλευτές θα πρέπει να αναφέρουν ε, αυτά τα θέματα και να ε, καλέσουν πρώτε ευθύνε τους και τους διαπραγματεύτέ για τον Brexit και τους αξιωματούχους της βρετανική κυβέρνηση. Ευχαριστούμε πολύ Κάθριν, ευχαριστούμε για τις προσπάθειές σας. Ε, είναι μια, υπάρχει μια άτυπη ομάδα που δραστηριοποιείται σε αυτό. Είναι άτυπη, δεν είναι μυστική ομάδα, οπότε μπορώ να την αναφέρω. Τζιουντ, ε, η Ρενάτα Βέμπερ μόλι ζήτησε από την Επιτροπή Απασχόληση ε, και αυτή γνωρίζει πολλά πράγματα και για τη ΛΥΜΠΕ. Θέλετε να πείτε κάτι και μετά, Τζούντι, θα κάνετε στην τελευταία ερώτηση πριν επιστρέψουμε στο πάνελ. Ευχαριστώ πολύ. Την πρώτη φορά που έγινε ακρόαση ε, ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Έτσι συμβαίνει και σήμερα. Σίγουρα έχουμε προχωρήσει. Έχουμε επιτύχει κάποια πράγματα, αλλά η αλήθεια είναι ότι σε ολόκληρη την Ευρώπη ο κόσμος ανησυχεί. Την περασμένη εβδομάδα μίλησα με μια αντιπροσωπεία από τη Χιλή. Ε, η δίπλα μου ήταν κάτι Βρετανοί που ζουν στην Ισπανία και δεν ξέρουν τι θα γίνει στο μέλλον. Θα μπορούν να μετακομίσουν σε άλλη χώρα, τι θα γίνει με τις συντάξεις τους, την κοινωνική τους ασφάλιση, τα ζητήματα ασφαλής υγείας. Έχουμε πει επανειλημμένω ότι η Βρετανική κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται και τόσο πολύ για τους Βρετανούς πολίτες, ούτε για τους Ευρωπαίους πολίτες. Αλλά πρέπει να σας πω πως από ιστορίες που εγώ ακούω και από παράπονα που ακούω, μαθαίνω ότι και οι άλλες κυβερνήσεις δεν ενδιαφέρονται τόσο πολύ να προστατεύσουν τα δικαιώματα των Βρετανών υπηκών. Έχουμε περιπτώσεις και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου κάποιοι που ήταν Ευρωπαίοι πολίτες βρίσκουν ξαφνικά ότι πρέπει να αιτιολογήσουν γιατί ως αυτοί ήταν Βρετανοί πολίτες αλλά τα παιδιά τους πηγαίνουν σχολείο στη Γαλλία ή κάπου αλλού. Οπότε δεν είναι να κατηγορούμε μόνο τη μία πλευρά. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι ότι εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο πρέπει να συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση στους διαπραγματευτές. Διότι πράγματι φοβόμαστε πολλοί από εμά εδώ ότι κάποια στιγμή αρκετά σύντομα ε, η συζήτηση θα περιστρέφεται γύρω από το χρήμα και οι πολίτες θα είναι κάπου θα έχουν μπει στην άκρη. Φυσικά, ναι, έχουν επιτευχθεί κάποια θετικά πράγματα μέχρι στιγμής και αυτό θα βοηθήσει πολλούς αλλά μην ξεχνάμε και τους υπόλοιπους. Δεν μπορούμε να αφήσουμε κόσμο πίσω μας, ε, ανθρώπους ε, των οποίων οι ζωές θα καταστραφούν εντελώς, ε, χωρίς να φταίνε οι ίδιοι. Απλώς και μόνο επειδή άλλαξαν κατά κάποιο τρόπο τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχω λοιπόν μια ερώτηση και θέλω μάλιστα να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές σήμερα διότι πραγματικά οι παρουσιάσεις τους ήταν εξαιρετικές και φυσικά πρέπει να ανησυχούμε ε, και αυτοί πρέπει να ανησυχούν ακόμη περισσότερο από ότι εμείς εδώ. Ναι, παρακαλώ, ανησυχείτε, ασκήστε πίεση και σε εμά. Αλλά η ερώτησή μου είναι ε, για μια κατηγορία ανθρώπων που δεν άκουσα ιδιαίτερα να αναφέρεται, οι φοιτητέ φοιτητές που είναι τώρα στο Ηνωμένο Βασίλειο που πρέπει να συνεχίζουν τις σπουδέ τους, ε, αυτοί που θέλουν να πάνε στο μέλλον. Τουλάχιστον ε, να πούμε κάτι για τους φοιτητές. Έχω την εντύπωση ότι οι Βρετανοί ε, υπηκοοί θα είναι πάντα ευπρόσδεκτοι σε οποιοδήποτε πανεπιστήμιο της υπηρετικής Ευρώπης. Αλλά δεν είμαι επεπισμένο ότι θα συμβαίνει και το αντίστροφο. Έχουμε τους ιδανικούς ανθρώπους για να απαντήσουν αυτό το θέμα. Έχει αναφερθεί αυτό το ζήτημα παλιότερα. Ε, Τζούντιθ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Κλοντ, που μου δίνεις ε, την ευκαιρία να δευτερολογήσω. Ήθελα να ε, επικυρώσω κι εγώ αυτά που είπε ο Τζόναθαν Πότερ ότι είναι πιθανό να αλλάξει η θέση του νομού Βασιλείου. Πολλοί από εμάς ε, έχουμε αγωνιστεί για να αλλάξει η θέση της κυβέρνησης του νομού Βασιλείου. Εξορισμού πολλές από τις κόκκινες γραμμές δεν συναντούν με πολλές από τις δηλώσεις των Υπουργών και με το τι προτείνεται να προσφέρουν. Οπότε κάποια στιγμή υποψιάζομαι ότι θα υπάρξει μια αλλαγή της θέσης, μια μεταβολή της κρατικής θέσης. Μπορεί να υπάρχει μια νέα ε, κυβέρνηση άλλου πολιτικού χρώματος. Ε, χρειάζεται μεταβολή της, της ε, κυβερνητικής θέσης. Τώρα από πλευράς Ηνωμένου Βασιλείου. Ε, το λιγότερο κακό μοντέλο Brexit είναι να παραμείνουμε στην Τελωνιακή Ένωση και στην ενιαία αγορά. Δεν υπάρχουν εδώ πολλοί μη Βρετανοί βουλευτέ λόγω τη ώρα που έλαβε χώρα η συνεδρία και λόγω του ότι ο κόσμο έπρεπε να προλάβει τα αεροπλάνα του. Αναρωτιέμαι αν στην Ευρώπη, στι 27 χώρε, χρησιμοποιείται το Brexit για να επανακαθορίσει και το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Μου έκανε εντύπωση η Τζέιν ανέφερε ότι εξεπλάγει πω ε, στο τελευταίο σχέδιο της συμφωνίας το Δεκέμβριο εμφανίστηκε ξαφνικά μια υποχρέωση για Βρετανού υπηκόους να εγγράφονται στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν υπήρχε παλιότερα. Ήθελα να πούνε οι άλλοι ομιλητέ, οι «Ε, Έστερ, εσεί από το συνδικάτα ή όταν συζητάτε την κοινωνική Ευρώπη, υπάρχει κάποια τάση ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση που αμφισβητείται σήμερα ω αποτέλεσμα των συζητήσεων για τον Brexit και υπάρχουν περαιτέρω ευρύτερε προκλήσει που να απειλούν το μοντέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ εμεί στο Ηνωμένο Βασίλειο προσπαθούμε να ε, πιέσουμε για να συνεχιστεί αυτή η στενότερη σχέση. Από την άλλη πλευρά των διαπραγματεύσεων, λοιπόν, μήπω κάποιε από τι ε, πολύ θεμελιώδει αξίε που έχουμε υπερασπίσει εδώ αμφισβητούνται αυτή τη στιγμή στι άλλε 27 χώρε του Ηνωμένου Βασιλείου ω αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων για τον Brexit. Γιατί τέτοια αίσθηση αρχίζουμε, αρχίζουμε να αποκτάμε, κάπω αφηρημένα. Είναι απλά μια αίσθηση. Καλό θα ήταν λοιπόν να μα πούν και κάποιοι εμπειρογνώμονε, κάποιοι ειδικοί τι απόψει του για το αυτό, για το πώ συμβαίνει ε, συγκεκριμένα. Ευχαριστούμε πολύ. Μπάρμπαρα, θέλετε να πείτε κάτι πριν πάμε στο πάνελ, παρακαλώ. Ένα λεπτό. Θέλω να πω κάτι για αυτά που είπε η Τζούντιθ. Είναι ζωτική σημασία ζήτημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να χρησιμοποιήσει αυτή την ευκαιρία για να κάνει νομοθεσία ακόμα πιο περιοριστική μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το είπα και εγώ στην εισαγωγή μου. το άνοιγμα αυτό στη διατύπωση τι θα γίνει με την Ευρώπη των 27 και τους Βρετανούς υπαλλήλους μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν πρέπει να παρθούν αποφάσεις που να αντιβαίνουν τελικά στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Ευχαριστούμε. Είμαι παδός της Μπάρμπαρα Σπινέλη, οπότε λέω πρόεδρος τη θαυμάζω. Το πάνελ μας τώρα. Έχουμε μισή ώρα στη διάθεσή μας. Γιάννη πρώτα. Είναι σαφές ότι με την ακρόαση αυτή θέλαμε να κάνουμε τη σύνδεση με αυτά που ισχύουν, με αυτά που έχουμε πετύχει μέχρι τώρα και τι μένει. Ευχαριστώ εγώ στην τελευταία μου διαφάνεια είχα μια σύσταση για τη διατύπωση, ακριβώς γι' αυτό που είπε η Μπάρμπαρα Σπινέλη, δηλαδή όλοι όσοι έχουν το δικαίωμα διαμονής βάσει του ευρωπαϊκού δικαίου. Αντί να λέμε βάσει αυτή τη οδηγία ή αυτού του κασμού ή αυτού του δεν ξέρω εγώ τι κάτι το οποίο υπονομεύει τελικά το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Γι' αυτό έβαλα αυτή τη διατύπωση που ελπίζω η διευθύνουσα ομάδα να την κοιτάξει. Τώρα, είπαμε για τους φοιτητέ. Τι θα γίνει με τους φοιτητέ, στη σύγκριση στην κοινή δήλωση το λέει, είναι το 3α που λέει αυτή η βάση του 7-1-C c καλύπτονται. Αλλά αυτό έχει να κάνει με την ασφάλιση. Και πάλι μπορεί να πει το Ηνωμένο Βασίλειο, εμείς δεν βασιζόμαστε σε αυτήν την συνολική κάλυψη. Θα έπρεπε γραπτά να συμπεριληφθεί στη συμφωνία από το Ηνωμένο Βασίλειο. Αλλιώς πολλοί θα μείνουν εκτός. Για παράδειγμα, όσοι φροντίζουν ε, συγγενείς τους, μέλη της οικογένειάς τους. Και είπατε κάτι για την καταγραφή. Θα το αφήσω για κάποιον άλλον ίσως για τον κύριο Πέρς. Και κατά πόσο είναι υποχρεωτική ή όχι και από τι εξαρτάται. Τέλο πάντων, νομίζω ότι καλύφθηκε. Ε, αν είχατε άλλε ερωτήσει, ευχαρίστω, αλλά μετά, αν κάτι ξέχασα. Μετά από αυτή τη συνάντηση και το λέω για να τα ακούσουν όλοι. Θα έχουμε μια συνάντηση της ομάδας Brexit. Ήταν να την έχουμε μάλλον, αλλά κυρώθηκε επειδή ακριβώ πολλοί έπρεπε να ταξιδέψουν. Θα επανέλθουμε όμως. Γιατί θα μας βοηθήσει αυτή η ακρόαση. Καλό είναι να κρατήσουμε την επαφή αυτή μαζί σας, η Διευθύνουσα Επιτροπή, ώστε να μπορείτε να μας ενημερώνετε πιο συγκεκριμένα. Είδατε, ο Ρομπερτό Κουαλτιέρη είναι σαφής. Οι τρεις επιτροπές μας θα προσπαθήσουν αυτή η επαφή να παραμείνει. Οπότε τις διαφάνειές σας, αν θέλετε να τις στείλετε στη διευθύνουσα ομάδα, βεβαίως. Εμεί θα συνεδριάσουμε κατά στο Στρασβούργο την επόμενη εβδομάδα, αυτή η επιτροπή που σα είπα. Και η Μαρίτα και άλλοι πρόεδροι που θέτει παρόντε θα ενημερώνουν τι επιτροπέ του. Λοιπόν, επόμενο η Έστερ. Έστερ να απαντήσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όσον αφορά την ανάλυση αυτή, είναι πολύ σωστή. Για κάποιες χώρες το μάθημα του Brexit είναι ότι χρειαζόμαστε λιγότερη Ευρώπη αντί για περισσότερη. Λιγότερα δικαιώματα υπέρ των εργαζομένων παρά περισσότερα, λένε μερικοί. Φυσικά αυτό είναι εντελώ λάθος. Το 2004, τρεις χώρες άνοιξαν τα σύνορά τους για την ελεύθερη κυκλοφορία Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο και Σουηδία. Η διαφορά ανάμεσα στη Σουηδία, την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ότι η Σουηδία και η Ιρλανδία είχαν νόμους στη διάθεσή τους που προστάτευαν τις συλλογικές συμβάσεις. Και τι κάνουν αυτοί οι νόμοι, λένε ότι αν είσαι ας πούμε στην οικοδομή Ακόμα και αν θες να πληρώσεις λιγότερο τον εργαζόμενο δεν μπορείς να το κάνεις. Στον Ηνωμένο Βασίλειο δεν υπήρχε αυτή η νομοθεσία. Στην Ιρλανδία οι εργαζόμενοι και στη Σουηδία δεν φοβούνται λοιπόν την ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων όπως οι υπόλοιποι. Το μάθημα συνεπώς είναι ότι μια χαρά είναι η ελεύθερη κυκλοφορία. Δεν είναι κάτι το απειλητικό, αν όμως διασφαλίσεις ότι δεν θα γίνεται εκμετάλλευση. Αν δεν το διασφαλίσεις αυτό, τότε οι εργαζόμενοι δεν θα έπρεπε να μας εκπλήσει που φοβούνται. Και αυτό είναι το μάθημα νομίζω που μπορούμε να πάρουμε και για να καταλάβουμε γιατί υπάρχει ο φόβος για την ελεύθερη διακίνηση. Τώρα μια άλλη ερώτηση θα ενδιαφέρουσα. όλοι θα ενδιαφέρουσες τέλος πάντων, λέω για μένα. τι σκέφτονται οι υπόλοιποι εργαζόμενοι στην Ευρώπη για το Brexit και τη συμφωνία αυτή. Θα σας εκπλήσει το ότι πολύ συχνά σε συναντήσεις με τους εργαζόμενους διαπιστώνουμε ότι ενδιαφέρονται πάρα πολύ. Καταλαβαίνουν ότι είναι μια μεγάλη χώρα η οποία θα εξακολουθεί να βρίσκεται στην Ευρώπη γεωγραφικά ως μια μεγάλη χώρα, δεν θα πάει να φύγει στο φαγκάρι, θα εξακολουθεί να είναι κομμάτι της αλυσίδας. Και παρόλα όσα λέει η Πρωθυπουργό για το social dumping και τα λοιπά, θα συνεχίσουν να ισχύουν πολλά. Οπότε δεν είναι μια συζήτηση από την οποία το Ηνωμένο Βασίλειο θα διαλέξει ότι θέλει και ότι θα υπάρξουν δίκες συνθήκε για όλους. Πρέπει να δούμε τελικά το Ηνωμένο Βασίλειο θα έχει πρόσβαση στην ενιαία αγορά, αλλά από την άλλη να μην μπορεί να συμμορφωθεί όσον αφορά τα δικαιώματα των εργαζομένων, υπερολλαντικές και δημοσιονομικές προδιαγραφές. Όχι, δεν γίνεται. Και αυτό είναι σημαντικό να το καταλάβει ο κόσμος. Πριν περάσουμε στις λεπτομέρειες. Οι άνθρωποι βιάζονται βέβαια και θέλουν να δουν τελικά αυτή η συμφωνία που θα καταλήξει. Τζούλια. Εγώ θα ήθελα να σχολιάσω αυτό που ακούσαμε πριν, δηλαδή ότι ε, τελικά υπάρχει ομοιομορφία σε σχέση με τις απαντήσεις που δίνουμε για την μεγάλη ανασφάλεια που επικρατεί. Πάντως είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί από όλες αυτές τις διαφορετικές οπτικές γωνίες ουσιαστικά τα ίδια λέμε. Είναι τόσο καταστρεπτικά και φοβερά τα αποτελέσματα του Brexit για τους πολίτες. Ε, συναντηθήκαμε έναν ε, διευθυντή μιας μεγάλης ε, εταιρείας πρέπει να επιστρέψει στην Ευρώπη και να ρωτιέται τι σημαίνει αυτό για την οικογένειά του που είναι στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μπορεί να το δει κάποιο το θέμα από διάφορα πρίσματα και υπάρχουν πολλές διαφορετικές περιπτώσεις. Ε, πάντως ε, τα πρέπει να δοθούν ε, απαντήσεις για τα δικαιώματα των Βρετανών πολιτών. Είναι πραγματικά κέρια σημασία. Το Υπουργείο Ιστορικών Υποθέσεων καταβάλει προσπάθειες για να απλοποιήσει το σύστημα καταγραφής και μάλιστα με καινοτόμο τρόπο. Δεν προσπαθούν να προσαρμόσουν κάποιο παλιό σύστημα, ένα νέο προσπαθούν να φτιάξουν για να λειτουργήσει εύρυθμα και κάνουν πολλές προσπάθειες για να βοηθήσουν αυτούς που έχουν περιέλθει σε επισφαλή θέση και δεν θα τους ζητηθεί χωρίς ε, υποστήριξη να έχουν πρόσβαση σε αυτό το νέο σύστημα. Για να πούμε και κάτι θετικό, έτσι, νομίζω ότι θα το βρουν θετικό όλοι όσοι θα κληθούν να το χρησιμοποιήσουν. Mm. Σας ευχαριστούμε. Ο Τζόναθαν. me what to what to pick up. I mean, pick up just anything that you've heard that you want to pick up. I'm going to put. Τι θα ήθελες να πω. Σ' αγαπώ, Τζόναθαν. Θα ήθελα να... εσύ να απαντήσεις ό,τι θέλεις. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Ό,τι θες, ό,τι θες πες. Ό,τι έχει σχέση ίσως με τη διευθυντική του Brexit. Αυτό που είπε για τη Τζούλη είναι καταστρεπτικά τα αποτελέσματα και για τις οικογένειες και για τις ε, επιχειρήσεις. Ε, είναι πάρα πολύ μεγάλη η ανασφάλεια. Πρέπει να κλειδώσουν αυτές οι διατάξεις ε, ούτως ώστε να ξέρουμε πώς θα αλλάξει η διοίκηση, πώς θα αλλάξει επιχειρηματικός κόσμος, να ξέρουμε τι θα γίνει μετά το Brexit. Και όντω, εντάξει, δεν έχει και απεριόριστου πόρου, αλλά το Υπουργείο Εσωτερικών Υποθέσεων ε, ε, καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια. Και σαν λέω, πρέπει να αποκρισταλωθούν, να κλειδώσουν οι διατάξει. Και τονίζω και πάλι όπως στην παρουσίασή μου, πρέπει να έχει δόντια και εξωπραγματικές εξουσίες ε, η ανεξάρτητη εθνική αρχή. Δεύτερο, τα κράτη-μέλη που χρησιμοποιούν χρησιμοποιούν το Brexit για να ε, υπαναχωρήσουν σε σχέση με το κατοχυρώμενο αυτό δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας. Ε, αυτό ρωτήσατε. Από τη δική μου οπτική γωνία δεν το βλέπω, ίσως φάλω από οικονομικής πλευράς. Ε, ένα από τα θετικά του Brexit είναι ότι στους 27 πλέον ε, έχει αναγνωριστεί ότι είναι αλληλένδετη σε τέσσερις ελευθερίες και ε, βασικές ελευθερίες και ότι υπάρχουν σημαντικά ωφέλη ε, που συνδέονται με αυτό, με το ότι είναι αλληλένδετη δηλαδή. Ε, ξε... Μην ξεχνάτε τι έγινε με τις περιπτώσεις Βίκινγκ και Λαβάλ και την απόσπαση των εργαζομένων. Υπάρχει Επίσης και ε, μειοψηφική η θέση ότι έχει αναβαθμιστεί ο πολιτικός διάλογος στο Ηνωμένο Βασίλειο με τον Brexit δημοσκοπήσεις ε, από τότε που έγινε το δημοψήφισμα για το Brexit ε, έχουν, δείχνουν αλλαγή ε, της ε, ε, άποψης του κοινού σε σχέση με την μετανάστευση και ξέρετε ότι συνειδητοποιούν οι άνθρωποι ποια, ποια αντισταθμιστικά ωφέλη τώρα θα προκύψουν από αυτές τις νέες διατάξεις και θα πρέπει να ξέρουμε τι είναι δυνατό και τι δεν είναι δυνατό να γίνει. Και όχι μόνο δεν μπορούμε αλλά να διαλέγουμε όποιο θεσμικό όργανο και όποια νομοθεσία μας βολεύει, αλλά το ίδιο δεν μπορούμε να κάνουμε με τους ανθρώπους και τους μετανάστες. Άμα πούμε ότι δεν θέλουμε ελεύθερη κυκλοφορία και θέλουμε μόνο τους επιθυμητούς ε, μετανάστες, μην ξεχνάτε πρέπει να θέλουν και αυτοί να έρθουν και αν το πούμε μπορούμε, μπορεί να συμβεί το εξή ότι ε, θα βρούμε αυτούς που θέλουμε. Ξέρω εγώ ότι να είναι ακαδημαϊκοί, ε, νοσοκόμες κτλ. Αλλά θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ακόμη και προ-Brexit πλήττεται η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου και υπάρχει μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού που ε, το έχαψαν ε, ε, για τα περί αποκατάστασης των συνόρων και της ανάσχεσης της μετανάστευσης συνειδητοποιούν ότι δεν είναι όλα τόσο ρόδινα και θα πρέπει λοιπόν να, το ταχύτερο δυνατόν να διαμορφωθούν οι εξελίξεις. Ευχαριστούμε και τέλος ο κύριος Πίερς. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να αναφερθώ στο ζήτημα της καταγραφής και αν υπάρχει κάτι που θα εμποδίζει το Ηνωμένο Βασίλειο να το πράξει. Να ξεκινήσω βέβαια, φυσικά αυτό θα ξεκινήσει πριν από την ημέρα του Brexit, αλλά το ζήτημα του κατά πόσο θα υπάρξει στασιμότητα ε, θα εξαρτηθεί από την κείμενο εγώ υποθέτω ότι οι επιλογές που έχει ήδη το Ηνωμένο Βασίλειο υπό οποιαδήποτε νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξακολουθήσουν να είναι διαθέσιμες για το Ηνωμένο Βασίλειο και μετά τον Brexit και μετά από τη μετάβαση. Διότι η μετάβαση περιλαμβάνει και τις επιλογές που υπάρχουν στην νομοθεσία και σε άλλες ε, ε περιπτώσεις ενδεχομένως να θέλει να ασκήσει κάποια άλλη επιλογή το Ηνωμένο Βασίλειο ε, για να προσαρμοστεί ε, στη διαδικασία. Σκοπός της ε, καταγραφής φυσικά είναι να ενταχθεί και στο σενάριο μετά τον Brexit φυσικά. Αν δεν υπάρχει λοιπόν κάποια ρήτρα διατήρηση του status quo στην ε, νομοθεσία, το ΕΒ Βασίλειο νομικά θα μπορεί Τώρα οι ρήτρες αυτές ε, μη αλλαγή ε, του στατοσκό θα θέσουν θέματα όσον αφορά τη μελλοντική σχέση για φορολογικά θέματα, θέματα απασχόλησης, περιβαλλοντικά θέματα. Αυτά θα παίξουν τεράστιο ρόλο. Θα τα δούμε λεπτομερώς. αλλά δεν υπάρχει ε, αρχή μη υποβάθμισης των δικαιωμάτων εάν δεν υπάρξει ρητά στην ε, συμφωνία. Εμείς ελπίζουμε ότι θα περιέχει κάποια εχέγγυα τα οποία θα αφορούν ε, τα διαφορά ζητήματα προστασίας και θα πρέπει να μεριμνηθεί ώστε να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα, να μην υπάρχει καμία αμφιβολία, να είναι σαφές από την αρχή ποια όρια υπάρχουν. Αυτό θα ήταν πολύ χρήσιμο. Ε, ευχαριστώ πολύ, Steve θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη των τριών επιτροπών που οργάνωσαν αυτή τη συνάντηση και τα μέλη του προσωπικού και ειδικότερα να ευχαριστήσω τους ομιλητές και όλους όσους τους συνόδευσαν διότι ήρθαν εδώ χάρη στο έργο που επιτελούν. Το εκτιμούμε ιδιαίτερα. και εδώ έχουμε πολλά στοιχεία τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στη Διευθύνουσα Επιτροπή για τον Brexit. Αυτό ήταν και ο σκοπό τη ακροασή. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να μεριμνήσουμε εδώ και στι τρει επιτροπέ για τη διαβίβαση αυτών των στοιχείων. Ένα από του λόγου ε, για του οποίου ε, απευθύνω τι ευχαριστίε μου, πέραν όλων των πολιτικών πραγμάτων που θα μπορούσα να πω φυσικά για να βγω στι επικεφαλίδε, ήμουν χθε ε, σε μια συνάντηση με τον κύριο Μπαρνιέ και με του προέδρου όλων των επιτροπών ο κύριος Φερχόφστα ήταν εκεί και αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν οι συζητήσεις για το τι θα γίνει από τώρα μέχρι τον Οκτώβριο. Πάρα πάρα πολλά πράγματα θα πρέπει να διαπραγματευτούμε. Το δικαιώματα των πολιτών έχει απομείνει ουσιαστικά από την πρώτη φάση. Αλλά συζητώνται αυτή τη στιγμή τα πάντα η Επιτροπή μου εμπλέκεται στα πάντα, σε όσα πρόκειται να συζητηθούν από την προστασία των δεδομένων, την ασφάλεια και όλα είναι κατεπήγοντα. Αυτό είναι εξαιρετικά ανησυχητικό, διότι κάποια πολύ σημαντικά ζητήματα ε, ναι, εντάξει, σας διαβεβαιώ, τα δικαιώματα των πολιτών είναι από τα πιο σημαντικά. Αλλά το πρόβλημα είναι ουσιαστικά ότι ο χρόνος εξαντλείται. Η σημερινή λοιπόν ακρόαση είχε σκοπό να σα διαβεβαιώσουμε ότι έχουμε δεσμευτεί, αντιλαμβανόμαστε τον επίγοντα χαρακτήρα του θέματο, αναγνωρίζουμε το έργο που έχετε επιτελέσει και αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να συνεργαστούμε ώστε να επιτύχουμε τα αποτελέσματα που χρειαζόμαστε μέχρι τον Οκτώβριο και πέραν αυτού στις 31 και μετά θα δούμε τι θα γίνει μετά από όλα αυτά. Όλα τα σενάρια είναι δυνατά. Εκτιμάμε ιδιαίτερα όλα αυτά που είπατε αυτή η ακρόαση είναι από τις ε, πολύ ενισχυμένες, πλας, πλας, πλας, την λέει ο πρόεδρος. Θέλουμε να παραμείνουμε σε επαφή μαζί σας ε, για να ακούμε τις ε, έμπειρες γνώμες σας, την εμπειρογνωμοσύνη σας. Θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη που συμμετείχαν ενεργά στον τομέα εδώ και είμαι βέβαιος ότι θα ακολουθήσουν πολλές άτυπες και τυπικές επαφές. Θα έχουμε το ψήφισμα το Μάρτιο που θα είναι το επόμενο βήμα. Και αυτό θα έχει και μεγαλύτερη προβολή στα μέσα, όπω θα εντείνεται η προβολή αυτή στα μέσα, καθώ θα κινούμαστε προ τον Οκτώβριο. Ευχαριστώ πολύ για τη συμβολή σα. Σήμερα το εκτιμάμε ιδιαίτερα και από τι τρει επιτροπέ μα. Σα ευχαριστώ και ελπίζω να σας ξαναδούμε, να σας ξανα... ξανασυζητήσουμε μαζί σας σύντομα. Ευχαριστώ.